της Επιτροπής ε, σχετικά με την προσφυγική κρίση, τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και το μέλλον της Σέγγεν, ε, τον σεβασμό της Διεθνούς Αρχής της Μη Επαναπροώθησης, τη χρηματοδότηση της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία και την ε, δήλωση της Συμβουλίου Κομισιών για την αύξηση του ρατσιστικού μίσους και της βίας κατά των προσφύγων και των μεταναστών σε όλη την Ευρώπη. Δίνω αμέσως το λόγο στο Συμβούλιο. Ο κύριος Κόντερς έχει το λόγο. Ε, Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα το επίγον πρόβλημα με το οποίο είναι αντιμέτωπη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να βρεθούν δηλαδή ε, ε, κοινέ ε, ε, λύσεις και σε επιχειρησιακό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την κρίση, την προσφυγική και τις επιπτώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο συγκεκριμένα. Το 2015 είδαμε την αύξηση άνω του 1,8 εκατομμυρίου παράνομα μεταναστών στην Ευρώπη και είχαμε 1,2 εκατομμύρια αιτήσει ασύλου. Έχουμε απώλεια ζωής, κατάχρηση από τους διακινητές της ανθρώπινης αυτής της που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, τα κράτη-μέλη. Πρέπει να είμαστε ένας ασφαλής τόπος για αυτούς που χρειάζονται προστασία. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει σημαντική πίεση που ασκείται στις κοινωνίες μας και στην ευρωπαϊκή συνεργασία. Είναι αυτό αληθές διότι σε πολλούς ε, πληθυσμούς ε, η κατάσταση δεν είναι υποέλεγχο και δεν γίνεται σωστή διαχείριση. Στα Δυτικά Βαλκάνια και στις χώρες πρώτης γραμμής είχαμε τις περισσότερες επιπτώσεις. Δεν υπάρχει δυνατότητα ένα κράτος μέλος από μόνο του να αντιμετωπίσει την κρίση. Με συνδυασμό δράσεων και με συντονισμένο τρόπο μόνο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Χρειαζόμαστε λοιπόν κοινέ ευρωπαϊκέ λύσει για να αντιμετωπίσουμε την κρίση και όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη του. Αυτό το έχουμε ξαναπεί. Ήρθε όμω η ώρα που εκπνέει ο χρόνο για να αντιμετωπίσουμε την κρίση την άνοιξη. Μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών αναμένεται ότι θα βγουν στη θάλασσα ή ακόμα και θα χάσουν τη ζωή τους κατά τη διαδρομή τα μέτρα πρέπει να είναι και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Το Συμβούλιο επιμένει να συνεχίσουμε τις συντονισμένες προσπάθειες για να διαχειριστούμε τις εισρωές, ε, την κατάσταση στα κράτη-μέλη και να εφαρμοστούν οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε υψηλό επίπεδο. Πρέπει να ενισχύσουμε φυσικά τα εξωτερικά μας σύνορα και να συνεργαστούμε με την Τουρκία έτσι ώστε οι συμφωνίες που έχουμε μαζί της να εφαρμοστούν. Να διασφαλίσουμε ότι τα hot spots ε, λειτουργούν σωστά ε, και η καταγραφή και η επιστροφή. Επίσης η ε, συνεργασία με τρίτες χώρες για την επανεισδοχή και την επιστροφή. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα για διεθνή προστασία και καταχρώνται το σύστημα. Πρέπει λοιπόν να εφαρμόζονται σωστά και οι διαδικασίε μετεγκατάσταση έτσι ώστε να παρακολουθούμε σωστά τι ροέ τη μετανάστευση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν σε επιχειρησιακό επίπεδο η Ιταλία έχει προσθέσει δύο τοποθεσίε και υπάρχει και μία τρίτη που αναμένεται να λειτουργήσει. Όπω ανέφερε η Ιταλία, όλε ε, Αφήξει ε, που γίνονται στα hot spots ε, αντιμετωπίζονται και με την δακτυλοσκόπηση και με την καταγραφή στην Ελλάδα παρόλο που έχουν γίνει σημαντικέ προσπάθειες, δεν ναι, υπάρχει πρόοδος ε, ε, παρά μόνο σε δύο τοποθεσίες. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις υπόλοιπε ε, Χαιρετίζουμε τι προσπάθειες της Ιταλίας και της Ελλάδος. Πρέπει όμως οι προσπάθειες να μην γίνονται μόνο από τα κράτη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, αλλά και από τις υπόλοιπε χώρες που θα πρέπει να απαντούν άμεσα και σωστά στις αιτήσει του Ευρωπαϊκού ε, Μηχανισμού για την Προστασία και των οργανισμών όπως ε, τη Frontex ε, και το Εάζο Για την μετεγκατάσταση, κάποια κράτη-μέλη έχουν επιτυχία κατά την μετεγκατάσταση και υπάρχει καλή κατανομή. Όμως, μόνο 400 αιτήσει ως τώρα έχουν τύχει μετεγκατάστασης σε και υπάρχουν και κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμα ορίσει θέσει. Οι αποφάσει του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου λοιπόν δεν εφαρμοζόνται από όλα τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να γίνουν περισσότερα για να αφαιρέσουμε πίεση από την Ιταλία και την Ελλάδα. Όλοι πρέπει να συμμετέχουν στη μετακατάσταση. Η Προεδρία άρχισε τι διμερείς διαβουλεύσεις με όλα τα κράτη-μέλη που ε, θα πρέπει να παρέχουν υπηρεσίε μετακατάσταση επανεκατάσταση, προσωπικού κτλ. Θα ήθελα μέσα σε αυτά τα πλαίσια να μιλήσω και για την ανθρωπιστική κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια. Υπάρχει μεγάλη απειλή. Πρέπει να υπάρχει συντονισμός έτσι ώστε να αποφύγουμε την περαιτέρω απώλεια ζωής, ειδικότερα την δέσμευση να έχουμε σωστή υποδοχή, ε, ειδικά τώρα το χειμώνα, και να λάβουμε υπόψη μας ε, και την αύξηση των ελέγχων στα διάφορα σύνορα και την μερική ή πλήρη ε, και το μερικές, μερικό ή πλήρες κλείσιμο των σύνορων στους ε, ανθρώπους που θέλουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Πρέπει να συζητήσουμε με όλες αυτές τις χώρες για να αποφύγουμε περαιτέρω ανθρωπιστικές καταστροφές. Επίσης, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, η Προεδρία θα εφαρμόσει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει και να τηρήσει τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων του Σέγγεν. Ειδικότερα μιλάμε για την εφαρμογή κανόνων όσον αφορά την αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης και, της, και των συνόρων, των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από την αίτηση να, ε, του Συμβουλίου να επανεξετάσουμε το πακέτο προτάσεων της Κομισιόν έχουμε ορίσει τα σώματα που θα κάνουν αυτή την επανεξέταση. Υπάρχει συγκεκριμένα η πρόταση για την ακτοφυλακή και συνοριοφυλακή, για τον ε, ε, συνοριακό κώδικα του Σέγγεν και για το δικαίωμα ελεύθερης κίνησης. Είναι λοιπόν το πεδίο εργασίας πολύ σημαντικό και πρέπει τα διάφορα σώματα του Κοινοβουλίου να μοιραστούν τη δουλειά για να επιταχυνθεί η εξέταση. Η Προεδρία θέλει τα κράτη-μέλη να δώσουν συγκεκριμένε προτάσει έτσι ώστε να επιτύχουμε αποτελέσματα. Ήδη έχει γίνει μεγάλη πρόεδρο. Οι Υπουργοί Εσωτερικών συζήτησαν σε άτυπη συνεδρίαση στο Άμστερνταμ την περασμένη εβδομάδα και θα επανέλθει στι 25 5 Φεβρουαρίου και στις 10 και 11 ε, Μαρτίου ε, το Συμβούλιο στο θέμα αυτό. Και θέλουμε και την συνεργασία του Κοινοβουλίου για αυτά τα θέματα, εφόσον είναι πεπισμένο ότι οι προτάσεις αυτές θα οδηγήσουν σε άμεσα αποτελέσματα το, συντομότερο δυνατόν υπό το φως της κρίσης. Τώρα για το Σέγγεν. Μετά από τις μεταναστευτικές ροές που είχαμε στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους τελευταίους μήνες, η Γερμανία, η Αυστρία, η Δανία, η Νορβηγία, η Γαλλία, η Σουηδία έχουν ε, επαναφέρει τους ελέγχους στα σύνορα. Ε, αυτό είναι ε, σύμφωνο με τον κανόνα του Σέγγεν που μιλάει για την ε, σημαντική απειλή για την εσωτερική ασφάλεια. Όμως οι εσωτερικές πιέσεις θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν μόνο αν διαχειριστούμε σωστά τα εξωτερικά σύνορα και γι' αυτό πρέπει να δούμε αυτά που όρισε το Συμβούλιο το Δεκέμβρη. Πρέπει να ε, υποστηρίξουμε την ακαιρεότητα του συστήματος Σέγγεν γιατί είναι στην καρδιά του ευρωπαϊκού εγχειρίσματος και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Κυρίες και κύριοι, η αρχή της μη επαναπροώθησης είναι ακρογωνιαίος λήθος ε, του διεθνούς μεταναστευτικού δικαίου. Και γι' αυτό ε, εκτιμώ ότι θέσατε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Συγκεκριμένα πρέπει να αφαιρθούμε στο άρθρο 33 της Σύμβασης της Γενέβης του 51 δεν πρέπει κανένα συμβαλόμενο μέρος ε, να απομακρύνει ή να χετήσει πρόσφυγα με οποιοδήποτε τρόπο από τα σύνορά του ε, όταν απειλείται η να προσφυγα με οποιοδηποτε τροπο απο τα συνορα του οταν απειλειται η ζωη του, η ελευθερία του λόγω του φίλου της θρησκείας, της εθνικότητας, ε, της συμμετοχής του σε συγκεκριμένη ομάδα ή της πολιτικής του θέσης. Η αρχή αυτή έχει ενσωματωθεί στο ευρωπαϊκό και κτημένο. Ο χάρτης ε, των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο άρθρο 18 μιλά για τη μία επαναπρόθεση στο άρθρο 2, στην παράγραφο 2 του άρθρου 19. Επίσης, η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει την δημιουργία ενός κοινού συστήματος ασύλου σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενέβης και ε, την αρχή της ε, μία επαναπρόθεσης. Υπάρχουν ε, νομοθετικά ε, μέσα που έχουν χρησιμοποιηθεί γι' αυτό τον το λόγο. Έτσι τα κράτη-μέλη πρέπει να ενσωματώσουν το κεκτημένο για το άσυλο και να σέβονται την αρχή της μία επαναπρόθεσης σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις μας όσον αφορά την ασφαλή χώρα προέλευσης αυτό ε, μπορεί να εφαρμοστεί μόνο όταν οι αρμόδιες αρχές διασφαλίσουν ότι τα άτομα που ζητούν διεθνή προστασία θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με την αρχή της μη επαναπροώθησης. Αυτή η αρχή πρέπει να μας καθοδηγεί όταν διαπραγματευόμαστε τις προτάσεις ε, της Κομισιόν για μια λίστα ασφαλών χωρών προέλευσης. Επίσης πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Συνεριακός Κώδικας του Σέγγεν ορίζει πως τα δικαιώματα των ανθρώπων και προσφύγων που ζητούν ε, διεθνή προστασία πρέπει να γίνονται σεβαστά όταν εφαρμόζουμε αυτόν τον κώδικα στα εσωτερικά και εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα για την αρχή της μια επαναπροώθηση. Επίσης πρέπει να έχουμε μια αποτελεσματική πολιτική επιστροφής για να έχουμε μια ισορροπημένη πολιτική μετανάστευση και ασύλου. Πρέπει λοιπόν το Συμβούλιο να θυμίσει πω οι πολιτικέ άμεσα και με επίγον ε, χαρακτήρα πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με το κεκτημένο. Η Προεδρία θα είναι προμηθής και πολύ συγκεκριμένη, θα συνεργαστεί για να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτά τα στοιχεία και να σεβόμαστε τα θεμελιώδη δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και την, των ανθρώπων και την αρχή της μη επαναπροώθησης. Όλα αυτά είναι σημαντικά για να βελτιώσουμε την λειτουργία του κοινού συστήματος ασύλου. Ε, αδειμονούμε να εξετάσουμε τις νέες προτάσεις της Κομισιόν όπως την αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου που θα παρουσιαστεί σύντομα. Θεωρούμε ότι αυτές οι προτάσεις λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους ακρογωνιαίους λήθους της αρχής ε, των αρχών του ασύλου όπως η μία επαναπροώθηση για να μπορέσουμε ε, να κάνουμε πιο αποτελεσματικά τα συστήματά μας στα κράτη-μέλη. Όλα τα κράτη-μέλη μοιράζονται τις ίδιες θεμελιώδεις αρχές και την ίδια ευθύνη να καλωσορίσουν με αξιοπρεπή τρόπο τους αιτούντες άσυλο. Ε, δεν πρέπει λοιπόν να υπάρχουν προκαταλήψεις και να μην βλάπτονται τα δικαιώματα των ανθρώπων που ζητούν προστασία στα σύνορα. Γι' αυτό υπάρχει μια ιδιαίτερη καταπώνηση, μια ιδιαίτερη πίεση όταν μιλάμε για τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν αυτό να συνδυάζεται σε όλα τα στάδια από την αύξηση των αιτούν των άσυλο και των προσφύγων μέχρι ακόμα και την επιστροφή αυτών που δεν έχουν δικαίωμα να παραμείνουν. Πρέπει να τονίσουμε ότι χρειάζεται αξιοπρεπής μεταχείριση και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών ε, περιλαμβάνουν και την προστασία από τα ρατσιστικά και άλλα εγκλήματα μίσους και καταδικάζουμε κάθε είδους εκδήλωση που ε, ε, περιέχει αυτό το μίσος έναντι των μεταναστών. Βέβαια υπάρχουν μικρές ομάδες που είναι υπεύθυνε για αυτά. Δεν είναι ο γενικότερος πληθυσμός της Ευρώπης ή οι αξίες της Ευρώπης αυτές. Οι περισσότεροι λοιπόν πρόσφυγες ε, από τους περισσότερους είναι ευπρόσδεκτοι. Υπάρχει ρατσισμό σε κάποια μέρη του πληθυσμού και πρέπει να ληφθεί υπόψη σοβαρά. Η βία ποτέ δεν είναι η απάντηση. Οι Υπουργοί Δικαιοσύνη τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβρη σε συνάντησή του συζήτησαν το θέμα και βρήκαν τρόπους για να αντιμετωπίσουν τα εγκλήματα μίσους, ειδικότερα κατά των μεταναστών. Έτσι πρέπει να δοθεί συγκεκριμένη σημασία στην καταγραφή αυτών των εγκλημάτων μέσα από τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, τι δικαστικέ αρχέ και να δοθεί προ προστασία στα θύματα. Πρέπει οι μετανάστες να προσέχονται γιατί δεν είναι εύκολο να προστατεύονται όταν πέφτουν θύματα αυτών των εγκλημάτων. Αυτό ήταν και ένα ουσιώδες θέμα για την Προεδρία μας. Γι' αυτό αποφασίσαμε να διοργανώσουμε σήμερα μαζί με το Συμβούλιο της Ευρώπης μία εκδήλωση για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ενσωμάτωση και τη μετανάστευση. Όταν άκουσα σήμερα το πρωί τη συζήτηση, να σας πω ότι ε, ε, κατάλαβα πως όλοι έχουν τις υποχρεώσεις τους. Οι αιτούντες άσυλο, οι, ε, μετανάστες, οι, οι οι πληθυσμοί των χωρών στους, στις οποίες μεταναστεύουν οι άνθρωποι αυτοί, όλοι έχουν τις ευθύνες τους και ανησυχίες υπάρχουν σε όλες τις κοινωνίες μας. Τέλος, τον Οκτώβριο, το Συμβούλιο ε, συμφώνησε για τις ε, δράσεις προτεραιότητας οι οποίες θα διασφαλίσουν ότι η μετανάστευση και το άσυλο θα την χάνουν όλων των διαδικασιών ε, νομικών και διοικητικών που θα διασφαλίσουν την προστασία ας πούμε των παιδιών ειδικότερα όπως ανέφερε και ο επικεφαλής του επιτελείου της Europol 10.000 ασυνόδευτα παιδιά έχουν εξαφανιστεί κατά την αύξηση του στην Ευρώπη έχουν πέσει ενδεχομένως στα χέρια του οργανωμένου και αυτό είναι ντροπή, είναι αξιοθρύνητο, πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Πρέπει λοιπόν να δούμε ακριβώς ποια είναι τα νούμερα, ποια είναι τα στοιχεία, δεν έχει ακόμα συζητηθεί στο Συμβούλιο, όμως αυτή η σκέψη μας αρρωσταίνει όλους. Τα ασυνόδευτα παιδιά είναι από τις πιο ευάλωτες ομάδες. Υπάρχουν ε, επαγγελματικέ συμμορίες που τα εκμεταλλεύονται. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνεργαστούν ώστε να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά δεν θα πέφτουν στα χέρια τους. Τέλος, όσον αφορά την Τουρκία και τη χρηματοδότησή της. Θα θυμάστε ότι οι αιγέτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, τον Οκτώβριο-Νοέμβριο 2015 δεσμεύτηκαν ε, για να προσφέρουν 3 δισεκατομμύρια προσθέτου πόρου για να υποστηρίξουν του Σύρου ε, στην Τουρκία που χρήζουν προσωρινή προστασία. Κατόπιν αυτή τη δέσμευση, η Κομισιόν στα τέλη Νοεμβρίου 2015 υιοθέτησε μια απόφαση για τη σύστηση ενό μέσου, το μέσο για την Τουρκία για να ζητήσει συντονισμό για την παροχή ανθρωπιστική βοήθεια. για τις κοινότητες σε αυτό το μέσο θα απαιτήσει να καταβληθούν 3 δισεκατομμυρία το 2016 και το 2017. Το τελικό πόσο προβλέπεται στον προπολογισμό της Ένωσης είναι περίπου 9 δισεκατομμύρια επομένως η πλήρη χρηματοδότηση τη διευκόλυνση ε, θα πιέσει όλα τα άλλα προγράμματα και δράσει προκειμένου να συμβαστούμε τι δεσμεύσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη-μέλη θα συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση τη διευκόλυνση τα δύο τρίτα του απαιτούμενου ποσό και οι συνεισφορέ των κρατών μελών ε, θα υπολογιστούν ε, βάση μια βάση κατανομή του ακαθόριστου εγχώριου εισοδήματο και το υπόλοιπο θα καταβληθεί το 2016 και 2017 από τον προπολογισμό τη Ένωση. Τα κράτη-μέλη εξετάζουν διάφορε πτυχέ σε σχέση με τη σύσταση τη διευκόλυνση, όπω ε, την διαχείριση τη διευκόλυνση ε, και ε, του όρου που πρέπει να γίνουν σεβαστοί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να είμαστε σίγουροι ότι οι προσπάθειε των κρατών μελών θα οδηγήσουν σε πραγματική υποστήριξη των προσφύγων και των κοινοτήτων του. Η Προεδρία δεσμεύεται στο να εγκρίνει γρήγορα τη διευκόλυνση και θα ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη σχετική περίοδο. Μπορείτε να βασιστείτε πάνω μας έτσι ώστε σε όλα αυτά τα θέματα θα υλοποιηθούν τα ζητήματα αυτά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό καθήκον για την Προεδρία. Μαζί με το Συμβούλιο και με την Κομισιόν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Τώρα είναι σημαντικό να τις θέσουμε και σε εφαρμογή. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κύριος Αβραμόπουλος, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του, Ευρωπαϊκού, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που δίνετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάλι την ευκαιρία να συζητήσει μαζί σας στην Ολομέλεια τη μεταναστευτική πρόκληση το συντομότερο αντιμετωπίσουμε την κατάσταση στα πλαίσια της αρχής της επιμερισμένης ευθύνης και αλληλεγγύης, τόσο καλύτερα θα πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο όλοι αναμένουν πρώτα οι άλλοι να κινηθούν και κάποιοι συμπεριφέρονται σαν επρόκειτο όλα να εξαφανιστούν αν κλείσουν για αρκετό καιρό τα μάτια τους, τότε μόνο θα χειροτερεύσουν τα πράγματα. Μία συντονισμένη και συνεπής ευρωπαϊκή προσέγγιση που θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή είναι η μόνη οδός προς τα μπρος. Πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Φεβρουαρίου, η Κομισιόν θα αναφέρει σχετικά με την εφαρμογή των δράσεων προτεραιότητας υπό την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση. Θα είμαστε ειλικρινείς και αντικειμενικοί για την μικρή πρόοδο που βλέπουμε σήμερα επί τόπου και σε σχέση με το τι θα πρέπει να γίνει τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες. Αυτό αφορά και τα κρατημέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, αλλά και όλους τους υπόλοιπους. Και τη διάσταση της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Τώρα, στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής, θα πρέπει να ενδυναμώσουμε τη συνεργασία μας με τις τρίτες χώρες για να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες και να καταπολεμήσουμε τους δουλέμπορους για να δημιουργήσουμε ασφαλείς διόδους ε, για όσους ε, το χρειάζονται και προκειμένου να επιστρέψουν όσοι δεν έχουν δικαίωμα να παραμείνουν στην Ευρώπη. Σε επίπεδο εσωτερικής πολιτικής έχουμε ακόμη περισσότερα πράγματα να κάνουμε με την κατάσταση τα hot spot, τις επιστροφές, κοινά επιχειρησιακά μέτρα που λαμβάνονται από τη Frontex και τον ΕΑΣΟ, το Γραφείο Υποστήριξης Ασύλου. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε επιχειρησιακά και οικονομικά τα κράτη-μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προς αυτό το σκοπό. Όμως, η κλίμακα του προβλήματος, η διάσταση του προβλήματος ε, των εισρώων των μεταναστών που μπαίνουν από την Ελλάδα και φτάνουν στα Δυτικά Βαλκάνια συνεχίζει χωρίς να μπορεί να αντιμετωπιστεί η Κομισιόν καταβάλει κάθε προσπάθεια για να πετύχει την εξομάλυνση της λειτουργίας του χώρου Σέγγεν και παράλληλα προετοιμάζεται για όλες τις επιλογές. Όμως, να επαναλάβω ξεκάθαρα, εδώ δεν μιλάμε για το τέλος της Σέγγεν ή για τον αποκλεισμό κάποιου κράτους μέλους. Σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης εξέδωσε μία δήλωση στον τύπο. Είναι δραματικά τα αριθμητικά στοιχεία. 13 φορές περισσότεροι άνθρωποι έχουν περάσει τη Μεσόγειο τον Ιανουάριο του 2016 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2015. 368 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο μόνο κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα αν και πολύ περισσότεροι διασώθηκαν από τις κοινέ επιχειρήσεις μας. Όμως, κάθε χαμένη ζωή είναι μια ζωή που δεν πρέπει να χάνεται. Θα πρέπει να διατηρήσουμε ακόμη και σε καιρούς κρίσης της Ευρωπαϊκής Αξίας και προσέγγιση, το να σώζουμε τις ζωές και η αρχή της μη προπρόθεσης δεν είναι υποδιαπραγμάτευση. Σήμερα η Κομισιόν υιοθέτησε μία έκθεση αξιολόγησης για την Ελλάδα αφού έλαβε θετική γνωμοδότηση από την Επιτροπή Αξιολόγησης Έγκεν. Είναι απόρριτο το έγγραφο και θα ακολουθήσουμε τους συνήθεις κανόνες για την γνωστοποίηση σε αυτό το Κοινοβούλιο έγιναν κάποιες επισκέψεις το Νοέμβριο του 2015. Βρήκαμε διάφορες ελλείψεις σε αυτή την έκθεση στην εξωτερική διαχείριση των συνόρων από την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, σημειώνουμε ότι η Ελλάδα ήδη ξεκίνησε προσπάθειες για να καλύψει αυτές τις ελλείψεις και η Κομισιόν θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ελλάδα η Ελλάδα δεν θα μείνει μόνη της για να αντιμετωπίσει τις σχετικές προκλήσεις με τις μεταναστευτικές πιέσεις. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε στενά με την Τουρκία για να μπορέσουμε να έχουμε μία τάξη στις μεταναστευτικές ροές και να ανακόψουμε την παράτυπη μετανάστευση στο Αιγαίο εφαρμόζοντας το κοινό σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Πρόσφατα, ο πρώτο αντιπρόεδρο τη Επιτροπή, ο κ. Τίμερμαν, συζήτησε με τον ε, Τούρκο μονολογό του για το πώ μπορούμε να δυναμώσουμε τη συνεργασία για να κατολμήσουμε του δουλέμπορου και να εντοπίσουμε του αριθμού των σύρων που διασχίζουν τα σύνορα. Οι ομόλογοι μας από την Τουρκία μας ενημέρωσαν για το ότι ε, άνοιξαν κάποια τμήματα της αγοράς εργασίας για να μπορούν να βρουν εργασία οι πρόσφυγες. Η Κομισιόν συνεργάζεται στενά και με τις ελληνικές και με τις τουρκικές αρχές ε, προκειμένου να επιτεχύνει τις επιστροφές στην Τουρκία βάσει της υφιστάμενης διμερούς συμφωνίας περιμένοντας να τεθεί πλήρως ισχύ και η Ευρωπαϊκή Συμφωνία με την Τουρκία. Διερευνούμε με την Ελλάδα ποιε ε, περαιτέρω δράσει υποστήριξη μπορούν να παραχθούν για να επιστραφούν οι μετανάστε που δεν έχουν δικαίωμα να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να επενθυμίσω όπως θα τονίσει και ο Πίτροπος Χάν, ότι η Τουρκία κάνει σημαντικές προσπάθειες για να φιλοξενήσει πάνω από 2,75 εκατομμύρια πρόσφυγες με κόστος πάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα υποστηρίζουμε ε, την Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να παρέχει χρηματοοικονομική βοήθεια στο ποσό των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα να, να δίνει αυτή τη βοήθεια το 2016 και το 2017 για να παρέσχει ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια αλλά και άλλη βοήθεια στους πρόσφυγες. Στη συνέχεια έχουμε την οδό των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτή είναι μια κύρια προτεραιότητα για την Κομισιόν και οργανώνουμε συντονιστικές συναντήσεις. Οι μετανάστες πάντοτε θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να ζητήσουν, να κάνουν αίτηση για διεθνή προστασία. Αλλά αν επιλέξουν να μην το πράξουν ή αν προκύψει ότι δεν χρειάζονται προστασία, τότε θα πρέπει να επιστραφούν ταχύτατα στις χώρες προελευσής τους ή σε χώρες διάλευσης. Αυτό θα γίνεται πάντοτε βάση της αρχής της μη επαναπροώθησης και δυνάμη του διεθνούς δικαίου. Η αρχή της μη επαναπροώθησης ε, είναι μια ασφαλιστική δικλίδα και νομική υποχρέωση που οφείλουμε σε κάθε πρόσφυγα. Παρόλα αυτά, αυτή η αρχή δεν είναι ασύμβατη με την προσπαθία μας να διασφαλίσουμε πιο αποτελεσματικές επιστροφές των παράτυπων μεταναστών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει συστηματικά και γρήγορα να επιστρέψουμε όσους δεν χρήζουν διεθνούς προστασίες. Αν θέλουμε να οικοδομήσουμε δημόσια εμπιστοσύνη και να επικεντρώσουμε τις προσπαθίες μας στο πώς θα υποδεχτούμε τους πραγματικούς πρόσφυγες. Αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να προωθήσουμε και την παροχή προστασίας σε όσους τη χρειάζονται, όπως και τα μέτρα επαναγκατάστασης. Όσο πιο αποτελεσματική και αξιόπιστη υποστήριξη δίνουμε σε όσους χρήζουν διεθνούς προστασίας, τόσο λιγότερο θα αισθάνονται την ανάγκη να ακολουθήσουν την οδό της παράτυπης μετανάστευσης. Και να κλείσω με ένα σύντομο σχόλιο για την άνοδο της ξενοφοβίας και του ρατσισμού απέναντι στους μετανάστες και τους πρόσφυγες είναι η κύρια ανησυχία μου. Και δεν ε, ήταν έκπληξη για μένα. Η Κομισιόν καταδικάζει ανεπιφύλακτα ε, αυτό που φαίνεται ήταν μαζικές ε, σεξουαλικές επιθέσεις κατά γυναικών στην κολονία την παραμονή πρωτοχρονιά. Όμως είναι πολύ απλουστευτικό να συμπεράνει κανείς ότι όλοι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες αποτελούν απειλή για τη δημοσία τάξη μας. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο και όσοι φεύγουν για να γλιτώσουν από τον πόλεμο και τη φρίκη του πολέμου χρήζουν περισσότερο σεβασμό από οποιοδήποτε άλλο. Επομένως, καταδικάζουμε έντονα κάθε εκδήλωση ρατσισμού και την δημόσια παρότρινση σε μίσος, ξενοφοβία και ρατσιστικές πράξεις. Θα χρειαστεί να ενδυναμώσουμε τις προσπαθίες μας και εδώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια κρίση πρωτόγνωρη. Είτε θα είμαστε σταθεροί και θα βρούμε λύσεις σύμφωνες με τις αξίες μας ή θα αλλάξει η Ευρώπη και θα επιστρέψουμε σε ένα παρελθόν που κανείς δεν θέλει να ξαναβιώσει. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Και τώρα ο Βέμπερ, εκ μέρου του ΕΛΚ για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, Πρόεδρε της Επιτροπής, Πρόεδρε του Συμβολίου. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την Κομισιόν γιατί τα θέματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο τραπέζι Ήρθαν με μεγάλη ε, ταχύτητα από την κοσμισο... με την Κομισιόν η συνεργασία με την ε, Τουρκία, οι τρίτες χώρες, η Frontex, ε, όλες οι λύσεις αυτές είναι κείμενα που η Κομισιόν με μεγάλη ταχύτητα επεξεργάστηκε. Δεν έχουμε πρόβλημα σε επίπεδο ιδιών. Έχουμε ένα μπλοκάρισμα στο Συμβούλιο και εδώ στο Κοινοβούλιο που το είδαμε σήμερα το μεσημέρι. Θα δούμε λοιπόν ότι υπάρχει ανάγκη αλληλεγγύης ε, στην Ευρώπη. Πρέπει να ε, το καταλάβουν και από την αριστερή πλευρά. Ε, πρέπει να ενεργοποιήσουμε τα σύνορα, είπε κάποιος, και πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Υπάρχει αυτό το μπλοκάρισμα. Πρέπει ακριβώς να ξεπεράσουμε τέτοια προβλήματα. Αν έχουν ε, στο μεταξύ 50.000 άνθρωποι χάσει τη ζωή τους στην ε, Συρία, μεταξύ αυτών 40.000 παιδιά, καταλαβαίνετε ότι εμείς αυτή την Ήπειρο από το βορρά μέχρι το νότο πρέπει να, ε, βοηθήσουμε. Έχουμε 60 εκατομμύρια ανθρώπους που αυτή τη στιγμή είναι υποδίωξη στον κόσμο εκατομμύρια καταλαβαίνετε. Δεν λειτουργεί το πράγμα αλλιώς ε, και οι δύο πλευρές ανήκουν η μία στην άλλη. Πρέπει λοιπόν να σταματήσει αυτό το μπλοκάρισμα. Ο δρόμος είναι σύντομος. Πρέπει να κατανοήσουμε ένα τον άλλον και να συνεργαστούμε. Και πολλά παίζονται, δεν είναι μόνο το Σέγγεν. Φυσικά η Ευρώπη, αν δεν είναι ενωμένη σε αυτό το θέμα, ε, θα έχουμε όλο και περισσότερα σουηδικά και δανέζικα παραδείγματα, θα έχουμε όλο και περισσότερους ελέγχους στα σύνορα. Και αυτό είναι δυστυχώς πάρα πολλά. Αυτή, αυτό το μπλοκάρισμα λοιπόν πρέπει να σταματήσει, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι. Τις τελευταίες ε, δεκαετίες ε, κάναμε τη δουλειά μας ε, με τέτοιο τρόπο ώστε τελικά να ξεπεράσουμε μέσα από την επανένωση της Δύσης και της Ανατολής την αντιπαράθεση που υπήρχε. Είχαμε ανάπτυξη, είχαμε την διάσκεψη για το κλίμα στο Παρίσι που είναι ένα πρότυπο για τον κόσμο. Αυτές οι ιστορικές κατακτήσεις ε, είναι κάτι που έφεραν εδώ οι πολιτικοί και πρέπει ε, πραγματικά αυτό που έγινε στο παρελθόν να θεωρηθεί ιστορικό παράδειγμα και στο και να ε, σταματήσουμε οποιαδήποτε μορφή ανυπαράθεσης όπως έγινε και τότε μεταξύ ημών. Πρέπει λοιπόν να απαντήσουμε σε αυτό το ζήτημα. Πρέπει να διασφαλίσουμε τα σύνορα, όπως ανέφερα. Ε, αυτό πρέπει να το κάνουμε σε συνεργασία με το Συμβούλιο. Αυτό είναι κάτι ε, ε, που κανείς δεν αρνείται. Πρέπει να, οι άνθρωποι που δεν έχουν βίζα να μην μπορούν να μπαίνουν. Πρέπει να ενισχύσουμε και τις αρχές, τους οργανισμούς. Όταν η Frontex λέει ότι χρειάζονται άνθρωποι της Frontex στην Ελλάδα, ότι πρέπει ε, να υπάρχουν ε, ανταλλαγή πληροφοριών που η Frontex δεν μπορεί να έχει γιατί εμείς οι νομοθέτες δεν καταφέραμε να δώσουμε αυτό το δικαίωμα στη Frontex. Ε, αυτά πρέπει να σταματήσουμε. Πρέπει να εμπιστευόμαστε τις αρχές μας ότι θα προστατεύσουν τους πολίτες και όχι ότι θα κάνουν το αντίθετο. Πραγματικά και όσον αφορά την κολονία, οποιαδήποτε μορφή βίας είναι καταδικαστή ακόμα και κατά των, και κατά των προσφύγων φυσικά και πρέπει ε, να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν εμφύλιο πόλεμο στη χώρα τους. Περιμένουμε οι άνθρωποι αυτοί βέβαια να μην εκμεταλλεύονται τη φιλοξενήμα μας και να σέβονται την κουλτούρα της χώρας μας. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι όταν κάποιος ε, παραβιάζει τους νόμους ε, και την κουλτούρα της χώρας φιλοξενίας ε, θα πρέπει να φεύγει από αυτή τη χώρα. Αυτές είναι οι αρχές που σέβονται οι δικοί μας πολίτες και δεν τίθενται υποσυζήτηση. Ευχαριστώ. Τώρα, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριος Πιτέλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με μεγάλο ρεαλισμό και ανησυχία θα πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς φυσάει κακός άνεμος στην Ευρώπη. Οι επιθέσεις των νεοναζί στη Γερμανία τις ε, τελευταίες μέρες ε, και οι ντροπιαστικέ προκλήσεις κάποιων πολιτικών να πυροβολούνται οι πρόσφυγες, ακόμη και τα παιδιά. Όλα αυτά μας λένε ότι ε, ουσιαστικά ένας ιός απλώνεται στην Ευρώπη, ο ιός του φόβου και εγώ ουσιαστικά δεν συμφωνώ με την ιστορία του μαστιγίου και του καρότου ε, σε σχέση με τους ε, πρόσφυγες. Μόνο για υποδοχή πρέπει να μιλάμε, γιατί δεν πρόκειται για ανθρώπους που θέλουν να έλθουν εδώ ε, για να στραφούν κατά της δικής μας ζωής. Πρόκειται απλώς για ανθρώπους που ξεφεύγουν από τον πόλεμο. Μιλάμε τις τελευταίες μέρες για τη Σέγγεν, για το σεβασμό της ανθρώπινης ζωής, για το δικαίωμα στην αστροπιστική βοήθεια. Δεν μπορούμε να συζητούμε μόνο εδώ για νομοθετικούς φακέλους στο Κοινοβούλιο. Πρέπει να, συζητάμε και για τις αξίες. Γιατί εμείς ανήκουμε σε μια κοινότητα αξιών. Δεν, υπάρχουν πια αυτές οι αξίες, δεν υπάρχει πλέον και αυτή η κοινότητα. Γιατί αυτοί οι θεσμοί έχουν νόημα μόνο όταν προωθούν και σέβονται τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και εγώ κάνω αυτή την ομιλία εδώ και αναφέρθηκαν ε, και οι προλαλήσοντες στα 10.000 παιδιά που αγνοούνται. Είναι δυνατόν κανείς να μην μιλά γι' αυτό και να μην το αναφερόμαστε. Μιλάνε μόνο για κίνδυνο. Ε, και ποιο κίνδυνο θέτουν οι πρόσφυγες. Αυτό πρέπει να νικήσουμε, αυτό το καταραμένο φόβο που δένει τα χέρια όσων πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Γιατί εδώ το παραδέχτηκε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα πράγματα. Συμφωνούμε κύριε Βέμπερ ότι πρέπει να ενισχύσουμε τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα και για την ταυτοποίηση. Συμφωνούμε και για τη μετεγκατάσταση. Τι εμποδίζει αυτό το σύστημα να λειτουργήσει, να σας το πω εγώ, ο φόβος. Ο φόβος εμποδίζει που ουσιαστικά γιγαντώνεται, διευρύνεται, τροφοδοτείται όλους αυτούς τους μήνες. Αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνος που βιώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και διαλύει την κοινότητα των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το θέμα είναι θεμελιώδες Διαφορετικά δεν θα λειτουργήσουν τα πράγματα ποτέ. Αν δεν επιστρέψουμε εδώ και αν δεν πούμε στους επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων μη φοβάστε δεν θα χάσετε ψήφους, δεν θα χάσετε συνενέσεις αν δείξετε ότι λειτουργεί το σύστημα και μπορεί το σύστημα να λειτουργήσει. Και προσοχή, δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο επιλύεται μέσα σε λίγους μήνες. Ήδη έχουμε και κάποιες ροές που αφορούν τη Φιλανδία, την Ανατολική Ευρώπη και όλες τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ε, θα έχουμε νέες ροές την Άνοιξη. Έτσι λοιπόν ή θα συστήσουμε αυτό το σύστημα και θα λειτουργήσει ή θα αποτύχουμε. Γι' αυτό κάνω αυτή την έκκληση. Δεν αναφέρομαι σε την ΤΑΔΕ ή τη ΔΥΝΑ νομοθεσία. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε στο αν συμφωνούμε στις αξίες μας για το αν είμαστε Ευρωπαίοι και αν είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. E Ο κύριος ε, Καμάλεκ, εκ των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ. Άλλη μια συζήτηση για πρόσφυγες και μετανάστες. Η άνοιξη συνήθως είναι πηγή αισιοδοξία. Αυτή όμως δεν μας επιτρέπεται γιατί καθώς λιώνουν τα χιόνια η κρίση οξύνεται. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε λύσεις αποτελεσματικές. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι όλοι από οποιαδήποτε χώρα μπορούν να εισέλθουν. Άλλοι λένε να προσέξουμε τα σύνορά μας. Άλλοι λένε να σφραγίσουμε τα σύνορά μας και να κάνουμε την Ευρώπη φρούριο. Ας αφήσουμε πίσω την πολιτική αυτή συζήτηση και ας κοιτάξουμε το πρόβλημα. Γνωρίζω ότι ο κύριος Προειδοποιεί τον τύπο για τα σχόλια της ομάδας μου. Λοιπόν, να τα δούμε αυτά τα σχόλια. Να τα συζητήσουμε. Θα τα δούμε σήμερα το απόγευμα. Όμως, πραγματικά απογοητεύομαι, διότι βάζετε την πολιτική πάνω από την εξέβρεση λύσης. Η ομάδα μου είναι συνεπής. Ήταν ανέκαθεν συνεπής από την έναρξη της κρίσης. Δεν θα ξαναγράψουμε τους κανόνες. Έχουμε μπροστά μας πολύ λίγο χρόνο, εβδομάδες και μόνο, να βοηθήσουμε όσους χρειάζονται βοήθεια και να προστατεύσουμε τους πολίτες μας. Όμω θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε μόνο όταν οι κανόνε είναι σαφείς και αυστηροί. Οι κανόνε του Σέγγι λένε ότι τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προστατεύονται. Εάν τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, να τα βοηθήσουμε μέσω τη Frontex. Όμω, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε βοήθεια σε δημοκρατικά εκλεγμένε κυβερνήσει. Εν τούτης, εάν κάποιο δεν μπορεί να συμμορφωθεί με του κανόνε που έχει αποδεχθεί βάσει Σέγγεν και Δουβλίνου, τότε είναι εκτό παιχνιδιού. Και οι, οι κανόνες, το ξαναλέω, αποδίδουν, λειτουργούν μόνο όταν τηρούνται οι συμφωνίες. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να φροντίσουμε η Τουρκία που παλεύει με τους πρόσφυγες να μην θεωρείται πλέον χώρα διέλευση. Τι γίνεται με το Πακιστάν. Το Πακιστάν υπέγραψε συμφωνία επανεισδοχή. Πού πάει αυτή η συμφωνία. Λοιπόν, α γίνουμε πιο αυστηροί με αυτές τις χώρες για να τηρήσουν και αυτέ τι υποχρεώσει του. Ο Δουβλίνο είναι σαφή. Στι περισσότερε περιπτώσει, η πρώτη ασφαλή χώρα είναι η χώρα στην οποία κάποιοι υποβάλλουν αίτηση. Όμω απέτυχε το Δουβλίνο. Διότι κάποιοι, ένα ηγέτη, άνοιξε τη χώρα του σε όλου. Όχι μόνο αυτού που προσπαθούν να γλιτώσουν από τον πόλεμο, αλλά και σε αυτού που ζητούν μια καλύτερη ζωή. Και απέτυχε διότι οι πρώτε χώρε, οι οποίε φτάνουν οι πρόσφυγε και οι μετανάστε, δεν τα βγάζουν πέρα. Το Δουβλίνο δεν χρειάζεται να, να συγγραφεί από την αρχή. Χρειάζεται τροποποιήσει για να αποδώσει και πρέπει να φροντίσουμε να μείνουν στις χώρες που, τους, που μπορούν να τους παράσχουν άσυλο. Όμως πρέπει να σταθεροποιήσουμε και κατεπηγόντως την κατάσταση βραχυπρόθεσμα. Λοιπόν, να συμφωνήσουμε ποιοι μπορούν να δεχθούν προσφύγες και πόσοι. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε οτιδήποτε. Ας ε, αφήσουμε τις χώρες που δεν μπορούν να δεχθούν πρόσφυγες να βοηθήσουν με χρήματα ή με προσωπικό. Κανείς όμως δεν μπορεί να ανύπτει τα σχήρα του και να περιμένει οι άλλοι και μόνο να λύσουν το πρόβλημα. Η Μεσόγειος είναι περιοχή διέλευσης. Λοιπόν, η Ιταλία και η Μάλτα δεν μπορούν να παλεύουν μόνες τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδείξει τις ικανότητές της. Ας αποδείξουμε ότι μπορούμε να είμαστε και ρεαλιστές, ότι μπορούμε να αναλάβουμε δράση για να υλοποιήσουμε στην πράξη τους κανόνες μας. Λοιπόν, ας μην ξαναγράψουμε τους κανόνες από την αρχή. Ας τους εφαρμόσουμε, ας εφαρμόσουμε τους κανόνες που ήδη διαθέτουμε και συνεργαστούμε για να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση και ας εστιάσουμε τις προσπαθειές μας στην βοήθεια αυτών που πραγματικά την χρειάζονται, που προσπαθούν να γλιτώσουν τη ζωή τους από τον πόλεμο. Να τους βοηθήσουμε βραχυπρόθεσμα, μέσοπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος εκ μέρους των κ. Φερχόφστατ. και κύριοι, Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τον κύριο Κούντερ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, διότι διορθώσετε τόσο είπε ο του κομματό σα που πρότεινε υποτίθεται ένα σχέδιο. Ε, Εσεί ε, το ακυρώσατε και χαίρομαι πάρα πολύ με την δήλωσή σα. Δεν είπατε ρητό, αλλά ετεύχετε υπέρ τη αρχή τη μη επαναπρόθεση και είπατε ότι οποιοδήποτε πρόσφυγας φτάνει στα σύνορά μα, πρέπει να τη χάνει τέτοια αντιμετώπιση ως πρόσφυγας που είχε ανάγκη προστασία. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν που διατυπώσατε αυτή την αρχή. Κύριε Καμάλ, πριν πω οτιδήποτε μου επιτεθήκατε. Κάνα πρόβλημα. Αλλά ξέρετε, απογοητεύτηκα. Γιατί η πρόεδρος τη ε, ομάδα ε, Ελευθερία και Εμεί Δημοκρατία, είπε κάτι το οποίο είναι ντροπή για τη δημοκρατία. Είπε δηλαδή βασικά ότι μπορούμε να πυροβολούμε ανθρώπου που ζητούν σωτηρία. Και μετά είπε, ναι, να το δούμε. Όχι, όχι να το δούμε. Να καταδικάσετε τη δήλωση τη EFT, τη ομάδα Ευρωπαϊκή και Εμεί Δημοκρατία. Και τρίτον, κύριε Βραμμαπουλέ, και το λέω και προ τον κύριο Κούντερ, ε, για την ουσία. Πιστεύω ότι έχουμε πάρει λάθος δρόμο. Δεν πρόκειται να λύσουμε έτσι το πρόβλημα. Διότι οι προτάσεις δεν αποδίδουν. Λέει και η Κομισιόν, ναι, οι Έλληνες βελτιώνονται. Κοιτάξτε τη δική σας αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δύο, τρεις μέρες πριν, την περασμένη εβδομάδα, εσείς προέβητε σε αξιολόγηση, αναλύσατε τους ε, ελέγχου των σύνορων μεταξύ Ελλάδο και Τουρκία. Και το πράγμα δεν αποδίδει. Κανεί δεν καταγράφεται και αυτό είναι και ο λόγο που υπάρχουν τόσε χιλιάδε νέοι πρόσφυγε. Α τα δει αυτά η Europol, α αναλύσει του αριθμού, τα αριθμητικά στοιχεία, διότι μετά οι άνθρωποι δεν την χάνουν αξιοπρεπούς μεταχείριση. μαζεύονται και ένα σωρό μετανάστες, όχι πρόσφυγες στα σύνορα. Το πράγμα δεν αποδίδει. Η πρόταση μας λοιπόν είναι πολύ απλή. Χρησιμοποιήστε το άρθρο 78 της συνθήκης, το οποίο σας δίνει την δυνατότητα να λάβετε κατεπήγοντα μέτρα στα σύνορα και να δημιουργήσετε δύναμη ταχεία αντίδρασης στα ευρωπαϊκά σύνορα για να προστατεύσετε τα ευρωπαϊκά σύνορα. Η Ευρώπη να το κάνει αυτό. Ε, όχι, ναι, θα δούμε βελτιώσεις, θα περιμένουμε βελτιώσεις, θα κάνουμε συστάσεις στην ελληνική κυβέρνηση. Πέρασαν ήδη τρεις μήνες. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων στα ελληνικά σύνορα. Αξιοποιήστε λοιπόν το άρθρο 78. Κύριε Κούντερ, είναι μια απόφαση που μπορεί να ληφθεί με ενισχυμένη με πλειοψηφία στις 18 Φεβρουαρίου ήδη. Αντί να καθόμαστε να ασχολούμαστε με τον κύριο Κάμερον. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε σύγκριση με τα αιτήματα της Βρετανικής κυβέρνησης. Αυτό πρέπει να κάνετε. Αν δεν το κάνετε, αυτό το χάλι θα συνεχιστεί. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να δώσει την απάντηση. Η Ευρώπη πρέπει να οργανώσει τα κέντρα υποδοχή, τα σύνορα με την Τουρκία. Μαζί φυσικά με τι ελληνικέ αρχέ. Και δεν μπορούν να κόπτονται οι Έλληνε περί θεμάτων κυριαρχία. Δεν είναι μόνο η ευρωπαϊκή κυριαρχία. Δεν μόνο συγγνώμη, η ελληνική κυριαρχία, είναι και η ευρωπαϊκή κυριαρχία. Λοιπόν, αυτό πρέπει να κάνετε. Στι 18 Φεβρουαρίου η Κομισιόν και το Συμβούλιο να πάρουν μια απόφαση να βελτιώσουν τι συνθήκε στα στρατόπεδα υποδοχή των προσφύγων. Μιλάμε για ανθρώπους που πρέπει να περάσουν με 7 δολάρια το μήνα. Πώς θα βρουν φαγητό για τα παιδιά τους. Πώς θα ντυθούν με 7 δολάρια το μήνα. 7 δολάρια το μήνα. Αντί να δώσουμε 3 δισεκατομμύρια στον Ερντογάν, χρησιμοποιήστε τα χρήματα αυτά για να βοηθήσετε τα στρατόπεδα των προσφύγων. Οργανώστε τα. Βελτιώστε τα. Φέρτε τα Ηνωμένα Έθνη. Και με βεβαίω ότι αν του δώσουμε κάτι παραπάνω, όχι χιλιάδες, αλλά 70, 80, 100, 200, τότε αυτές οι οικογένειες θα μπορέσουν με τα χρήματα αυτά να φροντίσουν τις οικογένειές τους. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν τίποτα. Δεν έχουν τα στοιχειώδη, να αγοράσουν φαγητό καθημερινά, να αγοράσουν ρούχα. Αυτό είναι το δεύτερο λοιπόν που πρέπει να κάνουμε. Και μην δώστε, επαναλαμβάνω, τα 3 εκατομμύρια στην τουρκική κυβέρνηση. Όχι, βοηθήστε του πρόσφυγε στα στρατόπεδα που ζουν. αν τα δώστε, να χρησιμοποιηθούν για τα στρατόπεδα στην Τουρκία, στο Λίβανο και αλλού. Περιμένουμε μήνε για μια απόφαση και τώρα, ε, αν πάρουμε μια απόφαση το Φεβρουάριο, πότε, το Μάρτιο. Τώρα ή ποτέ, κυρίε και κύριοι. Τώρα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση για την κρίση. Αποδείξτε ότι η Ευρώπη μπορεί. Μην περιμένετε τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη θα κάνουν όσο λιγότερα μπορούν. Αύριο θα κλείσουν τα σύνορα, Μεθαύριο θα πούνε ναι, ας αλλάξουμε το ένα ή το άλλο, να τροποποιήσουμε τον κανονισμό για τους ετούντε άσυλο κλπ. Όχι. Η Ευρώπη να αποδείξει ότι θέλει και μπορεί. Ευχαριστώ. Au nom de la GUE, Monsieur Papadimoulis. Papadimoulis από την e. Μικρό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης κύριε Κούντερς και κύριε Αβραμόπουλε απαιτεί ισχυρότερη και αποτελεσματικότερη ευρωπαϊκή συνεργασία όχι μια ευρώπη la carte που θέλει τις αγροτικές επιδοτήσεις ή τα διαρθρωτικά ταμεία για υποδομές για την πολωνία για την ουγγαρία για τη σλοβακία αλλά δεν θέλει την εφαρμογή των κοινών ευρωπαϊκών αποφάσεων για την αντιμετώπιση του προσφυγικού. και φυσικά μια τέτοια ευρώπη που σέβεται την υπογραφή της στη σύμβαση της γενέβης των ηνωμένων εθνών δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με την επιστροφή στους εθνικισμούς την ξενοφοβία τον ρατσισμό και τη διάλυση της ευρώπης που επιδιώκουν οι εξτρεμιστές της άκρας δεξιάς. η ελλάδα και η ιταλία χρειάζονται περισσότερη αλληλεγγύη και ευρωπαϊκή βοήθεια για τον έλεγχο των ευρωπαϊκών εξωτερικών συνόρων και όχι να μετατρέπονται σε εύκολους αποδιοπομπαίους τράγους. Πριν δύο μέρες διάβασα την εξής φράση όποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρισκόταν στη θέση της Ελλάδας θα είχε τα ίδια προβλήματα. Η Ελλάδα έχει αιτηθεί βοήθεια και πρέπει να την υποστηρίξουμε. Τα είπε ο Φαμπρίς Λεγκερή, Γενικός Διευθυντής της Frontex πριν τέσσερις μήνες σε αυτή την αίθουσα κάποιος είπε «Ευρώπη είναι ο φούρναριστικό που μοιράζει ψωμί στους πρόσφυγες και οι Ευρωπαίοι πολίτες που υποδέχονται τους πρόσφυγες στο σταθμό του Μονάχου». Ήταν ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Αυτό πρέπει να είναι Ευρώπη και όχι η πρόεδρος του ΑΕΦΔ, κύριε Καμάλ που ζητά να πυροβολούνται στα σύνορα οι πρόσφυγες και όχι οι φασίστες ακροδεξιοί που κυνηγούν με λαψούς στο σταθμό της Κοπενχάγης. Και επειδή διάφοροι ανεκάλυψαν ότι το πρόβλημα είναι η Σέγγεν και ζητούν κατάργηση της Σέγγεν ή μικρότερη Σέγγεν. Μικρότερη Σέγγεν σημαίνει καθόλου Σέγγεν και μια κατάρρευση της Σέγγεν θα είναι τεράστια ζημιά και για τη δημοκρατία και για τους πρόσφυγες και για την οικονομία η επαναφορά των συνοριακών ελέγχων θα είναι μια καταστροφή για την ευρώπη. και επειδή πολλοί μιλούν για εφαρμογή it's the implementation stupid αποφάσισαν συμβούλιο και επιτροπή το σεπτέμβριο με την κατάσταση 160.000 προσφύγων αναλογικά ποια είναι η εφαρμογή 400 μας το είπατε και σήμερα μπορεί να προχωρήσει έτσι η ευρώπη. βεβαίως η ελλάδα έχει κάνει ήδη σημαντική πρόοδο τώρα που μιλάμε σε σχέση με την έκθεση των αρχών του νοεμβρίου και είμαστε βέβαιοι ότι τον μάρτιο όταν θα αξιολογήσετε θα έχουμε ολοκληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα. Αλλά πρέπει και εσείς να τηρήσετε τις δεσμεύσεις κύριοι του Συμβουλίου και κύριοι της Κομισιόν για να έχουμε περισσότερη αποτελεσματική και δημοκρατική ευρώπη που να λύνει το πρόβλημα το προσφυγικό που δεν είναι ελληνικό ή ιταλικό πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. αλλιώς θα νικήσει η ξενοφοβία ο ρατσισμός η άκρα δεξιά η επιστροφή στους εθνικισμούς και η διάλυση της ευρώπης. σας ευχαριστώ. Η κυρία Άρμς από τους πρασένους, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να παραθέσω ένα θετικό στοιχείο έναντι των όλων όσων συζητιούνται εδώ. Όχι μόνο σε εμά στη Γερμανία, στην πατρίδα και στην πιο στενή μου πατρίδα, στην περιφέρειά μου, αλλά και στα ελληνικά νησιά, στην Ουγγαρία, στην Στοκχόλμη και στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία. Πραγματικά χιλιάδες πολιτείς εργάζονται εθελοντικά, εθελοντικά για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση η προσφυγική εισαγωγικά, η μεταναστευτική εισαγωγικά. Αυτό που ξεκίνησε με την Άγγελα Μέρκελ τον προηγούμενο Σεπτέμβριο θεωρώ ότι οδήγησε στην ενίσχυση της ε, Ευρωπαϊκής Κοινωνίας των Πολιτών και οι πολίτες κάνουν τη δουλειά τους με την επίγνωση, κύριε συνάδελφε Βέμπερ, όλων των προβλημάτων, όλων των θεμάτων που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αλλά αυτό το κάνουν επειδή θέλουν να ανταπεξέλθουν σε αυτή την πρόκληση. Και το φαινόμενο το οποίο βλέπω όλο και πιο πολύ από συζήτηση σε συζήτηση είναι ότι η κοινωνία των πολιτών αυτή χωρίς πάθος πράττει αυτά που πράττει, ενώ η πολιτική συζήτηση διέπεται βαθύτατα από τέτοια πάθη και ιδιαίτερο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και πραγματικά αυτοί οι πολίτες οι οποίοι δεσμεύονται και δραστηριοποιούνται φρύτουν για το γεγονός ότι το Συμβούλιο φαίνεται και παρουσιάζεται όλο ένα και πιο πολύ ως ένα Συμβούλιο το οποίο μιλάει υπέρ της φυγής. Αυτή η προδοσία λοιπόν της ε, κοινωνίας των πολιτών βαρύνει κάθε μέρα όλο και πιο πολύ. Κυρίες και κύριοι, το γεγονός ότι όλοι ε, μείναμε έκπληκτοι από την απόφαση της Άγγελα Μέρκελ τον περασμένο Σεπτέμβριο είναι ένα στοιχείο. Αλλά ένα άλλο στοιχείο είναι το ότι έχουμε μπει σε μια φάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου έχουμε σταματήσει να αποφεύγουμε πολύ απλά τα προβλήματα που μας περιτριγυρίζουν. Η κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Νότο και στην Ανατολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρόκειται να διαλυθεί έτσι εύκολη, εύκολα. Στο Μίνσκ, στη Συρία, δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσουν τα πράγματα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ως Ευρωπαίοι θα πρέπει να προσανατολιστούμε προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών τα οποία συζητάμε ως ε, ιδιαίτερα φλέγοντα και μάλιστα την μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση. Η δική μου ομάδα ζητά λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Συμβούλιο να κάνει και να επικεντρωθεί σε τέσσερα μεγάλα βήματα και επιτέλους να έχει κάποιο αποτέλεσμα, να μπορέσουν να ακολουθήσουν και οι πράξεις τα λόγια, γιατί από τη μία πρέπει να πείσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες, από την άλλη όμως θα πρέπει να βοηθήσουμε και τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κρίση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι υποδίωξη. Θεωρούμε ότι για παράδειγμα η συμφωνία Επανεγκατάσταση με τον ΟΗΕ πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα τα οποία δεν πρέπει να τα συζητάμε πλέον αλλά να τα εφαρμόσουμε. Είμαστε πεπισμένοι ότι οι επενδύσει για την Τουρκία για παράδειγμα ότι θα πρέπει να έχουν πιο μεγάλες και φιλόδοξες διαστάσεις και αυτά που λέει ο κ. Φερχόφστατ κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν μπορούμε τους πρόσφυγες να τους ε, κρατάμε ίσα ίσα στη ζωή. Όχι, θα πρέπει να τους δώσουμε μια πραγματική ζωή. Και να το πάρουμε στα σοβαρά. Όποιο δεν πάρει στα σοβαρά θα να του δώσει μια πραγματική ζωή, νομίζω ότι δεν θα καταφέρει να αντιμετωπίσει την κρίση σοβαρά. Και πραγματικά. Είμαστε βέβαιοι ότι η κατανομή των ε, μεταναστών στην Ευρώπη, στο εσωτερικό της Ευρώπης, θα πρέπει επιτέλους να γίνει με αλληλέγγυο τρόπο. Και αναμένουμε από το Συμβούλιο να κινηθεί κάτι, γιατί άλλως δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και τέταρτο σημείο αφορά τα σύνορα. Και εμείς είμαστε υπέρ της καλύτερης διαχείρισης των σύνορων και εμείς είμαστε υπέρ της ε, ανάληψης κοινή ευθύνη μαζί με την Ελλάδα. Αλλά ξέρουμε ότι αυτά τα σύνορα, τα εξωτερικά σύνορα, δεν μπορούν να είναι ερμητικά κλειστά. Και μας προκαλεί φρίκη η συζήτηση για να πυροβολούνται άνθρωποι. Και τότε οι συζητήσεις αυτές γίνονται μάλιστα στη Γερμανία. Και στο σημείο λοιπόν αυτό πιστεύουμε ότι έγινε η πρόκληση. Και σε ό,τι αφορά και όσους βρίσκονται στο δεξί φάσμα της Ευρώπης και χρησιμοποιούν και εκμεταλλεύονται αυτή τη συζήτηση των προσφύγων και του Σέγγεν για να καταστρέψουν την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Γιατί το ότι ξεπεράστηκαν τα σύνορα σημαίνει ότι ξεπεράστηκε ο πόλεμος, η καταστροφή. Όποιος θέλει να αρθώσει πάλι σύνορα στην Ευρώπη θα επανέλθει στις καταστροφές του τελευταίου αιώνα και αυτό θα πρέπει να βρει αντιμέτωπη στεναρά την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Όλοι ξεπερνούν λίγο το χρόνο τους, αλλά σας παρακαλώ να το λάβετε υπόψη σας. Φεράρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε από το EFDD. Η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση των μεταναστευτικών ροών απέτυχε. Έχουμε μια τεράστια πρόκληση μπροστά μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει τις πραγματικές της ικανότητες. Είναι ακατάλληλη η απάντησή της, συντίθεται από έλλειψη αλληλεγγύης και από εθνικούς εγωισμούς. Ασχολείται με τα αποτελέσματα και όχι με τις αιτίε. Ποτέ δεν συζητάμε τις αιτίε. Βλέπουμε ότι από τη μία μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες συνεισφέρουν στη δημιουργία των προβλημάτων, ρίχνουν όπλα, συμμετέχουν σε σειράξεις και προκαλούν τις μεταναστευτικές αυτές ροές. Από την άλλη ε, μπλοκάρουν, ε, ανορθώνοντας εμπόδια στις μεταναστευτικές ροές, εμπόδια διαφόρων τύπων. Υποπιτέλα στις αξίες. Ε, τότε πείτε το στην κυβέρνησή σας. Πείτε τους να σταματήσουν να πουλούν όπλα στη Σαουδική Αραβία η οποία τα χρησιμοποιεί για να πολεμήσει στη Συρία. Τότε θα μειωθούν οι μεταναστευτικές ροές και τότε μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Τότε θα υπάρξουν κάποιες λύσεις, αλλά δυστυχώς έχουμε να κάνουμε με ένα διεστραμμένο κύκλο εδώ ε, τα οικονομικά συμφέροντα και η προστασία των συμφερόντων πολιευτικών είναι πολύ πιο σημαντικά από την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Πρέπει βέβαια να δείξουμε και λίγο ρε παιδί μου μια ρίδα ανθρωπιάς. Οπότε γεια σου Σέγγεν και έτσι θα φροντίσουμε τον ευρικό λαό και τη δημόσια τάξη αλλά νομίζω ότι αυτό θα προκαλέσει βέβαια προβλήματα στην εσωτερική αγορά. Οπότε ας φτιάξουμε ένα καινούριο Σέγγεν, ένα μίνι Σέγγεν για το φρούριο της Βόρειας Ευρώπης. Δίνουμε και τρία δι στην Τουρκία. Ξέρουμε βέβαια ποιος παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός της Τουρκίας, αλλά μεταθέτουμε τις ευθύνες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απαντήσεις του κινήματος των πέντε αστέρων είναι εδώ και καιρό. Όχι στις βιομηχανικές και ενεργειακές πολιτικές όχι στην πολιτική του Δουβλίνου 2. Ας ξεκινήσουμε με τις αιτίε και μετά θα δούμε τις επιπτώσεις. Η κυρία Μάιερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, Κατακλείζεται η Ευρώπη από ετούντε άσυλο που αποτελούν κίνδυνο για την κοινωνία μα, την ελευθερία μα και την ειρήνη μα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει με κάθε κόστο να διατηρηθεί ε, στην Ευρώπη χωρί σύνορα, το οποίο είναι αρνητικό για όλου. Πρόκειται για έναν εφιάλτη για το 2016. Ε, έχουμε περάσει πλέον στην ελεύθερη κυκλοφορία τρομοκρατών, ετούντων άσυλο και καλάζνικοφ και θέλουν μάλιστα και δωρεάν ε, περίθαλψη, δωρεάν στέγαση και δωρεάν τροφή. Μιλήσατε για τη Σέγγεν και άλλε συνθήκε από την ευρωπαϊκή προϊστορία. Ενώ πρέπει να ασχολείστε περισσότερο με την κατάπτωση τη Ευρώπη. Ξυπνήστε. Έχει πτωχεύσει. Έχει ε, αποτύχει η Σέγγεν. Ακούστε τον λαό μας που πλέον ε, έχει ε, απαυδίσει με την ε, ανοιχτή Ευρώπη. Κλείστε τα Ολλανδικά σύνορα, προστατεύστε τους Ολλανδούς, προστατεύστε την ελευθερία μας και το μέλλον μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι αιτίες των μεταναστευτικών ροών είναι γνωστές έλλειψη οργάνωσης στον κόσμο με τη συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών σε χώρες όπως η Λιβύη, η Συρία, το Ιράκ. Και μετά η ρητορική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως ορισμένων πολιτικών δυνάμεων και ορισμένων χωρών μελών που ζητούν για ιδεολογικούς λόγους και για πολιτικούς λόγους ζητούν συνεχώς μετανάστες και η έκκληση της κυρίας Μέρκελ πέρασε, αλλά ε, ο κύριος Πιτέλα και η κυρία Χάρνους μας είπαν πολλά και ωραία πράγματα, συγκινητικά πράγματα. Βέβαια όταν γυρίσουν στις χώρες τους και δουν ξαφνικά τους παράνομους μετανάστες που χωρίς να το ξέρουν μπήκαν στα σπίτια τους, θα φωνάξουν την αστυνομία και θα βάλουν διπλές κλειδαριές, όπως επίσης θα κατεβάσουν και τα παντζούρια τους. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει τίποτα, μένει αδρανής. Βλέπουμε ότι σε επίπεδο ρητορική τουλάχιστον αυτοί που δεν θεωρούνται πολιτικοί πρόσφυγες και είναι η τεράστια πλειοψηφία των μεταναστών και το γνωρίζετε καλά οφείλουν να επιστρέψουν στην χώρα προέλευσής τους. Μα τι ωραία ιδέα, πού την πετύχατε. Εδώ στη Γαλλία, στη χώρα μου αποδείχθηκε από, μια, ε, ε, από το ελεγκτικό συνέδριο ότι το 95% αυτών των οποίων απερίπτεται η αίτηση για χορήγηση ασύλου παραμένουν στην χώρα με χιλιάδες τρόπους έφεσης, αμφισβήτησης, ανάκλησης ή όταν τους πηγαίνουμε στα βελγικά σύνορα για να φύγουν επανέρχονται την επόμενη ημέρα από τη χώρα από την οποία υποτίθεται απελάθησαν. Λοιπόν, η αρχή της μη επαναπρόθεσης είναι παράλογη για κάποιες χώρες. Ούτε το άρθρο της Σύμβασης της Γενέβης, ούτε το άρθρο 19 της χάρτας της Ευρωπαϊκής δεν αποκλείουν στο να μπορούμε να διώχνουμε αυτούς οι οποίοι έρχονται για αυστηρά οικονομικούς λόγους στην Ένωση. Ο κύριος Γκονσάλες Πόνς. Θα πω αυτά τα οποία έλεγα τον Δεκέμβριο, τον Νοέμβριο, τον Οκτώβριο Έχουμε μπει μέσα σε μία σύραγγα του χρόνου και δεν μπορούμε να βγούμε. Σήμερα υπάρχουν φυσικά περισσότερους νεκρούς μετανάστες από ό,τι είχαμε το Δεκέμβριο και το Δεκέμβριο περισσότερους από το ότι είχαμε τον προηγούμενο Οκτώβριο. Λοιπόν, ό,τι κάνουμε μέχρι τώρα έχουν αποτύχει. Οι νεκροί ο αριθμός τους αυξάνεται. Οι πολίτες αυτό το οποίο λέγουν είναι ότι το μόνο που ξέρουμε να κάνουμε και μάλιστα ούτε καν δεν λέμε καινούργια πράγματα. Επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα συνεχώς. Πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση να φέρουμε εις πέρας. πρέπει να ξεκινήσει και δεν ξέρουμε πώς η νέα υπηρεσία για τα σύνορα. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα δώσουμε τα χρήματα στην Τουρκία και χωρίς την Τουρκία δεν πρόκειται να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να έχουμε μια κοινή μεταναστευτική πολιτική καταργώντας τα σύνορα μένα ανάμεσα στις χώρες μας αλλά εξακολουθώντας να έχουμε 24 διαφορετικές πολιτικές μετανάστευσης. Δεν έχουμε ε, συμφωνήσει ακόμα ότι σε αυτούς οι οποίοι πρέπει να μοιραστούν τα δικαιώματά μας, πρέπει να μοιραστούν και τα καθήκοντά μας, τις αξίες μας, την ανοχή μας και την μεγάλη σημασία την οποία δίδουμε στην ισότητα των φύλων. Πολλά πράγματα μένει να γίνουν, πολλά πράγματα μένει να κάνουμε και το να περιμένουμε να μεγεθυνθούν οι συνέπειες του προβλήματος δεν βοηθά σε τίποτα. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις αιτίες. Δεν είναι αλήθεια ότι η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία δεν έχουν σύνορα, μα τα σύνορά τους είναι στην Ελλάδα. Η ελληνική αστυνομία φυλάσει τα σύνορα της Γερμανίας, στη συγκεκριμένη περίπτωση λέει ο μιλητής. Πρέπει λοιπόν να συντονιστούμε γιατί αν δεν γίνει αυτό τότε κάθε χώρα θα κλειστεί στα δικά της σύνορα. Λοιπόν, και δεν είναι ότι αυτοί που έρχονται και πνίγονται θέλουν ε, απλά ένα τρόπο καλύτερη ζωής, θέλουν να ξεφύγουν από τον θάνατο ε, και έχουν ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι χάσει τη ζωή τους αναζητώντας τη σωτηρία. Λοιπόν, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δημιουργεί προβλήματα στον εαυτό της με την πολιτική της της μετανάστευσης. Οι πολιτικοί μεταξύ τους ε, τσακώνονται αλλά δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Ή όμως θα το αντιμετωπίσουμε ή τότε θα ακολουθήσουμε δυστυχώς τις λαϊκίστικες πολιτικές. Του κυρίου Φροντσούλικα μπλε κάρτα. 30 δευτερόλεπτα κύριε Φροντσούλικα. Δεν νομίζετε ότι οι Ευρωπαίοι πολιτές περιμένουν να δουν από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να λαμβάνουν αποφάσεις, όχι μόνο να μιλούν σε ό,τι αφορά αυτή τη μεταναστική κρίση. Και δεν θεωρείτε ότι τα δικά μας θεσμικά όργανα επίσης θα πρέπει να εξετάσουν και το ζήτημα των αραβικών, των μουσουλμανικών χωρών, των χωρών του κόλπου, που επίσης θα πρέπει να υποδεχθούν μετανάστες, γιατί ανήκουν και στο δικό τους κόσμο. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι τα ευρωπαϊκά όργανα μπορούν να πάρουν αποφάσεις, αλλά δυστυχώς δεν τις εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη. Ε, νομίζω ότι δεν είναι επιλογή το να είναι κανείς ε, πρόσφυγας. Το θέμα είναι να μπορέσει κανείς να ξεπεράσει τις μικροπολιτικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω το έχει κατανοήσει. Madame Κυρία Φαγιόν, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όλο ένα και αυξανόμενο αριθμό Ευρωπαίων πολιτών φοβούνται τη μεταναστευτική κρίση. Έχουμε έω και 2.000 ετούντε άσυλο που εξέρχονται στην Ευρώπη κάθε ημέρα. Και τι θα γίνει την Άνοιξη που θα αυξηθούν μάλιστα οι ροές και όταν θα πρέπει να περάσουν από αυτά τα ασταθή Δυτικά Βαλκάνια και μετά Σλοβενία και το καθεξής. Από τα hot spots στην Ελλάδα μόνο ένα λειτουργεί. Οι μηχανισμοί μετεγκατάσταση και επαναπροώθηση δεν λειτουργούν ούτε το σχέδιο δράση με την Τουρκία. Ακόμα και η διάσκεψη τη ε, Γενέβη, ακόμα και αν ε, επιφέρει την ειρήνη, δεν περιμένουμε να υπάρχει ειρήνη από αύριο. Τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι δεν ξέρουμε καν ποια είναι η τύχη 10.000 ασυνόδευτων ανηλίκων. και μετά τα όσα έχουμε δει και στη Σουηδία, τι μπορεί να γίνει και στο μέλλον. Είναι τρομερέ οι προεκτάσει και απαιτούν άμεση ανάληψη δράση. Η Ευρώπη δεν έχει επιληφθεί επαρκώ τη μεταναστευτική κρίση. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα στατιστικά στοιχεία. 1,5 εκατομμύριο μετανάστε σε μια Ευρώπη 550 εκατομμυρίων. Είναι κάτι διαχειρίσιμο, αλλά κάποιο από τα ευρωπαϊκά όργανα πρέπει να αναλάβει την πολιτική ηγεσία. Όταν η Σλοβενία μπήκε στη Σέγγεν, εμεί ε, ε, είδαμε ένα νέο πρόσωπο τη Ευρώπη. Μια Ευρώπη ε, που μας υποδέχθηκε με τον πιο διαφανή τρόπο και τώρα κλείνει τα σύνορά της ε, με εθνικούς εγωισμούς. Ο κύριος Κέρκοπ για δύο λεπτά. Πρόεδρε. Ένα απλό μήνυμα. Έχω σε μια πολύ σύνθετη κατάσταση. Οι κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται και θα πρέπει να είναι και προτεραιότητα η υλοποίησή του. Ε, τα σημερινά συστήματα έχουν παραλύσει εξαιτία ε, μια έλλειψη βούληση και υιοθέτηση αποφάσεων σε ad hoc βάση. Ήρθε η ώρα λοιπόν να δείξουμε ότι έχουμε ένα σωστό σύστημα και πρέπει να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε τι αρχέ μα και μόνο έτσι θα αποκτήσουμε τον έλεγχο. Αν θέλουμε μαγικέ λύσει που θα πάρουν χρόνια να ελοποιηθούν, θα ξεφεύγει όλο και περισσότερο από τον έλεγχό μα κατάσταση. Πρέπει να παίρνουμε τελικά αποτυπώματα από του νεοαφιχθέντε. Αυτό δεν πρέπει να είναι ε, επιλογή, αλλά ε, να υπάρχει υποχρέωση για οποιονδήποτε θέλει να μείνει στην Ευρώπη, να τον υποδεχθούν οι χώρε. Εάν τα, τα μέλη ε, αποδεχθούν, πρέπει να αποδέχονται και την βοήθεια του Frontex. Θα πρέπει να επιστρέφονται αυτοί που δεν ε, ε, γίνονται δεκτοί ως πρόσφυγες. Ε, βλέπουμε ότι είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά επιστροφών. Τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να μεταθέτουν ε, το πρόβλημα και να κατανοούν ότι και η συμβολή του ε, είναι απαραίτητη. Το Δουβλίνο πρέπει να διατηρήσει τι βασικέ αρχέ και η μετεγκατάσταση θα πρέπει να είναι το δευτεροβάθμια διαδικασία, παρότι πρέπει να αναθεωρηθεί το Δουβλίνο. Εάν δεν, μπορούν δεν μπορεί μια χώρα να ελέγξει τα σύνορά τη και να εξασφαλίσει τι απαραίτητε συνθήκε διαβίωση, θα πρέπει να αναθεωρηθεί και η συμμετοχή στη Σέγγεν. Έχουμε τα περισσότερα μέσα που χρειαζόμαστε. Πρέπει τώρα να τα εφαρμόσουμε με θάρρος και αποφασιστικότητα. Ε, για τα σχόλια του κυρίου Βερχόφστατ ε, προηγουμένω. Κύριε Βερχόφστατ, ξέρετε ότι δεν πρέπει να λειτουργείτε υποκριτικά. Μπορείτε να καταδικάζετε μια άλλη πολιτική ομάδα και την ηγεσία τη σε σχέση με παρατηρήσει ενό μέλου ή τη συμπεριφορά του. Όμω δεν πρέπει να το κάνετε αυτό εάν δεν καταδικάζετε και την συμπεριφορά δικών σα μέλων, τη δική σα πολιτική ομάδα. Όταν το, ο αντιπρόεδρο του ΕΛΚ δεν ήταν. Ε, ε, ε, ε αποτέλεσε αντικείμενο εξυβρίσεω μια πρόσφατη πρόσφατη συνάντηση. Πρώτα να κοιτάξετε τα του οίκου σα, κύριε Βερχόφστατ, πριν ε, πιάσετε στο στόμα σα του υπόλοιπου. Ο κύριο Λάμσδορφ για 1,5 λεπτό. Ah, <laughs> Κυρίε και κύριοι, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια μεγάλη κρίση, η οποία απαιτεί μεγάλες προσπάθειες. Ε, θέλουν λύσεις οι πολίτες, θέλουν ένα τέλος ε, από την ε, αποστροφή της ευθύνης ε, από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό το παρουσίασε ο πρόεδρος του Συμβουλίου ότι ελήφθησαν αποφάσεις ε, και τώρα το θέμα είναι να τις, εφαρμόσουμε. Και μία απόφαση είναι η εξή. Το Συμβουλίο αποφάσισε να διοργανώσει κάποιες συναντήσεις των αρμόδιων οργάνων για να ελέγξει προσεκτικά το ότι αναφέρεται σε κάποια έγγραφα τα οποία υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, με αυτό το ρυθμό κυρίες και κύριοι, με αυτή τη στάση, δεν πρόκειται να την ξεπεράσουμε την κρίση. Έχει έρθει πια το πλήρωμα του χρόνου να αντιμετωπίσουν τι ευθύνε του στα κρατη και θα πρέπει να ηγηθεί το Συμβούλιο. Και αυτό που βλέπουμε στα κρατη είναι σκάνδαλο. Ο συνάδελφο του Καδημούλη, έχει δίκιο έχουν ε, ε, γίνει κατανομή λίγων μόνο μεταναστών. Αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία στην Ελλάδα να μην καταβάλει μεγάλες προσπάθειες. Έχουμε μια, ένα μεγάλο συνασπισμό στην ε, Γερμανία και απογοητεύει τους πολίτες. Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι η κατάσταση. Επικρατεί φόβος μεταξύ των πολιτών και αυτός ο φόβος είναι κακός και θα πρέπει να βρεθούν λύσεις για αυτό το φόβο, για αυτή την κρίση. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια κοινή ακτοφυλακή, κοινή συνοριοφυλακή, μια ε, γρήγορη ε, ομάδα για παρέμβαση βάσει του άρθρου 76, μια κοινή μεταναστευτική πολιτική, χρηματοδότηση για το World Food Program. Χρειαζόμαστε ε, δραστηριότητε τη κυρία Μογκερίνη. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε, μα τα κάνουμε επιτέλου. Ξεπεράσατε αυτό το χρόνο ομιλία σα και μιλάτε και πάρα πολύ γρήγορα, κύριε Λαμπστόρφ, λέει η πρόεδρο. Η κυρία Ένστη για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Η Ελλάδα πρέπει να προστατεύσει καλύτερα τα εξωτερικά τη σύνορα. Πέρα από το γεγονό ότι έχει 13.666 χιλιόμετρα ακτογραμμή η ε, Ελλάδα, σας ρωτώ, τι θέλετε και τι εννοείτε, τι φαντάζεστε ότι μπορεί και πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Στην Ελλάδα αναρωτιέμαι οι Έλληνες ε, οι οποίοι τώρα σώζουν χιλιάδες ε, μετανάστες χωρίς αλληλεγγύη από τα κράτη-μέρη. Τι θα τους κάνουν, τους στείλουν πάλι στις βάρκες τους, τους μετανάστες. Τι φαντάζεστε, να τους βγάλει εισιτήριο για το χαλέπι η Ελλάδα πάλι. Τι, τι, να κάνει. Τι καταλαβαίνετε με τον όρο ασφάλεια των συνόρων. Με φοβίζει εμένα αυτό. Με φοβίζει γιατί αυτό θα, θα στείλει σε θάνατο και άλλους ανθρώπους. Και ουσιαστικά αυτά είναι λόγια των ε, λαϊκιστών, των ε, ακροδεξιών, που θέλουν να επαναεισαγάγουν πρακτικές όπως αυτές των περιβολισμών. Και αυτά είναι εγκληματικά. Θα ήθελα να το τονίσω αυτό κυρίες και κύριοι. Θα πρέπει να πούμε ένα πράγμα ξεκάθαρο ότι η άνοδος της δεξιάς και η μαζική μετανάστευση έχουν τις αιτίες τους. Ε, γιατί το γεγονός ότι εμείς εδώ στον Κοινοβουλίο δεν λέμε και δεν καταδικάζουμε ξεκάθαρα τη βία κατά των μεταναστών. Δεν μιλάμε και να μην ξεχνάμε και να μην ανεχόμαστε τη βία και τα βασανιστήρια των μεταναστών. Και το γεγονός ότι έχουμε προσφυγικούς καταβλισμούς στη Γερμανία Μιλάει παράλληλα η Πρόεδρος και κόβει την ομιλητρία. Δυστυχώς. Ευχαριστώ κυρία Σαργεντίνη για ένα λεπτό. Κυρία Έρνστ, έχει τελειώσει ο χρόνο ομιλία σα Πολύ λυπάμαι, αλλά πρέπει να σεβαστούμε το χρόνο ομιλία. Η κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, πρόκειται για μια ευκαιρία διαλέφκανση ε, των ε, λόγων του πρώτου αντιπροέδρου του τη επιτροπή του κ. Τίμερμαντ, ο οποίο είπε σε μια συνέντευξη την προηγούμενη εβδομάδα ότι 60% των μενεστών που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πρόσφυγε, αλλά οικονομικοί μετανάστε. Εν τω μεταξύ, η Eurostat, η Frontex, ο ION, ο UNAGR, η EASO, όλοι έχουν διαψεύσει αυτή τη δήλωση. Ο κύριος Τίμερμανς όμως έχει σιωπήσει την τελευταία εβδομάδα και εντωμεταξύ τον παραθέτουν να εκμεταλλεύονται τα λόγια του αυτά και αυτό συνεχίζει να επηρεάζει και την υποδοχή των μεταναστών στη χώρα μου και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα λοιπόν είναι η στιγμή της αλήθειας και της διαλεύκανσης. Τα λόγια του κ. Τίμερμανς αποτελούν άραγε την επίσημη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ναι ή όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νουτάλ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Όλοι συμφωνούμε, πιστεύω, ότι η μεταναστευτική κρίση πέρυσι ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλη της την ιστορία. Μάλιστα, θα μπορούσα να πω ότι έχει θέσει την ίδια την ύπαρξη ολόκληρου του οικοδομήματος σε, κίνδυνο. Και θεωρώ εξωπραγματικό ότι οι ίδιες οι ενέργειές σας προκάλεσαν όλο το πρόβλημα από την αρχή. Όταν ε, κάλεσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες οποιονδήποτε έχει ένα διαβατήριο να έρθει ε, στην Ευρώπη ήταν σαφέ τι θα γινόταν. Ότι θα προσπαθούσαν οι άνθρωποι με κάθε κόστο, ε, θα θαλασσοπνίγονταν για να έρθουν στην Ευρώπη. Τα, τα κράτη-μέλη θα έρθουν το ένα αντιμέτωπα με το άλλο, ότι θα καταρρεύσει η συνθήκη Σέγγεν και θα είναι μια χρυσή ευκαιρία για τους ε, Ισλαμιστέ φονταμεταλλιστέ να φέρουν το μακελιό στην Ήπειρό μα. Ήταν επίση προφανέ ότι θα πρέπει να υπάρξουν και κολοτούμπε εντό εισαγωγικών, όπω είδαμε του περισμένου μήνε, από την γερμανική και σουηδική κυβέρνηση. Τώρα έχουμε μια μεγα... ακόμα μεγαλύτερη κρίση. Οι αριθμοί δεν θα μειωθούν σε σχέση με πέρσι. Το καλοκαίρι βλέπουμε ότι οι μεταναστευτικέ ροέ από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική σίγουρα θα φτάσουν, ε, ε, θα έρθουν σε επιβλικέ διαστάσει. Και τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίλυση του προβλήματο, τα ίδια και τα ίδια περισσότερε υπαναχωρήσει, περισσότερη Ευρωπαϊκή Ένωση, περισσότερα χρήματα και περισσότερα βάσανα όχι μόνο για του μετανάστε, αλλά και για πολλού από του πολίτε μα. Πρέπει να θέσουμε ένα τέλο σε αυτόν τον παραλογισμό, κυρίε και κύριοι. Και η απάντηση δεν είναι να κάνουμε τα ίδια ασφάλματα ξανά και ξανά. Είναι να αποκαταστήσουμε τον σύνορο, τον, ε, τον έλεγχο των συνόρων, όπω έχουν κάνει οι Αυστραλοί τα τελευταία πέντε χρόνια. Ωστόσο, για να πετύχει το Ηνωμένο Βασίλειο αυτόν τον στόχο, θα πρέπει να ψηφίσουμε να αποχωρήσουμε από τον οργανισμό στο επερχόμενο δημοψήφισμα. Ευχαριστώ. Κύριε Νουτάλ, δέχεστε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Ντελανό. Παρακαλώ. Το μικρόφωνο σας. Πιστεύετε ότι οι μετανάστες περίμεναν την άδεια της κυρίας Μέρκελ για να φύγουν από μια χώρα όπου πλέον δεν μπορούσαν να επιβιώσουν. Ε, Υφίσταν συνεχή τρομοκρατία ε, και τον φόβο της, ε, των βομβών. Περιμέναν λοιπόν την άδεια της κυρίας Μέρκελ. Μάλιστα, ναι. Θεωρώ ότι όταν η Άγγελα Μέρκελ είπε ότι η Γερμανία θα υποδεχθεί οποιονδήποτε μπορεί να αποδείξει ότι είναι Σύριος, ένα τεράστιο αριθμό ανθρώπων ήρθαν. Γι' αυτό και πολλούνται τώρα πλαστά σε διαβατήρια ε, στην Τουρκία στο διαδίκτυο για 300 400 ευρώ. Και βλέπουμε ότι και πολλοί σύρι, υποτιθέμενοι Σύριοι πρόσφυγες έχουν πλαστά διαβατήρια. Και έτσι θέτουμε τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών ε, σε κίνδυνο. Και βλέπετε τι συνέβη στην κολονία προσφάτως. Είναι μια πρώτη γεύση του τι θα συμβεί στην Ήπειρό μας. Παρακαλώ, Φοντάνα, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ και δύο χρόνια το πρόβλημα αυτό ταλαιπωρεί την Ευρώπη. Διαρωτώ με αν υπάρχει πολιτική βούληση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των χωρών να το αντιμετωπίσουν. Από αυτό το οποίο εγώ καταλαβαίνω και μετά και από τη σημερινή συζήτηση Υπάρχουν δύο εδώ απόψεις. Από τη μία είναι αυτή που είναι ιδεολόγη και λέει ότι όλοι οι πρόσφυγες είναι καλοί άνθρωποι, έχουν ανάγκες, ας τους υποδεχθούμε όλους, ας τους δώσουμε και τα σπίτια μας. 22 πρόσφυγες την προηγούμενη εβδομάδα στην πόλη μου τους βάλαμε σε ένα ξενοδοχείο και τους κάναμε και μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης, κάτι το οποίο οι Ιταλοί δεν έχουν την ευκαιρία να κάνουν. Λοιπόν, ε, πρέπει να προσέχουμε βέβαια γιατί ε, αυτοί που διαφωνούν τους κατηγορείται για λαϊκιστές, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω τι συμφέρον υπάρχει όταν εξαφανίζονται 10.000 ανήλικοι, όταν τα πρόσωπα αυτά προφανώς τα κατέχει η μαφία, τα εκμεταλλεύεται η μαφία όταν συνελήφθησαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Ιταλία πρόσφυγες που ζητούν άσυλο για ε, λαθρεμπορία ναρκωτικών, όταν γίνονται αυτά τα οποία γίνονται στην κολονία. Τότε μήπως δεν έχουμε συμφέρον να τους βάλουμε όλους αυτούς. Μήπως αν τους αφήνουμε θέλουμε να δημιουργηθεί ένα χάος. Ίσως να υπάρχουν συμφέροντα για τη δημιουργία αυτού του χάους. Κόρμιν Μίκη για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά την αίτηση για άσυλο στην πρώτη χώρα άφηξης, εκεί πλέον η ζωή του μετανάστε δεν απειλείται και γι' αυτό προχωρούν. Γιατί αυτή η ξανθιά από το Βερολίνο τους υποσχέθηκε να τους υποδεχτεί. Ίσως να έχει και όμως ο κ. Γκόλνης. Μπορεί κάποιος πραγματικά να θέλει να διώξει τους Ευρωπαίους από την Ευρώπη και να έλθουν άλλοι στη θέση τους. Όταν ε, πέθανε ο Μάο το σύστημα κατανομής ε, ρίζιου σταμάτησε και το είχε αυτό αποτέλεσμα για τον κινέζικο πληθυσμό και το ίδιο έγινε με τα δακτυλικά αποτυπώματα και τα παιδιά των μεταναστών. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες παιδιά. Η κυρία Χολμαϊρ. Έχετε το λόγο. Μάλιστα. Να, αγαπητοί συνάδελφοι, να καλωσορίσω και τον Επίτροπο και την Προεδρία του Συμβουλίου. Καταρχάς, κυρία Έρνστ, θα ρωτήσετε τι θα πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Μα επιτέλους να συνεργαστεί απόλυτα, επιτέλους να συνεργαστεί με την Frontex, με την ΕΑΣΟ, επιτέλους να δείξει απόλυτη ε, διαφάνεια για την καταχώρηση και επιτέλους να δείξει την προθυμία να καταρτήσει μια πολιτική ε, μαζί με τα κράτη-μέλη και να μην αντιμετωπίζει τον εαυτό της ως ε, κράτος διαμετακόμισης και διέλευσης πλήρη συνεργασία. Αυτό λοιπόν περιμένουμε από όλους τους από όλα τα κράτη-μέλη και να μην αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως τη χώρα που έχει τη μόνη ευθύνη. Αυτό θα ήταν κοινή στάση και συνεργασία ευρωπαϊκή. Αλλά πέραν από αυτό, περιμένω να επιδείξουμε και την ε, προθυμία να σκεφτούμε και λίγο πιο ευρέω. Για παράδειγμα, να δημιουργήσουμε ζώνε προστασία, νέου καταβλισμού εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί μόνο αν και άλλε χώρε στην Αφρική ή στην Εγγύη Ανατολή δείξουν την προθυμία να συμμετάσχουν, μόνο τότε θα μπορέσουμε ενδεχομένω να επιλύσουμε κάτι παραπάνω από το πρόβλημα κάποιων λίγων που έρχονται μέσω τη Μεσογείου σε εμά. Αν αναπτύξουμε ένα πιο ευρύ σχέδιο το οποίο θα οδηγήσει στην ε, μετακίνηση λιγότερων μεταναστών, θα πρέπει να εργαστούμε και στην Αφρικανική Ήπειρο και όχι μόνο, αποκλειστικά και μόνο, στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Χολμαϊρ, λέει πρόεδρος, έχετε δύο μπλε κάρτες, ε, Γκραπίνη και Έρνστ. Η κυρία Γκραπίνη και μετά η κυρία Έρνστ. Η κυρία Γκραπίνη λοιπόν πρώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε. Αγαπητέ συνάδελφε, ακούσαμε τι είπαν οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου και τη Επιτροπή, αλλά υπάρχουν μετανάστε που δεν έχουν δικαίωμα ασύλου. Δεν πιστεύετε ότι μετά από τόσο καιρό θα πρέπει να υπάρχουν σαφεί κανόνε για να εφαρμόσονται μάλιστα με ενιαίο τρόπο από τι κυβερνήσει, για να ξέρουμε ακριβώ τι πρέπει να κάνουμε με του ανθρώπου αυτού που έρχονται. Ασφαλώ, επειδή το χρειάζονται. Κάποιοι επειδή ξεφεύγουν από τη φτώχεια, κάποιοι από τον πόλεμο. Κυρία Χολμάιρε, έχετε το λόγο. Υπάρχουν σαφείς διαφορές. Καταρχάς, αυτοί που είναι μετανάστες, ε, οι οποίοι για ανθρωπιστικούς λόγους ε, πρέπει να μείνουν γιατί φοβούνται για την επιβίωσή τους και είναι και αυτοί οι οποίοι αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον, η μετανάσταση οικονομική. οι οποίοι ασφαλώς θα πρέπει να τηρήσουν και τους νόμους που ισχύουν σε κάθε χώρα και δεν θα πρέπει να επικάλυπτουν το ανθρωπιστικό δίκαιο. Αυτό σημαίνει ότι οι οικονομικοί μετανάστες θα πρέπει να επιστρέφονται, γιατί δεν μπορούν βάσει της αίτηση ασύλου να εισέλθουν, αλλά θα πρέπει να τηρούν τον νόμο της κάθε χώρας. Η κυρία Έρνστ έχει το λόγο για δεύτερη μπλε κάρτα. Μάλιστα παραδουλεύει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Χολμάιερ, για την Ελλάδα είπατε εξαιρετικά πράγματα. Εγώ λοιπόν έχω να ρωτήσω το εξή. Κατά πόσο συμφωνείτε μαζί μου ότι ενδεχομένω και τα κράτη-μέλη και μάλιστα με σημαντικό τρόπο θα πρέπει να συμβάλλουν για την υποστήριξη της Ελλάδα. Να πάρουν πιο πολλούς προσφυγε, για παράδειγμα. Εκεί που έχετε ενστάσεις, για πείτε μου. σε κάποιες ε, περιπτώσεις, ε, κυρία συνάδελφε, έν, θα ήταν καλό να με ακούτε κιόλα. Αυτό απάντησα στην ομιλία μου. Είπα ότι αφενός ε, αναμένω πλήρη συνεργασία από την Ελλάδα και σε θέματα καταχώρησης, σε θέματα δίωξης των εμπόρων ανθρώπων, αλλά και από την άλλη σας είπα ότι αναμένω και από τα κράτη-μέλη αν η Ελλάδα δείξει αυτή την προθυμία να δείξουν σοβαρές διαθέσεις, να ξέρει η Ελλάδα ότι έχουν σοβαρές προθέσεις και ότι θα κάνουν τα πάντα για την ανακατανομή των ε, ανθρώπων. Υπάρχει συνεργασία, αλλά μόνο από κοινού. I'm sorry, there is only one... Συγγνώμη, έχουμε μόνο μία δυνατότητα υποβολής ερωτήματος. Για τον κύριο... Ο κύριος Μποστινάρου για 1,5 λεπτό. declarații Το μόνο το οποίο εγώ θα ήθελα να, μην ακούω για τον χώρο του Σέγγεν είναι τέτοιου είδους δηλώσεις που ακούμε τελευταία. Νομίζω ότι διατρέχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα το Σέγγεν. Η Ρουμανία ξέρετε ότι έχει κάθε λόγο να προσβλέπει στην ένταξή της στη συμφωνία του Σέγγεν. Εμείς θέλουμε λοιπόν να εγκαταλείψουμε τις εθνικιστικές ρητορικέ οι οποίες δεν οδηγούν σε καμία λύση. Θέλουμε με συγκεκριμένο τρόπο να δράσουμε από κοινού και να ξεπεράσουμε το σύστημα του Δουβλίνου το οποίο είναι ιδιαίτερος ξεπερασμένο. Πρέπει επίσης να προστατεύσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα μέσω ακριβώς και της δύναμης άμεσης ε, ταχείας παρέμβασης όπως είχε πει το Συμβούλιο πρόσφατα και το οποίο ακόμα δεν έχει κάνει βήματα σαν απόφαση. Και έχουμε επίσης και στην Τουρκία ένα σημαντικό εταίρο για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Απαιτείται λοιπόν να εφαρμοστεί το πρόγραμμα δράσης με την Τουρκία. Πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως και από την Τουρκία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αντιστηρίξουμε αυτές τις αποφάσεις με συγκεκριμένα μέτρα έτσι θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα και να ελέγξουμε τις μεταναστευτικές ροές. Ε, Ο κύριος Κόλμελ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, βλέπουμε εδώ στη θέματα μεταναστευτικής κρίσης ε, όχι μία νομική κρίση, αλλά μία πολιτική κρίση. Υπάρχει το δίκαιο, υπάρχει νομοθεσία, πρέπει να εφαρμοστεί. Όμως η γερμανική κυβέρνηση με την κουλτούρα της υποδοχής έχει θέσει σε εφαρμογή μία τάση η οποία πιέζει τα κρατημέλη. Τώρα έχει έρθει η ώρα της αλήθειας. Τώρα θα πρέπει να αποδείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι σε θέση να αντιδράσει και να δράσει. Αλλά πριν από αυτό θα πρέπει να κάνουμε μια ειλικρινή ανάλυση. Μιλάμε για βοήθεια. Η βοήθεια είναι εθελοντική και θα πρέπει να είναι ε, να παρέχεται σε βάθος χρόνους. Δεν μπορούμε να δίνουμε και να περιμένουμε από κάποιον να, δίνει, να δίνουμε βοήθεια ε, μέχρι να γίνεται, να εξαρτάται από τη βοήθεια. Θα πρέπει λοιπόν να διαπιστώσουμε ποιες είναι οι δυνατότητες ε, πρόσληψης ανθρώπων, αποδοχής ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν τι μπορεί να κάνει κάθε χώρα και θα πρέπει να ερευνήσουμε το τι θέλει και τι προτίθεται να κάνει κάθε χώρα. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστό ότι μπορεί οι πολιτικοί ηγέτες από μακριά να επιβάλλουν πράγματα στους λαούς. Δεν πρόκειται να πετύχει αυτό. Και ούτε είναι δυνατόν η μεταναστευτική πολιτική να καταστεί απάνθρωπη. Και ένα κόμμα, ένας ε, ηγέτης ε, που λέει να πυροβολούνται οι πρόσφυγες, αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να τους πολεμήσουμε από κοινού. Γιατί τα κόμματα αυτά δεν μπορεί να έχουν πολλά επιχειρήματα. Μπλε κάρτα λοιπόν. Από την κυρία Γιακοντσάρη για τον κύριο Κολυμέλ την αποδέχεστε. Η κυρία Γιακοντσάρη. Πρόεδρε. Είπατε ότι οι πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι φύγονται από την κατάσταση. Προφανώς οι πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την πραγματικότητα της κατάστασης. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η κοινωνία των πολιτών έχει αντιδράσει. Ο Ερυθρός Σταυρός, σαν παράδειγμα, άλλες οργανώσεις και ο τρόπος που ανταποκρίθηκε η κοινωνία των πολιτών λοιπόν συμμετέχει στην προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος. Δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε το αντίθετο. Δυστυχώς οι αποφάσεις που λαμβάνονται στην Ένωση δεν εφαρμόζονται. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ συνάδελφε για την ερώτηση αυτή. όντω. είναι απόλυτα θετικό το γεγονός ότι πάρα πολλά κράτη-μέλη και οι πολίτες τους ε, εργάζονται και δεσμεύονται. Αλλά αυτό που είναι καθοριστικό είναι ότι θα πρέπει ο πολίτης να συμμετάσχει σε αυτό το βασικό ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί. Πόσους ανθρώπους θέλουμε να υποδεχτούμε και μπορούμε να υποδεχτούμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι καθοριστικό το ερώτημα αυτό και πρέπει να τεθεί προς τους πολίτες. Η κυρία Βίξτρομ, για λεπτό. Ευχαριστώ, πριν από μερικές ε, ημέρες ε, υπήρξε ε, ένα όχλος που επιτέθηκε σε πρόσφυγες στη Στοχόλμη. Ταυτόχρονα 39 παιδιά έχασαν τη ζωή τους, βελαμενόμενων και παιδιών, στα σκοτεινά κύματα της Μεσογείου. Τα όσα συμβαίνουν τελευταία στην Ευρώπη είναι τρομακτικά και έχουν προκληθεί από μία δυσεπίλητη ε, μεταναστευτική κρίση και δεν έχει επιληθεί γιατί ορισμένες χώρες έχουν αναλάβει μεγάλο μερίδιο των ευθυνών ενώ άλλες καθόλου. Μόνο από κοινού όμως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση αυτή. Μόνο μαζί μπορούμε να ανακτήσουμε τον ε, έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και πρέπει ε, να μεριμνήσουμε για τον κατάλληλο επιμερισμό και δίκαιο επιμερισμό των ευθυνών. Δεν μπορούμε απλώς να κλείσουμε τα σύνορα, να μην δεχθούμε κανέναν, να επιτρέψουμε στο μίσος να νικήσει. Ούτε να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια, εντελώς αδρανείς, περιμένοντας από κάποιον άλλον να αναλάβει την ευθύνη. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι έχει έρθει η ώρα να τα συνειδητοποιήσουμε όλα αυτά. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις ε, στην ιστορία της, αλλά και στο παρελθόν τα τα έχουμε περάσει όλα αυτά. Οι γονεί μα και οι παππούδε μα κατάφεραν να συνενώσουν την Ευρώπη μετά από δύο αιματηρού πολέμου. Έχουμε την ευθύνη να διατηρήσουμε αυτό το οικοδόμημα και κανένα δεν μπορεί να ε, μεταθέσει αυτή την ευθύνη. Παρακαλώ, έχετε μπλε κάρτα. Ναι, βεβαίω, Πρόεδρε, με τα χαρά λάβω οποιοδήποτε ερώτημα, οποιοδήποτε συνάδελφο. Παρακαλώ. Μπεύσκι. στην Πολωνία σεβόμαστε την απόφαση ε, της Σουηδίας. Τονίζω και πάλι ότι δεχόμαστε και σεβόμαστε την ευθύνη, συγγνώμη, την απόφαση ε, και την όλη νοοτροπία της φιλοξενίας ε, που ακολουθήσατε, αλλά και την επίπονη αυτή απόφαση να κλείσετε τα σύνορα και να επαναφέρετε τους ελέγχου. Όμως αυτή η απόφαση ελήφθη από τον Σουηδικό λαό. Μπορείτε εσείς να δεχθείτε μια αντίστοιχη ε, απόφαση της Πολωνίας ή της Τσεχίας σε αντίστοιχο θέμα. Ναι, είναι ευσταθεί το ερώτημά σας και εγώ δέχομαι να, να αναλάβω την ευθύνη για αντίστοιχε αποφάσεις. Τα Σουηδικά σύνορα είναι ίδια με αυτά της Ελλάδας ε, στη Μεσόγειο. Μαζί πρέπει να διασφαλίσουμε ε, την τήρησή τους. Όλοι πρέπει να θυμόμαστε και τις επιμέρους ιστορίες μας, την σύγχρονη ιστορία μας, στην Ουγγαρία, στην Τσεχοσλοβακία, όπου πολλοί κόσμος αναγκάστηκε να διαφύγει και τους υποδέχτηκαν. Στην Πολωνία, για παράδειγμα, έχετε υποδεχθεί πολλούς Ουκρανούς και το αναγνωρίζουμε. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να υποδεχθούμε και όσους ε, προσπαθούν να ξεφύγουν από τους πολέμους ε, στη Συρία, ε, από την Ερυθρέα και, και οπουδήποτε αλλού απειλείται η ανθρώπινη ζωή. Κυρία Μπιόρκη, 1,5 λεπτό. Κυρίες και κύριοι, η βία κατά των ε, μη λευκών, των μεταναστών και των προσφύγων συνεχώς αυξάνεται και στη Βουλγαρία και σε πολλές άλλες χώρες. Πολλές γειτονικές μας χώρες, πολλοί γείτονές μας μάλλον φοβούνται να βγουν στο δρόμο. Κοιτάζουν δεξιά και αριστερά, δεν παίρνουν καν τα παιδιά τους μαζί. Έτσι έχουν τα πράγματα σήμερα. Ξέρουμε ότι και οι νοναζοί είναι σε θέση ε, να διαπράξουν βιοπραγίες. Όμως εμείς τι τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε, τι είδους πολιτικές είμαστε διατεθειμένοι να υιοθετήσουμε. Κάτι το οποίο νομοποιεί την γνώμη του άκρος πολλωμένου κόσμου. Η Δανία υιοθετεί τρομερούς νόμους ε, που καταλυστεύει τους ε, πρόσφυγες. Η Σουηδία κλείνει τα σύνορα. Εμείς ε, συμβάλλουμε σε όλο αυτό. Και εσείς ανοίγεται το δρόμο για όλα αυτά. Και βλέπουμε ποιες είναι οι συνέπειες στην πράξη. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που θα σώζουν ζωές στη Μεσόγειο, που θα υποδέχονται πρόσφυγες. Χρειαζόμαστε έναν συνασπισμό ευρωπαϊκών κρατών φιλικές προς τους πρόσφυγες που θα συνεργάζονται από κοινού για την υποδοχή των προσφύγων. Χρειαζόμαστε μια νέα εξωτερική πολιτική, όχι μια νέα μεταναστευτική πολιτική που είναι απλώς οργισμένη με την Ελλάδα που δεν σταματά τους πρόσφυγες. Χρειαζόμαστε μια νέα συνολική πολιτική. Δέχεστε μπλε κάρτα από τον κύριο Γιούρεκ. Λυπάμαι. Ε, προχωράμε Λαμπέρ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ο μιλός στα πλαίσια και της διάσκεψης για τους δωρητές ε, για το Συριακό που διεξάγεται αυτή την εβδομάδα. Έχει καλυφθεί ε, κατά 60% η απόφαση που είχε ληφθεί στο παρελθόν και αυτό δημιουργεί προβλήματα και σε σχέση με τις ποσότητες των τροφίμων που είναι διαθέσιμες στο εσωτερικό της χώρας αλλά κυρίως και στις χώρες που περιβάλλουν την Συρία. Μόνο το 50% μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο από τα παιδιά των προσφύγων και γι' αυτό θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να συνεισφέρουν επαρκώς έτσι ώστε να υποστηρίξουν την τεράστια δουλειά των Ηνωμένων Εθνών η τεκμηρίωση όταν υπάρχει, όταν έχουν ε, οι πρόσφυγες κάποια χαρτιά έγκυρα μαζί τους, αυτό δεν δημιουργεί πολλά προβλήματα, αλλιώς όμως πάλι δημιουργούνται προβλήματα ακόμα και για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Πρέπει να επιληθεί το πρόβλημα ακριβώς του απάτριδος αυτού ο οποίος δεν έχει τα απαιτούμενα έγγραφα γιατί δεν μπορεί να τα έχει. Λούνγκρεν ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Παρά τα τόσο ωραία λόγια τα οποία ακούμε τελευταία μέσα στην Ολομέλεια θα πρέπει να μην απαραγνωρίζουμε την πραγματικότητα. Το πρόβλημα το οποίο έχουμε μπροστά μας είναι το πρόβλημα κυρίως των ανηλίκων, ιδιαίτερα των ασυνόδευτων ανηλίκων, που έρχονται σε καθημερινή βάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από ό,τι διαβάζουμε στα μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες μέρες εξαφανίζονται. Τα παιδιά αυτά ε, υφίστανται πιέσεις, υφίστανται βία, ενοχλήσεις, bullying ε, σε καθημερινή βάση από ε, άλλους νέους οι οποίοι παίζουν ένα συγκεκριμένο ρόλο. Εμείς τι του προσφέρουμε σε αυτά τα παιδιά, δεν έχουμε την δυνατότητα να διαχειριστούμε αυτή τη μαζική άφηξη των μεταναστών και παιδιών και ενηλίκων εδώ και ένα χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε για μια ακόμη φορά. Ο κύριος Λεμπρετό, ένα λεπτό. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Βοήθειας στους πρόσφυγες στην Τουρκία είναι μια κοροϊδία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει τρία δις έτσι ώστε να έχει μια ελπίδα να παραμείνουν τα δύο εκατομμύρια προσφύγων εκεί. Η Τουρκία δεν θα σεβαστεί αυτή τη συμφωνία. Είχε έρθει πριν λίγα χρόνια εδώ στο Στρασβούργο ο κύριος Ερντογάν, έκανε κριτική στην Ευρώπη και ζήτησε από τους Τούρκους της Γαλλίας να μην ενσωματωθούν. Ε, ο Ερντογάν αφήνει τους Σύρους πρόσφυγες να φύγουν επίτηδες προς την Ευρώπη. Χαίρεται για αυτό το οποίο συμβαίνει σε μας, τροφοδοτεί τα μεταναστευτικά ρεύματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ασθενής, είναι μια γραφειοκρατία δεν έχει βάση, δεν έχει στήριξη και θα χάσει αυτά τα τρία δις χωρίς να κερδίσει απολύτως τίποτα. Πρέπει να καταργηθεί η συμφωνία του Σέγγεν. Κάθε χώρα θα πρέπει να μπορεί να ελέγξει τα σύνορά της για να εμποδίσει τα ρεύματα αυτά και να διαπραγματευτεί με ισότιμο τρόπο με την Τουρκία. Στη δική μου χώρα επιβεβαιώνω ότι η Γαλλία θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της καλύτερα όταν βγει από τον Σέγγεν και κυρίως όταν βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παπαδάκης, για ένα λεπτό. η συζήτηση για τη σέγγεν και την ελλάδα αποτελεί μοχλό της ευρωπαϊκής ένωσης για πιο αποφασιστική εφαρμογή μέτρων καταστολής από την κυβέρνηση συριζα ανέλ με ξεδιάλεγμα των αναγκαίων για τα μονοπόλια προσφύγων δεν αποφασίζετε να επιστρέφουν όπως λέτε τους απελάβνετε πίσω στην κόλαση των πολέμων που η ίδια η ευρωπαϊκή ένωση και οι σύμμαχοί της δημιούργησαν και οξύνουν. τα ευρωπαϊκά σας σύνορα σημαίνουν γκριζάρισμα συνόρων στο αιγαίο τα τείχη ορθώνονται με τη σέγγεν σε ισχύ και έτσι φουντώνουν τα κυκλώματα διακινητών ενώ κατάσχονται οι τελευταίες οικονομίες των προσφύγων αποθρασύνοντας τις φασιστικές ορδές η σέγγεν δεν καταργεί τους ελέγχους αλλά τους επεκτείνει ηλεκτρονικά με βιομετρικά στοιχεία και φακέλωμα. είναι η εφαρμογή των διατάξεων 19 και 26 της σέγγεν που επιβάλλει συνοριακούς ελέγχους με τον ορατό κίνδυνο να εγκλωβιστούν μαζικά χιλιάδες απελπισμένοι πρόσφυγες στην ελλάδα. είναι άμεση ανάγκη απευθείας μεταφορά των προσφύγων στις χώρες τελικού προορισμού τους και οι λαοί να εντείνουν την πάλη τους για ένα κόσμο χωρί εκμετάλλευση υπεριαλιστικούς πολέμους και προσφυγιά. Ευχαριστώ κύριε Μαρινέσκου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Τα εξωτερικά σύνορα θα πρέπει να προστατεύονται και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ανταποκρίνονται και στις ε, απαιτήσει του Σόγκαν. και όποιος έχει προβλήματα θα πρέπει να υποστηρίζεται από τις ευρωπαϊκές ε, οντότητες από τη Frontex για παράδειγμα. Ελπίζω πολύ σύντομα να υπάρξει Ευρωπαϊκό Σώμα Συνοριοφυλάκων και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτήσει γρήγορα τα κοινά πρότυπα για την φύλαξη των συνόρων, όπω απαιτείται και από τη σχετική νομοθεσία. Ο χώρο Σέγγεν θα πρέπει να προστατεύεται και θα πρέπει να μειωθούν οι ροέ των μεταναστών. Θα πρέπει να σώσουμε τι ανθρώπινε ζωέ, αλλά δεν γίνεται αυτό βάζοντας αν θέλετε ένα τέρμα στη μετακίνηση των ανθρώπων από περιοχέ επικίνδυνε, θα πρέπει να υποστηρίξουμε και την Τουρκία και χρειαζόμαστε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στο πώ δαπανώνται τα κονδύλια ή τα χρήματα. Η πιο απλή λύση είναι αυτή των μεταφορών. Τα επόμενα χρόνια όλα τα χρήματα που δεν θα έχουν δαπανηθεί στο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο προβλέπεται ήδη 100, χρήση των μη κατανεμημένων ε, κονδυλίων για τέτοιες απρόβλεπτες καταστάσεις. Μάλιστα, έχετε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Μαυρίδη. Την αποτέχεστε. You have a Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, θέξατε στην αρχή αρχή ένα θέμα για τα εξωτερικά σύνορα, ότι θα πρέπει να προστατεύονται. Η ερώτηση που έχω να σα απευθύνω είναι πάρα πολύ απλή. Όταν πρόκειται για τα ελληνικά σύνορα με την Τουρκία, είπατε με σαφήνεια το θέμα αυτό και εσεί και άλλοι εδώ στην, ε, στο Κοινοβούλιο. Θα λέγατε τα ίδια σε ό,τι αφορά την Τουρκία και την παραβίαση του αέριου χώρου και του θαλάσσιου χώρου της Ελλάδας ή έχουμε διπλά μέτρα και σταθμά. Είναι ε, ευρωπαϊκά τα σύνορα ή δεν είναι ευρωπαϊκά τα σύνορα. Να είμαστε σαφείς. Τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης θα πρέπει να προστατεύονται, θα πρέπει να ασφαλίζονται, θα πρέπει να προστατεύονται ανεξάρτητα με το ποιος βρίσκεται από την άλλη πλευρά των σύνορων. Στην περίπτωση λοιπόν της Τουρκίας, στην περίπτωση της Ελλάδας κατά της Τουρκίας, ισχύει η ίδια αρχή. Η Ελλάδα αποτελεί εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει λοιπόν να πληρεί όλες ε, τις προϋποθέσεις της Συνδίκης Σέγγεν. Σα ευχαριστώ. Ο κύριος Τόμας για 1,5 λεπτό. Yes. Κύριε Αντιπρόεδρε, συμμεριζόμεθα την προσπάθεια την οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε μια αξιοπρεπή υποδοχή, να μοιραστούμε τους ετούντες ασύλου και να ενισχύσουμε τα μέσα συνεργασίας με τις χώρες εταίρους. Όλα αυτά τα μέτρα είναι θετικά. Τίθεται το θέμα της χρηματοδότησης των μέτρων αυτών και συνεπώς της ειλικρινιάς τους. Η συμφωνία που υπεγράφει εδώ και δύο μήνες εξάντλησε ουσιαστικά τα δημοσιονομικά περιθώρια. Η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγει ότι είμαστε καταδικασμένοι να προσπαθούμε με εφάνταστο τρόπο να βρούμε χρήματα. Τα χρήματα αυτά δεν υπακούν σε καμία τακτική δημοσιονομική διαδικασία και τα χρήματα για την Τουρκία το δείχνουν. Ενισχύεται ο προπολογισμό της Ένωσης χωρίς να φύγεται όμως το ανώτατο όριο του πολιετού δημοσιονομικού. Το υποκριτικό μήνυμα είναι ότι έτσι δεν θα πρέπει να ενισχυθεί η Ένωση. Ε, δυστυχώς ακούμε μισές αλήθειες, ακούμε άλοθη. Ας ε, προσπαθήσουν στο Συμβούλιο να μην κάνουν την Ευρώπη να ντρέπεται απαιτείται περισσότερη ευθύνη και απαιτούνται περισσότερα μέσα για την ανάληψη της ευθύνης. Φέτος είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε στην αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού. Πρέπει να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό της Ένωσης, να αναλάβει η Ένωση τις ευθύνες της. Σήμερα είπαμε με τον κύριο Μοσκοβισή για τα θέματα της φορολογίας των πολιεθνικών γιατί τα χρήματα από αυτούς τους φόρους να μην πηγαίνουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να καταργηθούν αυτοί οι στήροι ανταγωνισμοί φορολογικοί ανάμεσα στα κράτη-μέλη και εις βάρος της Ένωσης. Η κυρία Φωτίγκα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι απειλές προς την ε, ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η αποσταθεροποίηση αλλά και η ε, ρωσική πολιτική στην Ανατολή. Η μετανάστευση είναι ένα από τα κύρια αποτελέσματα. Δέχομαι ε, τη στήριξη προς την Τουρκία, αλλά και τα μέτρα στην Νότια Ευρώπη. Επίσης είμαι υπέρ της ε, υποστήριξης του Frontex και των νότιων μελών μας. Αλλά είμαι υπέρ και της στήριξης προς τη Γαλλία που ε, έκανε αυτή την επίκληση του συγκεκριμένου άρθρου της συνθήκης. Η Πολωνία έχει δεχθεί σχεδόν ένα εκατομμύριο κατά κύριο λόγο οικονομικούς μετανάστες. Δεν τους επιστρέφουμε, προσπαθούμε να τους βρούμε δουλειά και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, όμως ε, θα θέλαμε η Πολωνία να μην ε, στιγματίζεται ούτε στο Κοινοβούλιο, ούτε στον τύπο. Ευχαριστώ κυρία Εντφέλτ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλά έχουν ήδη υποθεί για το τι πρέπει να γίνει. Όμως, καλό θα ήταν να αναρωτηθούμε το εξής. Πώς θα μας κρίνει η ιστορία. Τι θα πούν τα εγχειρίδια της ιστορίας για αυτές τις συζητήσεις, ας πούμε, 100 χρόνια από σήμερα. Νομίζω θα πούνε ότι το 2016 ξεκίνησε με πολύ θετικό τρόπο, με ένα πραγματικό θαύμα την πρωτοχρονιά. Γιατί είδαμε ότι στην Ευρώπη έχουμε 500 εκατομμύρια φεμινιστές, δημοκράτες, ε, διαφωτισμένους που έχουν ε, κάθε σεβασμό για τα γενική δικαιώματα ξαφνικά. Αλλά εντάξει, πιο σοβαρά τώρα, δεν υπάρχει θρησκεία σε αυτά τα ζητήματα και να θυμίσω και στους Σουηδούς συναδέλφους και τους Βίκινγκς που πήγαν σε όλη την Ευρώπη, βίαζαν, σκότωναν και καταλήστευαν. Όμως τα ιστορικά εγχειρίδια θα μιλήσουν και για την απόλυτη παράλυση και ανικανότητα της μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο στην προσπάθειά της να επιλύσει ένα διαχειρίσιμο πρόβλημα. Γιατί είναι μεγάλη πρόκληση όντω, αλλά είναι απόλυτα διαχειρίσιμο. Τα ιστορικά εγχειρίδια λοιπόν θα μιλήσουν για την μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο που στρέφει την πλάτη στα παιδιά που πνίγονται, στα παιδιά που απάγονται από εγκληματικές οργανώσεις για να υποστούν εκμεταλλεύσει και καταχρήσει όταν οι γυναίκε γεννούν στα χωράφια. Και όλα αυτά από τη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο που κάθεται αδρανή και δεν κάνει τίποτα. Και ταυτόχρονα σπαταλούμε χρόνο μιλώντα ε, για την εθνική κυριαρχία για παράδειγμα που δεν όμω πληρώνει κανένα το ενίκιο. Δεν χρειαζόμαστε πιο πολλέ κόκκινε κάρτε ούτε παράλυση. Θέλουμε να μας γράψει ιστορία ως μία μαύρη περίοδο παράλυσης ή θέλουμε να είμαστε αρχιτέκτονες ενός μεγάλου βήματος προς το μέλλον και μιας νέας περίοδου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κατανοώ αυτό που είπατε για τις κόκκινες κάρτες, αλλά δέχεστε μία μπλε κάρτα. Κύριε Σόνια. Ναι, κοιτάξτε. Παρά το γεγονός ότι εν μέρη συμφωνώ με αυτά που έχετε αναφέρει ως τώρα, θέλω να θέσω μια απλή ερώτηση. Ποια θα ήταν η λύση. Όσο μιλούσαμε για διεύρυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι ήταν ενθουσιασμένοι. Τώρα που μιλάμε για εμβάθυνση, βλέπω ότι αποκλίνουν οι απόψει στη Γερμανία, στην Ουγγαρία. Ποια θα ήταν λοιπόν η λύση. Ξέρετε, δεν είναι και καμιά τρομερή επιστήμη. Υπάρχουν πολλές λύσεις επιτάπητος. Και το Κοινοβούλιο έχει προτείνει και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Συμβούλιο μάλιστα έχει αποφασίσει επί ορισμένων λύσεων. Καλό βέβαια θα ήταν να τις εφαρμόσουν κιόλα τι αποφάσει που έχουν λάβει. Θα μπορούσαμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Δεν έχουμε ούτε χρόνια ούτε δεκαετίε. Τώρα πρέπει να πάρουμε αποφάσει. Το θέμα δεν είναι καινούριε προτάσει και ιδέε. Το θέμα είναι η ανάληψη δράση η λήψη αποφάσεων, η εφαρμογή των όσων έχουν συμφωνηθεί. Εγώ αυτό προτείνω, αγαπητέ συνάδελφε. Ευχαριστώ η κυρία Άντερσον για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάνω από 10.000 παιδιά, όπως διαβάσατε, έχουν εξαφανιστεί στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μάθαμε πρόσφατα και δυστυχώς υπάρχει μια απόδειξη έμπρακτη πλέον της πλήρους αποτυχίας της ευρωπαϊκής πολιτικής. Τα ευρωπαϊκά όργανα απέδειξαν την έλλειψη ανθρωπισμού που τα χαρακτηρίζει απέναντι σε αυτή την κρίση εμείς κάνουμε ότι δεν βλέπουμε. Δυστυχώς οι πρόσφυγες έκαναν ένα τεράστιο και δύσκολο ταξίδι για να αποφύγουν την τραγωδία και διέσχισαν με εξαιρετικά κακούς όρους ε, την Τουρκία, την θάλασσα και έφτασαν στο τέλος να κρατούνται ουσιαστικά λόγω της πολιτικής την οποία ακολουθούν οι περισσότερες χώρες οι πρόσφυγες οι οποίοι προσπαθούν να ξεφύγουν από τις βόμβες συνάδελφοι θα πρέπει να τους αγκαλιάσουμε αλλά αντί να το κάνουμε αυτό τους βάζουμε σε ε, στρατόπεδα ή τους στέλνουμε στην αγκαλιά των ε, εγκληματιών αυτών που τους περνούν από τη μία χώρα στην άλλη κλέβοντας ε, τα λίγα που έχουν στην διάθεσή τους. Και ξέρουμε επίσης και τα τρομακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μικρά παιδιά τα οποία τα εκμεταλλεύονται σεξουαλικά και τα βάζουν να εργάζονται με καταχρηστικούς όρους. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ε, δώσουμε την ασφάλεια την οποία αναζητούν επιτέλους. Ευχαριστώ κυρία Κέλλερ ένα λεπτό. Thank Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι με επαναπρόθεση αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Συμφωνώ και ελπίζω ότι με τη δήλωσή σας σε ό,τι αφορά τις προτάσεις πολιτικής για την επιστροφή των προσφύγων στην Τουρκία, όπου δεν θα προστατεύονται ως πρόσφυγες και που ενδεχομένως θα ε, επιστρέφονταν στην Τουρκία, στην Συρία θα έλπιζα να είσαστε και πάρα πολύ σαφείς και προς τους ε, ηγέτες του Συμβούλιο που προτείνουν στην Ελλάδα να κλείσει τα σύνορά της. Και δεν μπορεί κανείς να κλείσει τα σύνορά του εκτός και αν ε, αφήσει τον κόσμο να πνιγεί και παραβιάσει και τη συνθήκη της Γενέβης. Αυτό θα πρέπει να είμαστε... Σε γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, γιατί αν συμβεί αυτό η Ευρώπη θα χάσει τον λόγο που υπάρχει. Είναι μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σίγουρα, αλλά μπορούμε να τα ανταπεξέλθουμε από κοινού. Και πρόκειται για μια στιγμή που και πάλι βλέπουμε ότι χρειαζόμαστε την Ευρώπη πιο πολύ παρά ποτέ και ότι θα πρέπει από κοινού να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση αυτή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άρνοτ για ένα λεπτό. Είδαμε επιθέσεις κατά των προσφύγων και μεταναστών σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες και είδαμε και επιθέσεις από μετανάστες στην Κολόνια και σε άλλες πόλεις γιατί βιαζόμαστε να τις καταδικάσουμε ως ομές επιθέσεις από του προς τους μετανάστες, αλλά καμία πλευρά δεν αναγνωρίζει και τις δύο επιθέσεις. Δεν θα πρέπει να καταδικάζουμε οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια, ανεξάρτητα από ποιος τη διαπράττει. Η βία που είδαμε από άτομα θα πρέπει να την καταδικάζουμε. Και όπως και τη βία από τους αντιφασίστες όπως αυτοαποκαλούνται. Να θυμόμαστε ότι οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποτύχει παταγωδός όταν χρειάστηκαν για μια τεράστια ανθρωπιστική ανταπόκριση και απάντηση. 2,5 εκατομμύρια Τούρκοι ε, πρόσφυγες και πολλά εκατομμύρια από άλλες χώρες. Οποιαδήποτε πρόβλημα έχει παρουσιαστεί σήμερα ήταν προβλέψιμο και το αγνόησε πολύ απλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Ανεμπέκα. Ο Ευχαριστώ. Η προσφυγική κρίση έχει αποδείξει δύο στοιχεία. Την αμέλεια ε, τη Ένωση ό,τι αφορά τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και την έλλειψη κοινών αποφάσεων σε ό,τι αφορά την επίλυση τη προσφυγική κρίση στα κράτη-μέλη. Οι ευρωπαϊκέ αρχέ έχουν λάβει κακέ αποφάσει του τελευταίου μήνε και σήμερα βλέπουμε τι αρνητικέ κοινωνικέ προεκτάσει που αφορούν και πλήττουν κυρίως ε, τα παιδιά και τις γυναίκες. Και η κατάσταση γίνεται ολοένα και χειρότερη. Πρώτον, πώς μπορούμε να ασφαλίσουμε τα σύνορα της Σέγγεν όταν είναι αδύναμα και ευάλωτα τα εξωτερικά σύνορα. Τα ξεχάσαμε αυτά όταν επιβάλαμε στα κράτη-μέλη ε, ποσοστώσεις σε ό,τι αφορά τις προσφυγικές ροές. Το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να προστατεύσει τα σύνορά της και ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει μέτρα προστασίας μας οδηγεί μόνο στο συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προληπτικά θα έπρεπε να ε, υιοθετήσει μέτρα προστασίας για τα κράτη-μέλη δεν μπορούμε μόνο να μιλούμε για τα λεγόμενα εγκλήματα των προσφύγων κατά των Ευρωπαίων πολιτών. Να μην ξεχνάμε ότι πέρσι δεχθήκαμε ε, πρόσφυγες από αυτές τις χώρες ενώ δεν δεχθήκαμε ε, να εντάξουμε στην ε, Σέγγεν χώρες όπως είναι η Ρουμανία για παράδειγμα. Πώς το εξηγούμε αυτό. Θα υπάρξει χάσμα πολιτισμών όπως είτε μας αρέσει είτε όχι και θα υπάρχουν και εντάσει μεταξύ των πολιτών και των ε, προσφύγων. Οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν θα πρέπει ε, να, να αισθάνονται μειονεκτικά επειδή ανήκουν σε κάποια ε, θρησκευτική ομάδα. Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά την πολιτική αυτοκτονία των ανοιχτών θυρών, ερχόμαστε τώρα στην απογοήτευση. Πρώτα απ' όλα, οικονομική απογοήτευση. Όσοι θεωρούν ότι είμαστε μόνο οικονομικοί φορεί, ανεξάρτητα από ε, την κουλτούρα μα, βλέπετε τώρα πόσο λάθο ήταν αυτό. Ε, πέραν του νέου οικονομικού θαύματο, ξέρουμε τώρα ότι ε, η μεγάλη πλειονότητα αυτών των ε, νέων ανδρών δεν θα μπουν στην αγορά εργασία και ότι δεν έχουν ε, ε, την ίδια κατάρτιση. Και πολιτισμική όμως απογοήτευση. Βλέπουμε ότι ο πλουραλισμό, ο πολιτιστικός πλουραλισμός ε, αποτυγχάνει από τα πρόσφατα φαινόμενα που βλέπουμε με τις παρενοχλήσεις, επιθέσεις και το καθεξής και με την τρομοκρατική επιλή βεβαίω. Ε, και βλέπουμε ότι πρέπει να ότι η πραγματική Ευρώπη ε, μπορεί να αποτελέσει μόνο ε, μια σε βάθος συνεργασία κυρίαρχων κρατών. Ευχαριστώ. Γαμπριέλ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποιοι από εμά είπαν ότι πρόκειται για ακόμα μία συζήτηση για τη Σέγγεν και του πρόσφυγε. Πράγματι, είναι ακόμα μια τέτοια συζήτηση, γιατί μία από τις βασικές αξίες ε, τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η ελευθερία, δικαιοσύνη ε, και ασφάλεια, έχουν τεθεί σε κίνδυνο και αναπόκειται σε εμά να υπεραμεινθούμε των ευρωπαϊκών αξιών ακόμα και σε περίοδους κρίσης κάνοντας λόγο για τις ευρωπαϊκές αξίε, πρέπει να μιλήσουμε και για τις ενέργειες που θα αναλάβουμε. Τα λόγια μας να γίνουν πράξεις. Ας επικεντρωθώ πρώτα στη Σέγγεν. Όλοι ξέρουμε ότι η Σέγγεν αυτή τη στιγμή ε, κινδυνεύει. Πρέπει να συνεχίσουμε να εξετάζουμε την διατήρηση ε, τη Σέγγεν. Γιατί εάν καταργηθεί, αυτό θα επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τι οικονομίε μα και τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Εάν ελέγξουμε τα ευρωπαϊκά σύνορα τη Ένωση, θα καταφέρουμε αποτελεσματικά να προστατεύσουμε και τη Σέγγεν. Πολλέ χώρε ε, συμμορφούνται με τι υποχρεώσει του στα εξωτερικά σύνορα. Όμω συμμορφούνται και με τι διαδικασίε καταχώρηση, καταγραφή των μεταναστών και επιστροφή του. Όπω είναι η Βουλγαρία, για παράδειγμα. Είναι ε, μια περίπτωση χώρας που έχει πετύχει θετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την ε, διακίνηση και την καταπολέμηση της διακίνησης ε, ανθρώπων και την προστασία των συνόρων της. Της αξίζει λοιπόν της Βουλγαρίας να μείνει στη Σέγγεν. Πρέπει να εντοπίσουμε τις τρίτες χώρες, να πάρουμε και τα αντίστοιχα μέτρα, αλλά να μην ξεχνάμε τις αρχές μας. Ευχαριστώ. Κύριε Βαντενχόλτσερ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τις 9 Σεπτεμβρίου που έγινε η δήλωση αυτή για την κατάσταση της Ένωσης ξέρουμε ότι θα πρέπει να γίνει και την, στην επόμενη, στις επόμενες ολομέλειες ασχολούμασταν διαρκώς με τα προβλήματα αυτά τα οποία όμως διωγγώνονται και μεταξύ έχουν φτάσει να υπονομεύουν όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν αλλάξει κάτι επί της ουσίας. Αν συνεχίσουμε να κάνουμε ιδεολογικές ε, συζητήσεις για ίσονος σημασία τέτοια θέματα, ε, θα χάσουμε το παιχνίδι. Φτάνει πια. Κάτι θα πρέπει να αλλάξει. Και ελπίζω και υπολογίζω στην αντικειμενικότητα των Ολλανδών την περίφημη για να ξεπεραστεί αυτό το μπλοκάρισμα γιατί χρειάζονται τα μέσα λοιπόν για τις χώρες προέλευσης και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία στα πλαίσια γειτονική χώρας και να εγγυηθούμε την ασφάλεια των συνόρων και χρειαζόμαστε και αλληλέγγυα κατανομή στην Ευρώπη. Αλλά όλα αυτά θα λειτουργήσουν μόνο αν επιτέλους δημιουργηθούν αυτά τα hot spots που έχουμε υποσχεθεί, κύριε Επίτροπε. Και νομίζω ότι επιτέλους θα πρέπει να καταχωρίζουμε και τον κόσμο που καταφθάνει. Γιατί τότε δεν θα συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν και συνέβησαν με τους νέους αυτούς ανθρώπους που, ουσιαστικά χάθηκαν από πρόσωπο γη. Χρειαζόμαστε πιο κανονικές και φυσιολογικές ε, καταστάσεις και πιο πολύ πρακτική πολιτική, ρεάλ πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Στίβενς για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Όποιος πιστεύει ότι η μαζική εισρωή ετούντων άσυλο και τείχο διακτών μπορεί να ε, συνδυαστεί με τις αρχές της κράτους πρόνοιας, ε, κάνει μεγάλο λάθος. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Αυτό το κατανοεί άλλωστε και η Ολλανδική Προεδρία, ότι οι αιτούντες άσυλο όσοι που, θέλουν να, ε, που θέλουμε να επιστραφούν στην Τουρκία με φέρι, με πλοία, ουσιαστικά θέλουν να έρθουν στην Ήπειρό μας. Εμείς στο κόμμα μου είμαστε υπέρ μιας πολιτικής ε, επιστροφής, ενεργούς. Πόσο αλλιώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις ροές. Δεν ε, φτάνει να φυλάμε τα σύνορα. Βλέπουμε λοιπόν καλές προτάσεις στην Ολλανδική αυτή, στο Ολλανδικό αυτό έγγραφο για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Το γεγονό ότι δεν συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοι προέκυψε και από τις παρεμβάσεις των συναδέλφων σήμερα και τις τελευταίες ημέρες. Κάποιοι προτείνουν να δώσουμε χρήματα στους ετούντες άσυλο, στους καταβλισμούς προσφύγων. Αυτό θεωρώ ότι θα έκανε τις τιμές να αυξηθούν στους καταβλισμούς αυτούς. Και αυτό ουσιαστικά θα σήμερα θα, ξεκίνησε, θα ξεκινούσε να χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τους διακινητές ανθρώπους. και η χορήγηση τουριστικής βίζας ε, προς τους ε, πρόσφυγες. Όλα αυτά αποτελούν μη ρεαλιστικές προτάσεις με πραγματικά παράλογες συνέπειες. Ε, συνάδελφοι, ας κάτσουμε να κοιτάξουμε μαζί με το Συμβούλιο επικοδομητικά τι μπορούμε να κάνουμε. Το χρωστάμε σε όλους. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος, αποδέχεστε μια μπλε κάρτα. Κυρία Στίβενς από τον κύριο Λάμστορφ. Mr. Uh, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Στίβενς. Και συμφωνώ με τη συστηματική προσέγγιση που προτείνεται και πιστεύω ότι είναι σωστό ότι θα πρέπει να ελέγχονται τα εξωτερικά σύνορα προκειμένου να παραμείνουν τα εσωτερικά σύνορα Σέγγεν ε, ανοιχτά. Αλλά πώς ε, λέτε στα σοβαρά ότι και ε, μέρη της κόμματός σας θα πρέπει να γίνουν πυροβολισμοί, να πυροβολούνται στα ιστορικά σύνορα ε, γυναίκες και παιδιά, άνθρωποι. Αυτό το έχουμε δει γραπτά. Δεν είναι μια τυχαία δήλωση αυτή που αναφέρω. Και θα ήθελα να πω με μεγάλη σαφήνεια το εξή ε, από πλευράς του κόμματός μας ότι ε, αποστασιοποιούμαστε απόλυτα από τη δήλωση αυτή. Το να περιβαλλείται ο κόσμος είναι τελείως απαράδεκτο και νομίζω ότι είμαι σαφής σε αυτά που λέω. You still have one more. Έχετε ακόμα μία μπλε κάρτα από την κυρία Ιντφέλτ. Κυρία Ιντφέλτ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λίγο με προκαλέσατε όταν είπατε ότι υπάρχουν άνθρωποι εδώ που μιλούν για ανεξέλεκτη μετανάστευση και τουριστικές βίζες προς τους έτοντες άσυλο. Και θα ήθελα να ακούσω ποιον να αν τα λέει αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν άκουσα τίποτα τέτοιο και νομίζω ότι καλό είναι να έχουμε μια σαφήνεια στη συζήτησή μας. Er Υπάρχουν ε, κάποιοι συνάδελφοι από κάποιες ομάδες που μιλούν για ανθρωπιστικές βίζες, θεωρήσεις, ως ένα νόμιμο κανάλι αυτό δεν μπορείτε να το αρνηθείτε. Σας ευχαριστώ. Τελίτσκα, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε, Υπουργοί. Νομίζω ότι σήμερα, αν βάζαμε την ταινία της τελευταίας ε, ε, συνόδου, δεν θα πρόσεχε κανείς τη διαφορά. Τόσο λίγες είναι οι διαφορές. Και δυστυχώς δεν βλέπουμε αποτελέσματα. Ο Υπουργός μιλά για hot spots. Ναι, εντάξει, ίσως σημειώθηκε κάποια πρόοδος. Αλλά νομίζω ότι η τρέχουσα κατάσταση εξακολουθεί να είναι απαράδεκτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί και μιλάει για ανεπαρκή εφαρμογή. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό αποτελεί την πραγματικότητα. Έχουμε κάνει λάθη. Και κάποια μέτρα προτάθηκαν την ακατάλληλη στιγμή και δεν ήταν τα σωστά. Αλλά αληθεύει επίσης ότι δεν εφαρμόζουμε τις αποφάσεις του Συμβουλίου. Το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει για το ότι θέλουμε μια ενωμένη Ευρώπη και θα πρέπει για το σκοπό αυτό να φροντίσουμε κανείς να μην μπορεί να κάνει κάτι, να μην μπορεί να ξεφεύγει χωρίς να διαβουλεύεται με τους εταίρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και τα δύο χρειάζονται. Χρειάζεται μια ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σταματήσουμε να κατηγορούμε και να επιρρύπτουμε ευθύνε ο ένα τον άλλον και μια μετατόπιση τη πολιτική. Υπάρχουν θέματα ε, προστασία ε, των συνόρων, ε, Frontex, ε, γρήγορη ανάπτυξη δυνάμεων, έλεγχο των επιστροφών. Και τη στιγμή που θα υπάρξουν και θα αποδώσουν καρπού, σε αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να υπάρξει και κατανομή των ευθυνών. Μετά από 70 χρόνια θα διαρωτάτε η ανθρωπότητα πώς είναι δυνατόν να φέρεται έτσι η Ευρώπη εις βάρος ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο πως είναι δυνατόν άνθρωποι να κατάσχουν τα τιμαλφή και τα χρήματά τους από τους πρόσφυγες. Η άκρα δεξιά δεν είναι μόνη η οποία ακολουθεί ξενοφοβικές απόψεις και ρατσιστικές απόψεις. Αρκετές κυβερνήσεις και αρκετά κοινοτικά όργανα ακολουθούν την ίδια ε, γραμμή, ε, δυστυχώς την ίδια μορφή βίας με διαφορετικούς τρόπους και μιλούν για εισβολή μεταναστών. Ε, χτες έγινε μια επιδρομή ακροδεξιών στους δρόμους της Σουηδίας ε, με επιθέσεις εις βάρος των μεταναστών και πολλοί έκαναν παρελάσεις με σβάστηκες εις βάρος βέβαια των μεταναστών πάντα. Βαλέρο ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος μας είπε ότι απαιτούνται λύσεις οι οποίες να είναι αντίστοιχες με τις αξίες μας. Ποιος μπορεί να διαφωνήσει με αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτές οι λύσεις που προτείνονται δεν σέβονται τις αρχές μας. Σαν παράδειγμα ε, η εισαγωγή εσωτερικών ελέγχων είναι εναντίον των ισχυουσών ρυθμίσεων, εναντίον του Σέγγεν <laughs> και επίσης δεν μπορούμε να τις δεχτούμε. Δεν μπορούμε να δεχθούμε επίσης τις επαναπροωθήσεις. Δεν μπορούμε να δεχθούμε τις συστηματικές αρνήσεις χορήγησης ασύλου. Εάν πράγματι θέλουμε να σεβαστούμε τις θεμελιώδεις μας αξίες θα πρέπει να αναρωτηθούμε. Αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εδώ γιατί έρχονται και τότε θα φανούμε αλληλέγγυοι και δεν πρέπει να δεχόμαστε μία χώρα να δέχεται χιλιάδες μετανάστες και κάποιες άλλες χώρες γύρω γύρω να δέχονται κάποιες εκατοντάδες. Ε, η έλλειψη αυτής της σωστής πολιτικής οδηγεί χώρες όπως η δική μου, τη Σουηδία, να παίρνει μέτρα τα οποία στην ουσία θέτουν σε κίνδυνο την Ευρωπαϊκή Συνοχή. Νομίζω ότι οι εγωισμοί των κρατών μελών δημιουργούν συνθήκες απαράδεκτες, μετατίθενται οι ευθύνες και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από το τι θέλει να κάνει και από την καλή βούληση του Ερντογάν. Η Ευρώπη μεταφέρει τα προβλήματά της στην Τουρκία, αλλά στην ουσία βλέπουμε τι συμβαίνει στην Τουρκία. Τα χρήματα κανονικά θα έπρεπε να πάνε στους μετανάστες. Πώς ε, πιστεύετε ότι θα το εξασφαλίσετε αυτό. Πιστεύετε ότι θα είναι εύκολο να ελέγξετε τον τρόπο χρησιμοποίησης των τριών δις. Τον τελευταίο καιρό πολλοί φεύγουν απελπισμένοι προς την Ευρώπη με τη συνενοχή των τουρκικών αρχών. Γιατί να μην συνεχιστεί το ίδιο πράγμα. Εγώ θα πάω σε μία εβδομάδα στην Τουρκία να συλλέξω περισσότερες πληροφορίες για μία κατάσταση απαράδεκτη. Αλλιώ ένα λεπτό συνάδελφοι, ο τρόπος με τον οποίο θα έλεγα συμπεριφέρεται η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη σφραγίδα της αποτυχίας, την αποτυχία του Σέγγεν, γιατί πολλές χώρες αποκαθιστούν τα σύνορα, γιατί τα σύνορα είναι κομβικό σημείο της πολιτικής των χωρών. Ταυτόχρονα ένα ανθρώπινο δράμα, ένα εκατομμύριο έρχεται, τρία εκατομμύρια περιμένουμε. 10.000 παιδιά έχουν εξαφανιστεί. Εκρηκτικές καταστάσεις όπως την Κολονία, όπως το Καλέ και το 60% αυτών των μεταναστών είναι απλοί οικονομικοί μετανάστες και όχι πρόσφυγες. Τουρκία, χώρα που συμπεριφέρεται άσχημα στα ανθρώπινα δικαιώματα, παίζει με την Ευρώπη με το ένα χέρι και με το άλλο παίζει με το Ισλαμικό κράτος και από την άλλη η κακοφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι με αισθήματα ευγενή υπάρχουν αλλά όλα πάνε χάλια. Ακόμα και το ελεγκτικό συνέδριο λέγει ότι οι πολιτικές μας είναι ανεπαρκείς και οικονομικά ανέφικτες. Λοιπόν πρέπει ο λαός να αποφασίσει, ο λαός είναι κυρίαρχος. Ο κύριος Επιτίδιος ένα λεπτό. Η αρχαία ελληνική λέξη πανικός είναι ο πλέον ακριβή χαρακτηρισμό του τρόπου με τον οποίο η ευρωπαϊκή ένωση αντιμετώπισε και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το σοβαρό πρόβλημα των προσφύγων και των μεταναστών. στην αρχή αδιαφόρησε και στη συνέχεια όταν το θέμα πήρε ανεξέλεγκτε διαστάσει άρχισε τα ανατολίτικα παζάρια με την τουρκία για το πόσα χρήματα θα πρέπει να τη δώσει ώστε να απαγορεύσει στα κυκλώματα τη διαφθορά τη χώρα στα οποία συμμετέχουν και κρατικοί λειτουργοί να μην προωθούν στην ελλάδα παράνομου μετανάστε η τουρκία όπω ήταν αναμενόμενο εκμεταλλεύτηκε αυτή την ευκαιρία και άρχισε να εκβιάζει την ευρωπαϊκή ένωση για να ζητά περισσότερα χρήματα από τα τρία δισεκατομμύρια που έχουν εγκριθεί να λάβει. οφείλετε να αντιληφθείτε ότι η τουρκία δεν είναι ένα αξιόπιστο συνομιλητή δεν εκπληρώνει τι υποχρεώσει τη και εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για να προωθήσει τα εθνικά τη συμφέροντα. εάν θελήσουμε να πιέσουμε οικονομικά την τουρκία θα πρέπει για κάθε παράνομο μετανάστη που έρχεται από την τουρκία στην ελλάδα να εξασφαλίσουμε να βάλουμε ένα βαρύ πρόστιμο το οποίο να αφαιρείται από τα χρήματα που πρέπει να λάβει η τουρκία. θα της δώσουμε έτσι να καταλάβει ότι ξέρουμε να κάνουμε και εμείς οικονομικά ανατολίτικα παζάρια. Ευχαριστώ. Είναι ανεξέλεγκτη αυτή η διαδικασία και ουσιαστικά μόνο ένα κλάσμα καταγράφεται των ε, ανθρώπων που καταφτάνουν. Τα hot spots δεν λειτουργούν. Θα πρέπει λοιπόν να μην έχουμε αυταπάτες. Δεν ε, συνδράμει αυτό στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Το σύστημα πολύ απλά δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο φορτίο και έτσι δημιουργούνται τριβές μεταξύ των κρατών μελών. Χιλιάδες άτομα καταφθάνουν κάθε χρόνο και αυτό αποστατεροποιεί την Ευρώπη. Η σταθερότητα της Ευρώπης και η προστασία της Ευρώπης είναι το πιο σημαντικό ζήτημα. Και αυτό το βλέπουμε από το καλοκαίρι και μετά. Οι πιο πολλοί πρόσφυγες και οι πιο πολλοί μετανάστες δεν έχουν δικαίωμα σε άσυλο. Οι πιο πολλοί είναι οικονομικοί μετανάστες, νεαροί άνδρες. Και σε ό,τι αφορά τα παιδιά, συχνά είναι ε, νεαροί 14 έως 18 ετών. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρώπη να διαχειριστεί αυτή την κρίση, άλλως θα έχουμε προβλήματα. Μία τεχνική λοιπόν, είναι τεχνικό το ζήτημα. Μόνο μία σταθερή Ευρώπη μπορεί να δείξει αλληλεγγύη και να βοηθήσει αυτούς που πραγματικά έχουν δικαίωμα σε άσυλο. Ευχαριστώ. Ενάμιση λεπτό, κύριε Φλέκενστάιν. Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να μακρηγορήσω. Είναι πραγματικά πάρα πολύ συναρπανιστική η συζήτηση. Βλέπουμε ότι έχουμε 10% των συναδέλφων εδώ και τα έδρανα τα μπροστινά είναι άδεια. Δεν κατηγορώ βέβαια τους συναδέλφους του το 90% που λείπει θα έχουν όρεξη να δουλέψουν και όχι να ακούσουν για έκτη φορά αυτά που έχουμε ήδη ακούσει και δεν έχω και όρεξη να επαναλάβω πάλι και εγώ αυτά που είπα και έχω πει προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ούτε εσάς μπορώ να σας ξανακούσω που λέτε εκ νέου πόσο καλά εργαστήκατε κι εσείς, πόσο καλά εργαστήκαμε κι εμείς και πόσο δεν, καλά δεν εργάστηκε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όλα αυτά είναι πραγματικά δυσβάσταχτα. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει και κάποιος που μας ακούει στο ίντερνετ θα πρέπει να κάτσουμε και να σκεφτούμε από κοινού πώς μπορούμε τα μέτρα που πρότεινε ο κύριος Φερχόφστατ ε, να πετύχουμε κάτι παραπάνω. Δεν ε, έχω λοιπόν διάθεση και δεν έχει κανένα νόημα να με γρηγορήσω άλλο, γι' αυτό και σας χαρίζω και 22 δευτερόλεπτα. Αλλά αχώ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, πέρυσι οι μεταναστευτικές πιέσεις μετατοπίστηκε από την Κεντρική Μεσόγειο προς την Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα δεν καταγράφει τους μετανάστες όπως θα έπρεπε, το οποίο είναι κατανοητό από ελληνική άποψη, καθώς ο μηχανισμός μεταγκατάστασης ε, δεν λειτουργεί και ούτε πρόκειται να λειτουργήσει. Η ανάπτυξη, η εξέλιξη αυτή μάλλον δεν είναι βιώσιμη. Για παράδειγμα, η Γερμανία αναμένεται να δαπανίσει 50 εκατομμύρια ευρώ για τους μετανάστες για φέτος και του χρόνου εκατοντάδες χιλιάδες νέοι ε, μετανάστες ε, στην Γερμανία, Σουηδία, Φιλανδία και αλλού δεν έχουν καμία προοπτική εξέβρεσης, ε, ανέβρεσης σε μια θέση εργασίας ή αξιοπρεπούς ζωής. Οι συνέπειες θα είναι πολύ σοβαρές. Πρέπει να έχουμε το θάρρος να παραδεχθούμε ότι δεν μπορούμε να λύσουμε την κρίση με τον να περισσότερους ανθρώπους. Όσους και να πάρουμε, θα υπάρχουν ακόμα εκατομμύρια που θα έρχονται από την Αφρική και τη Μεσανατολή. Θα πρέπει να αρχίσουμε συστηματικά ε, τις αποθήσεις, τα pushbacks, τουλάχιστον στην Αυστραλική Μεσόγειο ε, και στα Δυτικά Βαλκάνια. Να στέλνουμε πίσω τους ε, μετανάστες και εκεί να ε, επεξεργαζόμαστε τις αιτήσει. Και... Γιατί οι δάλος θα μένουν εδώ είτε του χορηγηθεί άσυλο είτε όχι. Θα πρέπει να σταματήσει το asylum shopping. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να υποχρεούται να ε, αρνηθεί και να απορρίψει τις αιτήσει ανθρώπων που έρχονται από άλλο κράτος μέλος. Ευχαριστώ η για σε λεπτό. Ευχαριστώ. Ήθελα να πω στα θεσμικά όργανα, στο Συμβούλιο και την Κομισιόν, ότι το μήνυμα που μα ε, μετέδωσαν πριν από ορισμένε ημέρε, ε, που αψηφά ουσιαστικά την ε, Ελλάδα και τη βάζει εντό αγωγικών σε καραντίνα, δεν ήταν ένα μήνυμα θετική πολιτική θέλετε να διατηρηθεί η Σέγγεν, όπω όλοι. Α διατηρήσουμε λοιπόν τα ελληνικά σύνορα ω ευρωπαϊκά σύνορα και να μην αρχίσουμε να ρίχνουμε ένα την ευθύνη στον άλλον. Εγώ πήγα στη Λέσβο το Σαββατοκύριακο, είδα τη δουλειά που κάνει η ελληνική ακτοφυλακή και συνοριοφυλακή, είδα τα ελληνικά σκάφη, περισσότερα από ότι τα σκάφη της Frontex. Είδα τη δουλειά που έκαναν ε, υποδοχής και διάσωσης των προσφύγων ε, στη θάλασσα. Ε, και επισκέφθηκα και τα hot spots στη Λέσβο, που είναι ένα από τα νησιά με, τη, με τις μεγαλύτερες ζωές στην Ευρώπη. τον Ιανουάριο είχαμε 33.000 αφήξεις που, τις οποίες διαχειρίστηκαν οι Έλληνες ε, και με τη μικρή και περιορισμένη βοήθεια του Frontex. Πράγματι γίνεται έλεγχος, καταγραφή, φωτογράφηση. Γίνεται δουλειά λοιπόν. Επομένως πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη μεταξύ μας και μετά να πάρουμε και αποφάσεις. Η πρώτη απόφαση που ζητώ είναι να απαιτήσουμε από την Τουρκία να σταματήσει η διακίνηση να σταματήσει τα κυκλώματα. 3.000 ανενήλικα, χίλια συγγνώμη, αναενήλικα, χίλια αν, για ανήλικο και χιλιάδες ε, ε, σωσίβια που συνήθως είναι και ψεύτικα. Πρέπει λοιπόν να σταματήσει όλη αυτή η προσπάθεια. Ε, ναι, Θα δεχθείτε μια μπλε κάρτα. Okay. Madam James. Thank you very much, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα μια έκκληση, ένα αίτημα. Η Τουρκία να κάνει περισσότερα. Η συνάδελφος που το ζήτησε αυτό πιστεύει ότι μήπως θα πρέπει να επιταχύνουμε και την Τουρκία στο να ενταχθεί στην Ένωση με όλα τα πλεονεκτήματα τα οποία θα φέρει είσοδο της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Εγώ είμαι αντίθετη πάντα για την είσοδο της Τουρκίας στην Ένωση. Νομίζω ότι θα ήταν λάθος για μας. Μπορούμε να σκεφτούμε ίσως μια Ευρωπαϊκή Ένωση πολλών κύκλων, ομόκεντρων βέβαια, αλλά όχι όμως μέλος. Μπορούμε όμως να έχουμε με την Τουρκία λίγο πιο έντονες σχέσεις, να υπάρχει περισσότερο πολιτικό θάρρος και βούληση σε μας απαιτούμε από τους Τούρκους να εμποδίσουν τους εγκληματίες πριν συζητήσουμε μαζί τους. Και φοβάμαι ότι θα δώσουμε αυτά τα τρία δι στην Τουρκία, δεν τα έχουμε αυτά τα λεφτά και ότι αν τα δώσουμε ξαφνικά θα σταματήσουν οι πρόσφυγες. Αποκλείεται. Βεργιά ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε μια ακόμα συζήτηση, μια ακόμα αποτυχία, μια ακόμα χειροτέρευση της κατάστασης. Η απάντηση δεν είναι στο ύψος του προβλήματος. Αυτή οι λίγοι τελικά σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού της Ευρώπης απειλούν λέει τη συνοχή της Ευρώπης. Ντροπή. Ε, επιτιθέμεθα στην Ελλάδα μια από τις πιο φτωχές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δέκα φορές μικρότερη από τη Γερμανία και πρέπει να κάνει το χωροφύλακα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλιώς υποτίθεται θα τους διώξουμε. Κανένας μήπως δεν σκέφτεται το πώς εξελίσσονται οι μεταναστευτικές ροές ε, στην αρχή του 2015 στην Κεντρική Ευρώπη. Προφανώς και έχει η Τουρκία ευθύνες και πρέπει να αναρωτηθούμε τι θα γίνει με τις ευθύνες αυτές να δούμε πώς χρησιμοποιούνται και τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ελεκτικό συνέδριο δημοσίευσε μια έκθεση, πρέπει να την εξετάσουμε. Και τι συνέχεια θα δώσουμε στην έκθεση της Europol για τα 10.000 παιδιά που χάθηκαν στην Ένωση. Η κυρία Εύα ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, τα τέσσερα θέματα αυτής της συζήτησης δείχνουν την ηθική αποτυχία και κατάπτωση της Ένωσης. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δεν έχει τίποτα να πει όταν τα μέλη της παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και αγνοούν τα ευρωπαϊκά καταστατικά κείμενα. Δυστυχώς αφήνουμε μια χώρα να προχωρά στην κατάσχεση των, των χρημάτων και των τιμαλφών των μεταναστών βλέπουμε ότι η Ολλανδή θέλει να κάνει ανταλλαγές προσφύγων με μια χώρα που ξέρουμε ότι δεν σέβεται τα δικαιώματά τους. Και ένα τμήμα της άκρας δεξιάς κάνει εγκληματικές προτάσεις έτσι ώστε να, να ποινικοποιήσει α, τους ανθρώπους της κοινωνίας των πολιτών που σώζουν από τον βέβαιο θάνατο απειλούμε την Ελλάδα, απειλούμε τους Έλληνες που με τα λίγα μέσα που έχουν τιμούν τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχουν χώρες βέβαια όπως η Γερμανία που σέβεται την, κοινωνική, την κοινοτική αλληλεγγύη αλλά δυστυχώς οι περισσότερες χώρες αγνοούν τις εκκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη δυστυχώς σήμερα. Αποδέχεστε μπλε κάρτα από τον κύριο Μπονάνο. Yes. Okay. Mr. Bonanno. Ακούγοντας τη συνάδελφο θα ήθελα να κάνω ένα ερώτημα. Εσείς πόσους πρόσφυγες έχετε πάρει στο σπίτι σας, είστε τόσο γενναία θα έχετε πάρει πολλούς, πόσους. Η Γαλλία πρέπει να υποδεχθεί πρόσφυγες, πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της και μέχρι τώρα νομίζω έχει δεχθεί 160.000 ή μάλλον από τις 160.000 έχει πάρει μόνο 62. Η Νορβηγία η οποία έχει προχωρήσει σε αυτό που έπρεπε είχε υποσχεθεί 10.000 μείωσε την ποσόστοση σε 7.000 και τώρα με μείον 28 επαναπροώθησε 28 σύρους στα σύνορα της Σουηδίας δυστυχώς και είναι η πιο πλούσια χώρα της Ευρώπης. Άνεμαν σε ένα λεπτό. Ο κύριος Μπάτεν δεν είναι στην αίθουσα. Ε, Συνάδελφοι, μου κάνει εντύπωση πραγματικά ε, το πόσο αποξενωμένη είναι η συζήτηση εδώ στη συζήτηση, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Αποξενωμένη, θα τα αντιμετωπίσουμε. Το Σέγγεν έχει πεθάνει. Δεν υπάρχει καμία υποστήριξη από την κοινή γνώμη. Όπως και το αστείο σχέδιο να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία. Μια χώρα με μια καλή σχέση εκκλησίας και κράτους σιγά σιγά ξεγλιστράει και γίνεται Ισλαμικό κράτος με πολύ αμφιλεγόμενο ρόλο σε θέματα ίσης, ε, Κούρδων η Τουρκία που μας εκβιάζει με τη ροή ε, παράνομων προς την Ευρώπη. Αυτό αρκεί ως ε, λόγος θεωρώ για να μπει στα σκουπίδια αυτό το ανόητο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί το να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα κράτος που είναι όλο και πιο Ισλαμικό ουσιαστικά είναι ό,τι πιο ανόητο μπορούμε να κάνουμε. Ε, ε, κυρία Βίμπερ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρία δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό θα πάρει η Τουρκία για να χρηματοδοτήσει την υποδοχή των μεταναστών. Την τελευταία φορά που άκουσα να μιλάμε για τέτοια ποσά, μιλήσαμε για 5 δισεκατομμύρια. Αλλά πώ θα καταφέρουν να βρουν τα χρήματα αυτά, το τεράστιο αυτό ποσό τα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταφέρει να πληρώσει αυτό θα σήμαινε ότι η χώρα μου, η Σουηδία, που έχει ήδη υποδεχτεί περίπου 200.000 από άσυλο το τελευταίο χρόνο, θα χρειαστεί να δανειστεί για να δώσει τα χρήματα αυτά, για να πληρώσει πέρα από τους ε, πρόσφυγες που έχει ήδη φιλοξενήσει μία χώρα ε, όπως η Τουρκία, διέλευση των μεταναστών, η οποία θέλει να συνεχίσει να παίζει το ρόλο που παίζει με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συνεχίσει να ασκεί πίεση στην Μεσόγειο. Βλέπετε τι συνέβη τον Ιανουάριο. 30 φορές πιο πολλοί μετανάστες ε, ε, ήλθαν από την Τουρκία σε σχέση με το περασμένο έτος. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος, ο κ. Στούγκε. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Βίμπεργκ το εξής. Για αυτήν δεν είναι σουρεαλιστικό να βρίσκεται σε μια συζήτηση όπου μιλάμε για τη βία κατά των προσφύγων, κατά των των άσυλων. ενώ στη χώρα της έχουμε χιλιάδες περιστατικά σε κέντρα υποδοχής προσφύγων και ε, ασκείται βία κατά των ε, ανθρώπων που εθελοντικά δουλεύουν και μάλιστα είχαμε και μία νεκρή πρόσφατα. Πώς κάνουμε τη συζήτηση αυτή εδώ, ενώ αυτά γίνονται στη χώρα σας, την ίδια. Όντως, είναι εξαιρετικά περίεργο και ήθελα απλά να σας πω ότι καταδικάζω οποιαδήποτε μορφή ρατσισμού και βίας. Και όντως, ε, πριν από δύο εβδομάδες, μία νεαρή γυναίκα δολοφονήθηκε από έναν ανήλικο ασυνόδευτο. αναφέρθηκε ότι το προσωπικό κρύφτηκε και δεν ε, σηκώθηκε γιατί ε, φοβήθηκε τον ε, ασυνόδευτο αυτόν υλικό. Και αυτό είναι ενδεικτικό του φόβου που επικρατεί. Αυτοί οι, οι, νέες, για παράδειγμα, έχουν πλέον δισταγμού και φοβούνται να πάνε στις πισίνες, για παράδειγμα. Και είστε δίκαιο, είναι παράλογη αυτή η κατάσταση. Κύριε Σπόχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Γιατί δεν ε, παραδεχόμαστε ότι δεν λειτουργούν τα hot δεν ε, λειτουργεί η επιστροφή, η προστασία των εκτορικών σύνορων δεν λειτουργεί, το Δουβλίνο δεν λειτουργεί, η επιστροφή των προστίγων στην Τουρκία δεν λειτουργεί, η εκπαίδευση στην Τουρκία δεν λειτουργεί, η κοινή μεταναστευτική πολιτική και πολιτική ασύλου δεν λειτουργεί και από την αριστερή πλευρά του πολιτικού φάσματος μας μιλούν για την τήρηση των ε, αρχών, των πολιτικών αρχών. Πού είναι όμως οι απαιτήσει και οι αξιώσεις έναντι των έτων των άσυλων και των προσφύγων. Αυτοί μπορούν να κάνουν τι θέλουν. Ε, απειλούν, βιάζουν, δολοφονούν και αν δεν τηρούν τις αρχές μας, δεν μπορούν να μπουν σε ρυθμό ενσωμάτωσης. Δεν μπορούν να μείνουν στην Ευρώπη. Πρέπει να φύγουν από εκεί που ήλθαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Όλμπριχτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε και κύριοι. Ο τρόπος με τον οποίο χειριζόμαστε την κρίση αυτή θα έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία μας στο μέλλον και στο λόγο ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντικά χαρακτηριστικά της αποτελεσματικότητάς μας είναι η δυνατότητα να αξιοποιούμε διαφορετικά μέτρα, αλλά και πόρους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει με προσοχή ένα μηχανισμό στήριξης της Τουρκίας. Και έτσι θα ήθελα να ρωτήσω την Προεδρία. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό το μηχανισμό και πώς θα συμβάλλουν τα κράτη-μέλη σε αυτό το μηχανισμό αυτό. Πώς θα επηρεάσει αυτός ο μηχανισμός ε, την ακαιρεότητα του προπολογισμού. Χρειαζόμαστε επιπρόσθετα μέσα συμμετείχαμε σε μια διάσκεψη επί του προπολογισμού και νομίζω ότι υπό αυτό το φω θα πρέπει να σκεφτούμε και να βρούμε νέα μέσα που θα αλλάξουν τον τρόπο λειτουργία ε, του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Θα πρέπει να το σκεφτούμε τώρα αυτό γιατί στο μέλλον θα βρεθούμε αντιμέτωποι με αντίστοιχε καταστάσει και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για πολύ σύνθετε καταστάσει. Τι συμβαίνει λοιπόν με τον μηχανισμό υποστήριξη τη Τουρκία, Έχετε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Έθριτζ. Ευχαριστώ. Αναφερθήκατε στις πληρωμές ε, προς ε, την Τουρκία. Δεν συμφωνείτε μαζί μου ότι η κατάσταση στην Τουρκία είναι μια ένδειξη αδυναμίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανικανότητα να αντιμετωπίσει την ε, μεταναστευτική κρίση. Μας κοροϊδεύει η Τουρκία, παίζει μαζί μας και ουσιαστικά μας εκβιάζει και εμεί μάλλον λαδώνουμε τόσο ρογικών ε, την Τουρκία για να κάνει αυτά που θα πρέπει να κάνει έτσι κι αλλιώ. Το ερώτημά σας έχει και μία κατηγορία. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να κατανοήσουμε ποιο είναι το κίνητρο. Είναι σαφές όμως ότι εκμεταλλεύεται την κατάσταση η Τουρκία για να επιτύχει τους σκοπούς της. Συμφωνώ. Όμως για μα το πιο σημαντικό είναι τα δικά μας ε, συμφέροντα και τα συμφέροντα των πολιτών μας. Επομένω, το θέμα είναι αν θα υπάρξει ένα δίκαιο, διαφανή και αποτελεσματικό μηχανισμό. Συμφωνώ ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και βέβαια ε, αυτό έχει σχέση και με τα τουρκικά συμφέροντα. Για 1,5 λεπτό, Νέντρ Μίλλερ. Ευχαριστώ. Η συμφωνία, η συνθήκη του Σέγγεν Εκφράζουμε το βέλτιστο δυνατό τρόπο το γεγονός ότι η Ευρώπη αποποιείται τους εγωισμούς. Πρόκειται για μια Ευρώπη όχι των συνόρων, αλλά μια Ευρώπη η οποία συνδέεται και συνενώνεται από την ελευθερία. Και τώρα λοιπόν απειλείται το Σέγγεν. Το θέμα δεν είναι οι πρόσφυγες. Το θέμα είναι ότι ο εθνικισμός διευρύνεται στην Ευρώπη. Και όσοι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθούν τόσο πολύ τα εθνικά αυτά σχέδια, θέλουν να κάνουμε ένα βήμα πίσω στην ιστορία μας. Δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε αυτό. Δεν μπορούμε να μας επιβάλλουν αυτά τα κόμματα την ε, θέλησή τους. Δεν μπορούμε να μας ε, κρατούν, ε, δεν επιτρέπουμε να μας κρατούν ομήρους σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής. Χρειαζόμαστε λοιπόν άλλα μέτρα, όχι φράχτες, ευρωπαϊκή συνεργασία. Και φυσικά η ασφάλεια του πολίτη αποτελεί πρώτη προτεραιότητα, αλλά δεν μπορούμε να θυσιάσουμε στο βωμό αυτή στην ελευθερία μας. Η επαναφορά των συνόρων και η κατάργηση του Σένιεν θα ήταν το τέλος αυτό των ευρωπαϊκών ιδεών. Κάποιες κυβερνήσεις στην Ευρώπη ενδεχομένω να χαίρονταν, αλλά δεν θα τους δώσουμε την ικανοποίηση αυτή. Η Ευρώπη αποτελεί βάση για την ελευθερία, όχι τέτοιο ζήτημα για κάποιε κυβερνήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μακοβέη. Δύο εκατομμύρια πρόσφυγες έχει η Τουρκία και πρέπει να υποστηριχθεί στα πλαίσια της διαχείρισής τους. Τα τρία δις ε, τα οποία προβλέπονται ε, προβλέπουν ταυτόχρονα εθνικές συνεισφορές από τις διάφορες χώρες. Είναι ένας καλός μηχανισμός γιατί στην παρούσα φάση η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η βασική δωρήτρια για τη διαχείριση της χρήσης. Χρηματοδότρια καλύτερα. Ταυτόχρονα η κρίση από ό,τι φαίνεται τους επόμενους μήνες θα χειροτερεύσει. Υπάρχουν πάρα πολλές συγκρούσεις που προκαλούν τις ροές της προσφυγικές και μόνο συλλογικά πρέπει να αντιμετωπιστούν και γι' αυτό η συνεργασία με την Τουρκία είναι απαραίτητη. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω κάτι και για το θέμα της ε, ανοχής. Όταν ε, μια κοινωνία η οποία έχει την έννοια της ανοχής στο εσωτερικό της ε, δέχεται μια άλλη κοινωνία που δεν την έχει τότε κινδυνεύει να καταστραφεί. Μπλε κάρτα. Ευχαριστώ την κυρία Μακοβέη, λέει ο κύριος Γιάνκοβιτς για την ε, μπλε κάρτα που δέχτηκε. Σας άκουσα προσεκτικά όταν αναφερθήκατε στην ανάγκη να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε την ε, Τουρκία. Ενώ σήμερα ο βασιλεύς ε, Αμπτουλά δήλωσε ότι η Ιορδανία που έχει υποδεχθεί ένα εκατομμύριο μέχρι τώρα δεν μπορεί να υποδεχθεί άλλους. Ένα εκατομμύριο διακόσες χιλιάδες έχει δεχθεί μέχρι τώρα. Μήπως πρέπει να μιλήσουμε και για την χώρα αυτή ε, και να βοηθήσουμε τα Ηνωμένα Έθνη να ελέγξει κάπως την κατάσταση επί τόπου. Μία τεχνική ερώτηση έχω να κάνω για την Προεδρία σας, την οποία πραγματικά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλή, αλλά έχω προβλήματα γιατί εγώ ε, επανειλημμένα ζητώ μπλε κάρτα και οι υπάλληλοι κοιτούν μπροστά. Πώ να του ενημερώσω, να χτυπήσω το τραπέζι, να χτυπήσω παλαμάκια. Σα παρακαλώ, βοηθήστε με, γιατί θέλω να τραβήξω την προσοχή του και θέλω κι εγώ να μου δίνετε μπλε κάρτε. Ε, ε, συνάδελφοι, είστε. Οι συνάδελφοι ενδεχομένω να μην σα πρόσεξαν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Τώρα όμω που ε, μας είπατε ότι θέλετε να θέσετε μπλε κάρτα, θα σας προσέχουμε όλους ιδιαίτερους και πολύ ζητούμε συγγνώμη αν δεν σας προσέξαμε. Άλλη μια μπλε κάρτα όμως για την κυρία Μακοβέη. Ο κύριος Φουντούλης. Ε, ε κύριε Πρόεδρε, ε, δεν θέλω μπλε κάρτα, αλλά θέλω να επισημάνω κάτι που ίσως διέφυγε της προσοχής σας. Προηγμένως η συνάδελφος Γκούσμαν μίλησε στο κοινοβούλιο και φερούσε μία μπλούζα η οποία έγραφε πάνω antifascist action και έχει μπει στο twitter και σε όλα τα μέσα δικτύωσης. αυτό νομίζω απαγορεύεται από το κοινοβούλιο γιατί μπορούσα και εγώ να φορέσω μία μπλούζα του λαϊκού συνδέσμου χρυσή αυγή και να είμαι εδώ όμως βλέπετε δεν το κάνω. πρέπει να επισημανθεί και να της γίνει παρατήρηση. Ε, Σημειώνω το ζήτημα που αναφέρεται, όμως τώρα πρέπει να δώσουμε το λόγο στην κυρία Μακοβέ για να απαντήσει. Και μετά θα το συζητήσουμε. Τέλος πάντων, ε, το σημειώνω. Ευχαριστώ. Είναι πολύ απλή απάντηση. Πρέπει να συνεργαστούμε με όλες τις χώρες που έχουν υποδεχθεί πρόσφυγες και ε, να προσδιορίσουμε και τα κοινά μας συμφέροντα, που είναι να μην υποδεχθούμε τους πάντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με κάποιον τρόπο να καταφέρουμε ε, να τους μοιράσουμε, κάποιους να τους στείλουμε και στις αραβικές χώρες, εκεί που θα είναι ασφαλής Η κυρία Χιούσμε τώρα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και η διάσκεψη της ε, Γενέβης του 51 προβλέπει ότι όταν κάποιος ε, παράνομα έχει διέλθει τα σύνορα, απευθεία θα πρέπει να εμφανιστεί ενώπιον των αρμοδίων αρχών. Ε, Δυστυχώ, οι πρόσφυγε πολύ συχνά ε, δεν κάνουν αυτό. Κρύβονται και έτσι κινδυνεύει η ζωή του, γιατί γνωρίζουν ότι οι διαδικασίε για τους πρόσφυγε πρέπει να ολοκληρωθούν στην πρώτη χώρα εισόδου. Αυτό θέλουν να αποφύγουν. Δεν θέλουν η διαδικασία να γίνει στην πρώτη χώρα εισόδου. Από την άλλη, τα κράτη-μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετωπίζουν αυτή την τεράστια πρόκληση. Ε, πρέπει να φιλτράρουν τους πρόσφυγες. Όταν οι αιτούντες άσυλο επιλέγουν τις επικίνδυνες οδούς μέσα στη νύχτα αντί να προχωρήσουν στις νόμιμες οδούς, είναι δύσκολο να μην μιλήσουμε για ε, την αρχή της μη επαναπρόθεσης. Τα συστήματα μας δεν είναι παρκή. Εάν δεν έχουμε ένα κοινό σύστημα υποδοχής βάσει ενός δίκαιου συστήματος για καθεστώτος μετεγκατάστασης, θα έχουμε τέτοια φαινόμενα και στο μέλλον. Ευχαριστώ κύριο Χατζηγεωργίου για ένα λεπτό. Οι συνάδελφοι, νομίζω ότι είμαστε τραγικοί. Είμαστε τραγικοί γιατί επαναλαμβάνουμε μια συζήτηση κάθε μήνα χωρίς ουσιαστικά να υπάρχουν προτάσεις, προτάσεις από πουθενά. Δεν υπάρχουν προτάσεις από το Κοινοβούλιο, από την Επιτροπή, δεν υπάρχουν προτάσει από τα Ηνωμένα Έθνη. Υπάρχει όμω μια βασική διαφορά αυτή τη συζήτηση από τι προηγούμενε. Στι προηγούμενε λέγαμε έρχεται χειμώνα. Τώρα λέμε ότι έρχεται άνοιξη. Υπάρχει ακόμα μια βασική διαφορά. Έχουν προσθεθεί μερικοντάδε νεκροί. Η Τουρκία έχει δεχτεί μεγάλο βάρο, αλλά ποιο ελέγχει τα λεφτά αν πηγαίνουν πράγματι για τον λόγο που δίνονται. Δέστε το Λίβανο, έχει δεχτεί 20% του πληθυσμού του είναι πρόσφυγε αυτοί οι αριθμοί για τους οποίους εμείς αναφερόμαστε είναι το 0,1 του πληθυσμού της Ευρώπης. Οι φράχτες, αγαπητοί συνάδελφοι, τι ρόλο παίζουν. Οι φράχτες οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Ποιοι δίνουν τα όπλα στις εμπόλεμους ε, στη Συρία. Γιατί δεν το καταγγέλει κανείς αυτό. Στην προηγούμενη συζήτηση είχα πει ότι αν ήμουν πρόσφυγας και άκουγα αυτή τη συζήτηση θα έβρισκα τρόπο να πάω να πνιγώ νομίζω ότι μας έχουν ακούσει οι άνθρωποι και αυτό ακριβώς είναι που κάνουν. κλείνω με μια, διατύπωση δεν έχω ακούσει πρόταση ούτε από την επιτροπή και διαρωτούμε τι πραγματικά σκέφτονται σήμερα μετά από δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και μετά από δέκα χιλιάδες... Διακόπτε πρόεδρε. Ούρτασουν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Επιτροπής θα ήθελα να νιώσω μια κάποια δυστημία για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ευρώπη. Φοβάμαι ότι δεν βλέπουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Είναι, είμαι ιδιαίτερα ανήσυχος και από τα στοιχεία τα οποία έχει δημοσιεύσει η Europol όπως επίσης και από τους αριθμούς των νεκρών στην Μεσόγειο. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση που συμβαίνει στην Ευρώπη που ισχύει στην Ευρώπη έχουν παραλύσει τα ευρωπαϊκά όργανα. Καμία χώρα δεν σέβεται πλήρως το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Το μόνο το οποίο ζητώ λοιπόν από εδώ είναι τουλάχιστον ας αντιδράσουμε σαν άνθρωποι. Ας σεβαστούμε τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και δεν ξέρω τι συμβαίνει στην Πολωνία ή στη Δανία. Νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά και η Ισπανία μέχρι τώρα έχει δεχτεί 18 πραγματικά πρόσφυγες. Είναι ντροπή τώρα αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτο. Ας σεβαστούμε τουλάχιστον τις υπογραφές μας πριν δύο μήνες. James, δύο λεπτά. E ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο και η πρόσβαση στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής είναι μια φιλοδοξία για ε, εκατομμύρια ανθρώπου σε όλο τον κόσμο που βλέπουν ότι θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι του για να πετύχουν αυτό το στόχο. Όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Η Μέρκελ και η Γερμανία έχει ξεκινήσει μία διαδικασία που απειλεί τα κρατημέλη, τη συνοχή και την οικονομική ευημερία. Η Σένγκερ και η Frontex προφανώς δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτές τις τεράστιες μεταναστικές πιέσεις δεν αντιδρά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οποιαδήποτε ανταπόκριση βλέπουμε ότι δεν λειτουργεί. Το βλέπουμε σε όλε τι περιστάσει, όποτε το συζητούμε εδώ στην Ολομέλεια. Απαιτείται λοιπόν επανεξέταση και λήψη σκληρών αποφάσεων. Η άμεση προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να βγάλουμε το καρότο από τη μέση. Και μετά δεν χρειαζόμαστε και το μαστίγιο. Όμω πρέπει να σταματήσουμε τη ροή και τα προβλήματα που τη συνοδεύουν. 27 κράτη-μέλη δεν πρέπει να επομιστούν τις συνέπειες ε, ε, της ε, προσέγγισης ενός άλλου κρατούς μέλους, της Γερμανίας, που έχει μια λανθασμένη ιδεολογία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Ζήλιστρα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ο Υπουργό Κούντερ είπε στην αρχή τη συζήτηση ότι το πόσο εξετάζουμε και μεταχειριζόμαστε του μετανάστε αντικατοπτρίζει το ποιοι είμαστε. Όμω, λέμε επίση ότι ο τρόπο με τον οποίο εκείνοι οι μετανάστε ε, ε, μεταχειρίζονται τι γυναίκε μα και τα παιδιά μα δείχνουν και ποιοι είναι εκείνοι και στο ε, καταπλησμό προσφύγων στο Αλμύρι υπήρξε αντίστοιχο περιστατικό με μαχαίρωμα. Τι συμβαίνει λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν απελάσσονται απευθεία. Πρόεδρε, Έχουμε εκατομμύρια τέτοιου ε, τυχοδιώκτε και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει 3 εκατομμύρια για να σταματήσει αυτή, 3 για να σταματήσει αυτή η διαδικασία. Όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχώ εκβιάζεται, δίνει ε, χρήματα, αλλά έτσι δεν μπορούμε να αγοράσουμε την ασφάλειά μας. Ούτε σεντ δεν πρέπει να δώσουμε στην Τουρκία, γιατί το μόνο που θα μας δώσει σε επιστροφή είναι η μιζέρια. Ο εκβιασμό δεν είναι ε, η λύση, είναι τμήμα του προβλήματος. Ευχαριστώ. Λέναρς, για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι απαράδεκτη. Επίτροπε Αβραμόπουλε, σήμερα μιλήσατε για στατιστικά στοιχεία ε, με τα οποία τονίσατε ακριβώ αυτή την κατάσταση και δικαίω. Ο συνάδελφό σα, κύριο Τίμερμαν, δυστυχώ δεν είναι εδώ μαζί μα, επίση ε, ε, χειρίζεται τέτοια στατιστικά στοιχεία και είπε την περασμένη εβδομάδα ότι το 60% των ετούντων άσυλων στην Ευρώπη δεν είναι πρόσφυγε. Δεν μπορούν να λάβουν τέτοιο καθεστώ πρόσφυγα και πρόκειται κυρίως για άτομα από την Βόρεια Αφρική. Από τα στοιχεία του Frontex προκύπτει ότι 89 με 97% των ατόμων που ε, εισήλθαν στην Ευρώπη προέρχονται από Συρία, Ιράκ ή Αφγανιστάν. Είτε η Frontex λοιπόν κάνει λάθο, είτε ο πρώτο αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ξέρει τη διαφορά μεταξύ Μαρουκινού και Αφγανού. Όμω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και στι δύο περιπτώσει εκτίθεται. Γι' αυτό εσεί τουλάχιστον θα πρέπει να δώσετε κάποια σαφήνεια, γιατί η σαφήνεια είναι απαραίτητη και κρίσιμη σημασία. Και ένα ερώτημα προ τον κύριο Κούντερ. Ε, για τα σχέδια του, ε, του ηγέτου του κόμματός του, κυρίου Σάμσον. Δεν πρέπει να υπάρξει παράνοια για τις θέσεις ε, της Ολλανδικής Προεδρίας. Πραγματικά θα ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα η Ολλανδική Προεδρία ή εδώ πέρα πρέπει να θεωρήσουμε ότι ε, είναι μάλλον κάτι, μια κίνηση εντυπωσιασμού για τον τύπο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μωράς για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλοί βουλευτές αναφέρθηκαν στην έκθεση της Europol, όπου αναφέρεται ότι 10.000 ασυνόδευτοί ανήλικοι είναι πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη χάνουν εκμετάλλευση. Συνάδελφοι, η Europol είναι από τις πιο αξιόπιστες ε, υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρουμε ότι αυτό είναι στιγμιότυπο μόνο. Ποτέ δεν υπήρξε μεταναστευτική κρίση τόσο, με τόσο συστηματική και ε, μεγάλη παραβίαση των δικαιωμάτων των ανελίκων και θα δείτε τους επόμενους μήνες να ανακύπτουν ε, ιστορίες φρίκης για την εκμετάλλευση αυτή. Αυτό το λέμε για όλους όσους ε, θεωρούν ότι έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε πίσω από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την ανάληψη δράσεων. Αν πιστεύετε ότι έχουμε την πολυτέλεια αυτή, να καταλάβετε ότι τις επόμενες εβδομάδες οι ανήλικοι αυτοί που είναι πραγματικοί ετούντες άσυλο που έρχονται από, το, από τη Συρία και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία βάσει της συνθήκης της Ζενέβης. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε δουλειά να κάνουμε στο Κοινοβούλιο για το Δουβλίνο, για τα σύνορα, προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους οι υπεύθυνοι. Αλλά ας ξανακάνουμε αυτή την έκκληση, τη βρετή έκκληση προς την Ολλανδική Προεδρία για τα κρατη που δεν κάνουν τη δουλειά τους, δεν προστατεύουν τα εξωτερικά του σύνορα, δεν ε, κάνουν ανακατανομή. Ας επαναλάβουμε το μήνυμα αυτό. Τα κράτη-μέλη που δεν κάνουν τη δουλειά τους να αναλάβουν τις ευθύνες τους να μην αλληγορήσουν Τώρα. Ευχαριστώ. Μπλε κάρτα. Από την κυρία Μουσολίνη την αποδέχεστε. Έχει δίκιο ο πρόεδρος Μωράες. Νομίζω ότι εδώ και τρία χρόνια είχαμε εγκρίνει στην Ιταλική Βουλή του να δοθεί ένα νομικό καθεστώς ειδικό στους ανηλίκους, χωρίς να περνούν από τις κανονικές διαδικασίες για το άσυλο. Έτσι μόνο θα προστατευθούν και έτσι θα γλιτώσουν από τα νύχια της αγκληματικότητας. Θα ήθελα τη γνώμη του Πρόεδρου μας. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ποτέ δεν μου κάνουν ερωτήσεις με μπλε κάρτα γιατί είναι βαρετές μάλλον οι μιλίες μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Μουσολίνη, η Ιταλία ήταν μία από αυτές τις χώρες στην εμπροστοφυλακία. Η Ιταλία, η Ελλάδα, ενώ χώρε, η Σουηδία και η Γερμανία παίρνουν πιο πολλού ε, μεταναστέ από κάθε άλλη. Το θέμα δεν είναι να επιτρέψουμε ευθύνε. Το θέμα είναι ότι η Ιταλία, επειδή είναι μπροστά-μπροστά, και έχει τις πολιτικές που έχει. Συμφωνώ με αυτά που λέτε, αλλά προς τους συναδέλφους εκείνους που δεν θέλουν να αναλάβουν πιο πολλούς μετανάστες, θα ήθελα να πω το εξής, ότι αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η, η Ορδανία και το πόσο κοντά είναι, ε, τα άτομα αυτά θα είχαν έλθει στην Ευρώπη και θα είχε τα θέματα αυτά η Ιταλία, ακριβώς επειδή είναι στην εμπροστοφυλακή. Συμφωνώ λοιπόν ότι θα πρέπει να βρούμε όλοι μαζί μία λύση. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό κύριε Στάνοκ. Πρόεδρε, η τρέχουσα μεταναστευτική κρίση καταδεικνύει ότι η συνθήκη της Γενέβης του 59 και το πρωτόκολλο του 57 δεν ταιριάζουν στον κόσμο των παγκόσμιων ταξιδιών και της μαζικής επικοινωνίας. Μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βασιστήκαμε τις ρυθμίσεις για τα άτομα που από... αντιμετωπίζουν πραγματική δίωξη. Δεν είχαν σχεδιαστεί αυτά για χώρες που ταξιδεύουν μέσω διάφορων χωρών για να καταλήξουν σε μια χώρα που έχουν ένα εύρωστο σύστημα πρόνοιας. Ούτε έχει σχεδιαστεί για να μπορεί να μεταφέρει το καθεστώς του ένα άτομο ως πρόσφυγας από χώρα σε χώρα, όπως γίνεται σε πολλές περιπτώσεις από την Τουρκία στην Ευρώπη. Το 2016 θα έχουμε νέο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, κατά πάσα πιθανότητα από την Ανατολική Ασία. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσει λοιπόν επί την ευκαιρία αυτή μεταρρύθμιση, αναθεώρηση τη συνθήκη του 51 για να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη όλες αυτέ τις εξελίξεις. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρούις, για μισή λεπτό. Ε, ναι, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ για τα μέλη και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αντιστέκονται σε αυτήν την τόσο μακρά συζήτηση. Εμείς μιλήσαμε για αξίες ε, και με τον κύριο Πιτέλα και με την κυρία Φεράρα είπαν για τις αξίες, αλλά οι αξίες επιβεβαιώνονται όχι με τα λόγια, αλλά με τις πράξεις, με συγκεκριμένες ενέργειες. Πολλές από τις χώρες όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδεικνύουν ότι δεν σέβονται τον, τον ανθρωπισμό που διέπει τις αξίες. Δυστυχώς ε, ε, δέχονται νοοτροπίες και εφαρμόζουν ενέργειες για τις οποίες αυτοί οι οποίοι έχουν διαπράξει εγκληματικές ενέργειες εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι ικανοποιημένοι. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε επίσης και σε σχέση με τους μη συνοδευόμενους ανηλίκους. Αυτό είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο. Έχουμε μια τεράστια αλυσίδα λαθών, μια τεράστια αλυσίδα αμελιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Πρέπει να δούμε τι ανθρωπιστικές ανάγκες υπάρχουν και ελείπει η κοινή πολιτική στον τομέα της χορήγησης του ασύλου. Αυτούς τους οποίους πρέπει να προστατεύσουμε, αυτούς τους ίδιους τους στιγματίζουμε. Νομίζω ότι υπάρχουν ΙΙ αυτή τη στιγμή που έχουν χτυπήσει τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Φορέντσα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την ευχή το ότι κάποιοι συνάδελφοι έβαλαν μια φανέλα που έλεγε αντιφασίστα είναι πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα αυτό όταν νέες μορφές φασισμού έχουν δείξει ότι αρχίζουν να έρχονται στην επικαιρότητα στην Ευρώπη και όταν βλέπουμε τους νεκρούς στη Μεσόγειο δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να είμαστε λοιπόν ειλικρινεί σε σχέση και με τα τρία δις τα οποία δώσαμε ή θέλουμε να δώσουμε στην Τουρκία, στην κυβέρνηση Ερντογάν, η οποία συνεχίζει να λειτουργεί εις βάρος του κουρδικού λαού. Εμείς δίνουμε υποτίθεται τα χρήματα αυτά για να εξωτερικοποιήσουμε το πρόβλημα, για να μπλοκάρουμε τους πρόσφυγες που είναι στην Τουρκία και να αποτρέψουμε την είσοδό τους στην Ευρώπη. Δώσαμε, λέει η ομιλήτρια, τρία δις σε μια κυβέρνηση η οποία έχει σχέσεις αμφιλεγόμενες με τον ΤΑΕΣ ε, για να υποδεχθεί καλύτερα τους πρόσφυγες. Εγώ θα πρότεινα τα τρία δις να τα δώσουμε στην αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών σε όλες τις ΜΚΟ που καθημερινά εργάζονται για την δημιουργία ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου. Ευχαριστώ κύριος Μαραγκάλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν με ικανοποιεί να γνωρίζω ε, ότι επανειλημμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Και δεν με ικανοποιεί το ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή μας ε, λέγουν ότι έχουμε δίκιο. Αυτό είναι άχρηστο, δεν οδηγεί πουθενά. Ε, έχουμε την υποχρέωση να φέρουμε εις πέρας ε, τις ανηλυμένες μας δεσμεύσεις και όχι να επιδεικνύουμε αδράνεια και έλλειψη ευθύνης. Το λέω αυτό και προς τον ε, κύριο Επίτροπο. Η συμφωνία με την Τουρκία είναι μια πάρα πολύ ανησυχητική βάση. Τρεις μήνες έχουμε καθυστερήσει για να το επιβεβαιώσουμε και δεν ξέρουμε πώς θα το εφαρμόσουμε. και δυστυχώς συνεχίζονται να πνίγονται οι αθώοι πρόσφυγες μπροστά στα μάτια των εθελοντών οι οποίοι προσπαθούν να τους φροντίσουν και να τους υποδεχθούν. Λοιπόν, πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες σε όλα τα κράτη-μέλη να τους κατανείμουμε σωστά και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Η Ευρώπη πληρώνει και θα πληρώσει ένα υψηλό τίμημα γιατί δεν λειτουργεί σαν Ευρώπη, δεν βοηθά σαν Ευρώπη. Ε, και νομίζω ότι όλοι μαζί ενωμένοι πρέπει να βοηθήσουμε και την ε, Ελλάδα και την Τουρκία. Χωρίς μικρόφωνο συνεχίζει ο κύριος Μαραγάλ, δεν ακούγεται. Δεν έχει μικρόφωνο πλέον ο κύριος Μαραγάλ. Κύριε Μαργάλ, υπάρχει μπλε κάρτα τον κύριο Ντέιος. Ε, τον κύριο Επιτίδιο, συγγνώμη. Θέλετε να το δεχτείτε, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Όμω η ερώτησή μου δεν είναι για τον κύριο Μαραγκάλ, είναι για την προηγουμένη ομιλήτρια, η οποία είπε ότι πρέπει να δίνουμε τα τρία δισεκατομμύρια στι ε, ΜΚΟ. Γνωρίζει ότι οι ΜΚΟ εμπλέκονται σε παράνομε ενέργειε πρόσφατα στην ελλάδα συνελήφθησαν μέλη των ΜΚΟ, τα οποία ήταν μέλη κυκλώματος προωθήσεως παρανόμων μεταναστών από την τουρκία προς την ελλάδα. σε αυτούς τους ανθρώπους θέλει να δώσουμε τα χρήματα; αυτές τις ενέργειες θέλει να επιβραβεύσουμε; ευχαριστώ. Ναι, το ερώτημα πρέπει να απευθυνθεί στην προηγούμενη μιλήτρια. Κυρία Φορέντσα, θέλετε να απαντήσετε. εκτός μικροφώνου. Ε, a rispondere, ma è ε, ε, rivolta la domanda ha fatto un po' di confusione forse. Έχει δημιουργηθεί μια μικρή σύγχυση. Δεν, εν πάση περιπτώσει, είναι για μένα η ερώτηση. Εγώ νομίζω ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με το ολοκαύτωμα αυτών των ανθρώπων, γυναικών και ανδρών και παιδιών. Νομίζω ότι θα πρέπει εμείς να χρηματοδοτήσουμε αυτούς οι οποίοι αναλαμβάνουν την ευθύνη και σαν πολιτική ένωση. Αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα σαν παράδειγμα Νομίζω ότι αυτά που συμβαίνουν δείχνουν την αδιαφορία και την έλλειψη πολιτισμού με την οποία η Ευρώπη υποδέχεται ε, τους ε, πρόσφυγες. Η κυρία Αρνοτού. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η ανεκανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει την μεγάλη μεταναστευτική κρίση που ε, στην Ευρώπη δείχνει ποιο θα είναι και το μέλλον της ε, Ευρώπης. Όμως ε, σήμερα το επίγον είναι να σταματήσουμε την μαζική εισρωή λαθρομεταναστών, ε, να αποκαταστήσουμε τον έλεγχο στα σύνορα για να σταματήσουμε και να επιστρέψουμε όλους αυτούς τους ετούντες άσυλο που δεν έγινε δεκτή η αίτησή τους και η ευρωπαϊκή νομοθεσία που ε, πρέπει να αλλάξει αυτή που δεν μας επιτρέπει να ε, τους επιστρέψουμε. Δεν πρέπει να δώσουμε ε, δισεκατομμύρια στην Τουρκία, αλλά να επανεξετάσουμε τις σχέσεις μας με αυτή την Τουρκία που στηρίζει τους τζιχαντιστές. Μιλήσατε για την ε, ρητορία μίσους κατά των ε, ε, προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη, ενώ γυναίκες στην Ευρώπη πέφτουν θύματα σεξουαλικής παρανόχλησης ή ακόμα και χριστιανοί πλήττονται και δέχονται επιθέσεις εξαιτία της θρησκείας τους. Είναι λοιπόν κάτι παραπάνω από μια ιδεολογική συζήτηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αγγέλη. Κυρία Πρόεδρε. Είμαι αρκετά ικανοποιημένος που βλέπω ότι έχει επανέλθει το Συμβούλιο γιατί βλέπω ότι για έκτη, 8 8η φορά που κάνουμε αυτή τη συζήτηση και θα ξανακάνουμε και άλλε 10 συζητήσεις κατά ψευθενότητα υπάρχει ε, μία συμφωνία, μία σύμπνοια απόψεων σε ό,τι φορά το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν. Το Συμβούλιο είναι αυτό που δεν θέλει και δεν είναι διατεθειμένο να αναλάβει δράση. Είτε αυτό αφορά την κοινή προστασία των εξωτερικών μα συνόρων, γιατί όλα τα εξωτερικά μα σύνορα είναι κοινά μα σύνορα, ανήκουν σε όλου και τα κρατημέλη είναι αυτά που θα πρέπει να τα ελέγξουν, είτε σε ό,τι αφορά την μεταγκατάσταση μεταναστών σε όλη την Ήπειρο όπου ορισμένε κυβερνήσει θεωρούν ότι αυτό δεν τι αφορά και έτσι και οι υπόλοιποι δεν μπορούν να αναλάβουν δράση, είτε αφορά το ζήτημα την Τουρκία ή οποιοδήποτε άλλον που δεν μπορούμε ε, να καθορίσουμε κατά πόσο τον προλογισμό έχουμε αρκετούς πόρους για να το αναλάβουμε. Μιλούμε για μεμονωμένες πληρωμές όπως μιλούμε για μεμονωμένες μεταγκαταστάσεις προσφύγων. Αυτό είναι ένα από τα κύρια ζητήματα σήμερα και στο πλαίσιο αυτού του ζητήματο ανέρχεται και ο λαϊκισμό. Κυρία Πρόεδρε, κλείνοντα, θα ήθελα να πω ότι μία από τι πολιτικέ ομάδε των συντηρητικών μεταρρυθμιστών αυτή τη στιγμή τυχαίνει να είναι αυτή η ομάδα και ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι του. Ένα ευρωβουλευτή τουλάχιστον αυτή τη ομάδα θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει άδεια να πυροβολούμε όσους βρίσκονται στους μετανάστες. Και μάλιστα αυτή η πολιτική ομάδα το περιθάλπει αυτή την, ε, αυτό το πολιτικό πρόσωπο. Δεν γίνεται να επιτρέψουμε τέτοιες ε, πολιτικές. Κύριε Βανιθιάνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ δεν είμαστε σε ένα θέατρο. δεν είναι απλά ένας χώρος στον οποίο κάθε τόσο εκφράζουμε εμεί οι βουλευτές την απελπισία μας ή τις διαμαρτυρίες μας και το Συμβούλιο που έρχεται εδώ και που αλλάζει η Προεδρία μας ακούει υπομονετικά να τελειώσει ο γύρος των ομιλιών των βουλευτών. Εδώ γράφουμε ιστορία, η ιστορία την ιστορία της πιο σκληρής ανεπάρκειας που έχει ποτέ χαρακτηρίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ είμαστε μια συνάντηση πολιτικών ανδρών και γυναικών υπεύθυνο που απαιτούμε από τις κυβερνήσεις μας, απαιτούμε από το Συμβούλιο, απαιτούμε από την Επιτροπή να ξεπεράσουν αυτήν την απάνθρωπη ανεπάρκειά τους. Μπορεί κανείς να είναι ανεπαρκή σε διάφορους τομείς, αλλά εδώ μιλάμε ε, για, ε, για τους ανθρώπους. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα τον τελευταία χρόνια είναι απαράδεκτο. Εκατοντάδες άνθρωποι πνίγονται ε, στην θάλασσα. Είναι ε, μια τραγωδία. Έχει μετατρέψει τη Μεσόγειο σε νεκροταφείο. Και είμαστε υπεύθυνοι κύριοι του Συμβουλίου, κύριοι της Επιτροπής. Εμείς έχουμε την υποχρέωση να απαιτήσουμε από τις κυβερνήσεις μας να πάρουν τα απαιτούμενα μέτρα, να βρουνε λύσεις. Υπάρχουν λύσεις, εφικτές λύσεις για να σωθούν οι ανθρώπινες ζωές. Είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστούν οι νομικές ρυθμίσεις που ισχύουν. Εδώ είμαστε κοινοβούλιο, δεν είμαστε θέατρο. Πρέπει να εισακουστούμε. Κύριε Βαλισιάνα, έχετε μπλε κάρτα από τον κύριο Φουντούλη. Θέλετε να την δεχτείτε. Κύριε Φουντούλη, έχετε λόγο. Κυρία συνάδελφε, κυρία Βαλεντσιάνο. είπατε προηγουμένω ότι έχει καταντήσει το Αιγαίο και η Μεσόγειο σε ένα απέραντο νεκροταφείο. Σα ερωτώ λοιπόν, ποιο σπρώχνει αυτού του ανθρώπου να μπουν σε κάραβα και να περάσουν τα νερά του Αιγαίου. Απαντώ εγώ για σας, η Τουρκία. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα και πρέπει να το παραδεχτείτε. Δεν είναι ερώτηση αυτό το οποίο μου κάνατε, είναι μια άποψη. Εγώ δεν μιλάω για υπευθύνου μόνο. Εγώ λέω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διευκολύνει κανένα νόμιμο τρόπο για να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι στα σύνορά μας. Και αυτοί οι άνθρωποι ξεφεύγουν από τον πόλεμο και προστατεύονται από τις διεθνείς συμβάσεις. Αλλά δεν τους δίνουμε νόμιμα μέσα. Τους στέλνουμε στα χέρια των εγκληματιών ή τους στέλνουμε στο βυθό των θαλασσών. Αυτή είναι η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν τους υποδεχόμαστε, δεν τους βοηθάμε σε επίπεδο ανθρωπιστικό. Μιλάμε τρομερά λάθη αυτά τα οποία κάνουμε, είναι απάνθρωπα λάθη. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όλοι συμφωνούμε ότι η ανεξέλεκτη εισρωή μεταναστών προς την Ευρώπη θα πρέπει να πάρει ένα τέρμα. Θα πρέπει να το βάλουμε ένα τέλος. Και επίσης τα εθνικά κράτη είναι αυτά που πρέπει να προστατέψουν τα σύνορά τους. Κάποια ε, μπορούν να το κάνουν, κάποια άλλα δεν είναι σε θέση να το πράξουν αυτό ακόμα. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουν να, κάτσει, να κάνουν κάτι ουσιαστικό θα έπρεπε να αλλάξουν τον προπολογισμό, να πάρουν κονδύλια από αλλού και να αφιερώσουν πολύ πιο πολλά κονδύλια για την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Άρα, η μοναδική λύση είναι να μείνουν αυτά στα χέρια των κρατών μελών, των εθνικών κρατών μελών. Να μην τους κατηγορούμε, να μην επιρρύπτουμε ευθύνες σε όσους αποφασίζουν να προστατέψουν τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσοι δεν μπορούν να το κάνουν, πολύ απλά δεν θα μπορούν να είναι μέλος του Σέγγεν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να ετοιμάσει κάποιους πιο απλούς κανόνες για την ε, ανοικοδόμηση κάποιων εσωτερικών συνόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Δεπχέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο τελών ε, καθήκοντα Προέδρου του Συμβουλίου είπε ότι απέναντι στην προσωπική κρίση θα πρέπει να βρούμε κοινέ και αποτελεσματικέ λύσει. Και έχει απόλυτο δίκιο και συμμερίζουμε αυτή τη θέση. Πρέπει όμω να δούμε κατάματα την ε, πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ούτε κοινή διαχείριση των ε, κοινών συνόρων και βλέπουμε ότι η άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα έρεται σε ολόνα και φαινόμενο αριθμό χωρών και πρέπει να σταματήσει. Το σχέδιο ε, κατανομής ε, των προσφύγων αυτή τη στιγμή είναι μία φαρσοκομωδία. Και με το πρώτο τσεκ αυτών των τριών δις, παρόλα αυτά η Τουρκία ούτε περιορίζει τις ε, ροές και μάλιστα αυτή η μαφία έχει γίνει μια πραγματική βιομηχανία. Πρέπει να σταματήσουμε να χορεύουμε το χορό της κοιλιάς μπροστά στον Ερντογάν και θα να η λειτουργία του ε, hot γιατί πρέπει να υπάρξουν κέντρα υποδοχή στα hot Η πολιτική επιστροφή είναι μια, μια παρέστηση και αυτή τη στιγμή θα πρέπει να το ε, διοργανώσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ε, μια ανάκαμψη ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή πλευρά και έχετε το μπαλάκι στο δικό σα γήπεδο. Κύριε Ντεπχέ, υπάρχει μπλε κάρτα για εσά από Βούζεμπεργκ. Θέλετε να απαντήσετε. Κυρία Βόζεμπεργκ, παρακαλώ ήθελα να σας ρωτήσω εκτός από την αναγκαιότητα των hot spots που αναφερθήκατε και συμφωνούμε συμφωνείτε ή όχι ότι θα έπρεπε να αποφασίσουμε και την σύσταση hot spots εκτός, χωρών, των κρατών μελών όπως καταγράφει στο ψήφισμά του το συμβούλιο της ευρώπης. ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Αρχικά θεωρώ ότι εάν υπάρξουν hot spot στην ε, επικράτειά μας, αυτό είναι για να επιτελέσουμε κάποιο σκοπό, όχι μόνο για την καταγραφή γραφειοκρατικά. Αν τον αφήσουμε να φύγει τον πρόσφυγα οπουδήποτε, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε το κύριο χαρακτηριστικό του προγράμματος της Κομισιόν, που είναι η μετακατάσταση. Και έτσι δεν έχει κανένα νόημα ε, αν απλώς γίνεται καταγραφή και μετά δεν γίνεται τίποτα άλλο. Πρώτη απέτηση λοιπόν είναι να κάνουμε πολύ σωστά και αποτελεσματικά αυτό που έχουμε δεσμευτεί να κάνουμε. Η κυρία Σακοράφα. Συνάδελφοι, αντιλαμβάνεστε φυσικά ότι συζητάμε επιπτωμάτων που ο αριθμό του μεγαλώνει καθημερινά και μιλάτε για καλύτερη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και προτείνετε κιόλα συνεργασία με την Τουρκία, η οποία αμφισβητεί ακριβώ αυτά τα σύνορα. Ξεκαθαρίστε λοιπόν, τι εννοείτε, δεχόμαστε επίθεση από στρατό, απελπισμένου και πεινασμένου, γυναίκε και παιδιά έχουμε απέναντί μα. Τι προτείνετε, ναρκοπαίδια τάφρους ελεύθερους σκοπευτές. και μην ακούσω πάλι για επαναπροωθήσεις για αναστολή σέγγεν και λοιπές μεγαλοστομίες. και επιτέλους σταματήστε να κρύβεστε πίσω από την ελλάδα τις φορτώνετε ευθύνες για άλοθη επειδή αρνείστε εσείς να αναλάβετε έστω και τις ελάχιστες δικές σας ευθύνες για πρόβλημα που δημιούργησε και η δική σας πολιτική και σήμερα δεν άκουσα καμία αυτοκριτική σε αυτή την αίθουσα. τι θέλετε λοιπόν τι απεξεργάζεστε, τι έχετε αποφασίσει να ξαναφτιάξετε στρατόπεδα συγκέντρωσης να γίνει η ελλάδα ο λίβανος της ευρώπης να ξαναγίνει η ευρώπη το εκολαπτήριο του ναζισμού και του φασισμού. η λύση είναι μία κύριοι συνάδελφοι και την έχω ξαναπεί πολλές φορές σε αυτή την αίθουσα πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα ασφαλείς δρόμοι για τους πρόσφυγες και κατά αναλογία φιλοξενία τους σε όλα τα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στην ε, συζήτηση για το προσφυγικό τα τελευταία χρόνια ακούμε από την αριστερά το μάντρα ότι ε, λέμε φρικτά ψέματα και ότι η Ευρώπη είναι κάστρο απόρθεντο. Αλλά δεν έχουμε προστασία των εξωτερικών μας σύνορων. Πάνω από ένα εκατομμύριο μετανάστες ε, φέτος. Με την Τουρκία θέλουμε να δώσουμε μία ε, μέθοδο περιορισμού αυτής της ροής. και γι' αυτό αφιερώνουμε κονδύλια. Πρόκειται όμω για παζάρια. Αυτή είναι η τιμή. Και πολύ φοβάμαι ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα, να συλλαμβάνει δημοσιογράφος και το καθεξή. και θα κορυδεύει την Ευρώπη. Δεν υπάρχει, δεν αποτελεί λύση η Τουρκία για να αντικαταστήσουμε τους ελέγχους των συνόρων μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Μωράνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σταματήστε αυτή την πολιτική των ποσοστώσεων. Είναι ένα μήνυμα που προκαλεί την παράνομη μετανάστευση. Εγώ πήγα στο Λίβανο και στην Ιορδανία. Είδα το μεγάλο πρόβλημα βλέπουν ε, στις ειδήσει ε, στις παλιές τους τηλεοράσεις ότι η Ευρώπη θα τους υποδεχθεί, θα τους φροντίσει, θα τους ε, φροντίσει την υγεία τους, θα τους θρέψει. Έχουν τεράστιες ψευδεστήσεις. Εκεί βρίσκεται η πηγή του προβλήματος. Είναι καταδικασμένοι σε δύσκολες συνθήκες ζωής και προτιμούν να διασχίσουν τη Μεσόγειο ακόμα και αν κινδυνεύσει η ζωή τους. Η πραγματικότητα δεν είναι το, το, δεν είναι η ελπίδα αυτή την οποία θέλετε εσείς ε, ε, να τους εμφυσίσετε. Η Ευρώπη δεν μπορεί πια να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Δυστυχώς ούτε η φωτογραφία του φτωχού μικρού ε, στην τουρκική ακτή δεν μπόρεσε να έχει αποτελέσματα. Δυστυχώς είμαστε ανίκανοι να προσφέρουμε την ασφάλεια στους λαούς μας και φυσικά να υποδεχθούμε τόσους πολλούς μετανάστες και τόσους πολλούς παράνομους που εκμεταλλεύονται το σύστημα ασύλου. Απειλείται το Σέγγεν, η ζούγκλα του Καλέ έχει γίνει η ντροπή της Γαλλίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι να εκριζώνει τους πληθυσμούς. Πρέπει η πολιτική μας να είναι σωστή απέναντι στο Λίβανο, την Ιορδανία και τις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις για να βοηθήσουν οι λαοί αυτοί να μείνουν στις χώρες τους. Σταματήστε να ευνοείτε μια πολιτική που τους, αστεθερο... τους αποσταθεροποιεί και τους ανησυχεί. Η κυρία Σίπελ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα πρέπει να σας πω με πάσα ειλικρίνεια ότι έχω μείνει άφωνη. Ε, πραγματικά ντρέπομαι, είμαι εντελώς απογοητευμένη και φρύτω από τη συζήτηση τη σημερινή εδώ στο Κοινοβούλιο. Λέμε ότι θαυμάσιο είναι ότι η Τουρκία μπορεί να φροντίσει 2 εκατομμύρια ε, μετανάστες, να τους δώσουμε και λίγα λεφτά. Μα πραγματικά πιστεύουμε ότι εμείς ως Ευρωπαίοι, ως Ευρωπαϊκή Ήπειρος, με 500 εκατομμύρια πολίτες, δεν είμαστε σε θέση να φροντίσουμε 2 και 3 εκατομμύρια μετανάστες, πρόσφυγες. Αυτό είναι το μήνυμα λοιπόν που ε, στέλνουμε. Είναι πραγματικά φρικτό το πώς μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν για να ξεφύγουν από τον πόλεμο, την πολιτική δίωξη, από τη φτώχεια και τους οποίους τους αντιμετωπίζουμε σαν ε, ε προϊόντα, σαν αγαθά που κάπου θα τοποθετούμε. Όπου και αν τα βάλουμε, ε, εν πάση περιπτώσει μας απασχολεί εμάς. Ο αριθμός των προσφύγων που έρχονται προς εμάς ε, δεν αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση. Το πρόβλημα έγκυται στο ότι εδώ και χρόνια δεν υπάρχει ευρωπαϊκή στρατηγική για την αντιμετώπιση των προσφύγων. Καταφθάνουν όπου καταφθάσουν, στην Ιταλία, στην Βουλγαρία, στην Ελλάδα και αναμένεται ότι θα μείνουν εκεί. Η Γερμανία διαμαρτύρεται και λέει ότι ένα εκατομμύριο μετανάστες εντάξει, αλλά φτάνει τώρα. Στην Ελλάδα τον τελευταίο ε, χρόνο 800.000 είναι οι πρόσφυγες που κατέφθασαν σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν θα έπρεπε να μείνουν όλοι στην Ελλάδα. Πώς θα γίνει αυτό. Δεν έχουμε προσφυγική κρίση, έχουμε ευρωπαϊκή κρίση ανευθυνότητας, ολιγορίας και είναι πραγματικά φρικτό το πόσο εύκολα κάνουμε πίσω και πόσο εύκολα θα μπορούσαμε να καταστρέψουμε την Ευρώπη που έχουμε χτίσει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σίπελ. Έχουμε μπλε κάρτα, έχετε από την κυρία Χόλμα, την δέχεστε. Όχι. Next speaker ο ο κύριος Βάγγελ. sorry, uh, uh, Mrs. Ashford. Συγγνώμη, ο κύριος Ashford. Πρόεδρε, άκουσα την σημερινή συζήτηση και θα πρότεινα συνάδελφοι ε, το εξής. Υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι με τις λέξεις που χρησιμοποιούμε και την ορολογία. Λέτε μετανάστες, μάλιστα για ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν από το πόλεμο και τη δίωξη. Δεν είναι μετανάστες, είναι πρόσφυγες. Άνθρωποι τους οποίους πρέπει, μπορούμε και οφείλουμε να προστατεύσουμε. Μιλούτε για μετανάστες για να περιγράψετε ανθρώπου από όλο τον κόσμο που έρχονται στην Ευρώπη αναζητώντα μια καλύτερη ζωή. Δεν είναι μετανάστε αυτοί οι άνθρωποι είναι οικονομικοί μετανάστες. Άνθρωποι που δεν έχουν ε, καμία αξίωση να ζήσουν εδώ ή κανένα νόμιμο δικαίωμα μάλλον. Και τέλος, ε, μιλούνται για μετανάστες ε, αναφερόμενοι και σε Ευρωπαίους που ζουν σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, που δεν είναι η χώρα ε, καταγωγής τους. Δεν είναι μετανάστες αυτοί, είναι Ευρωπαίοι πολίτες που ασκούν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας όπως ε, προβλέπεται και έχουν κάθε δικαίωμα να πράξουν. Αν δεν είμαστε πιο συγκεκριμένοι στην ορολογία μας, όχι μόνο δημιουργούμε σύγχυση και στην κοινή γνώμη, όμως κάποιες φορές ε, δημιουργούμε σύγχυση και σε εμάς τους ίδιους. Κύριος Βάγκαλ. Ευχαριστώ. Αξιότιμα ε, Πρόεδρε, αξιότιμα κύριε Πίτροπε, κύριε Υπουργέ δεν πρέπει να υποτιμούμε πόσο ενημερωμένοι είναι οι μετανάστες και πρόσφυγες ε, στην Ευρώπη. Ξέρουν ότι δεν είναι πλέον ευπρόσδεκτοι. Ξέρουν ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητούμε περισσότερο πώς θα τους ε, αποτρέψουμε να έρθουν, πώς θα τους επιστρέψουμε, δεν θα τους υποδεχθούμε. Απλώς είναι πάρα πολύ για να τους υποδεχθούμε όλους με ανοιχτέ αγκάλες στην Ευρώπη ε, με βάση και τις ε, αξίες τις οποίες ε, παραπέμπουμε συνήθως. Δεν σκεφτήκαμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη όταν συμμετείχαμε σε πολέμους που τους εκδίωξαν από τις αιστείες τους και τους έκαναν να ταπεινωθούν ερχόμενοι με τι οικογένειέ του στα σύνορά του και στου δρόμου μα. Δεν τα σκεφτήκαμε όλα αυτά όταν ε, προτιμήσαμε την βία υπέρ τη διπλωματία. Ακούσαμε πολλούς συναισθηματισμούς ε, σήμερα, αγανάκτηση. Ε, δεν θα συμμετάσχω σε αυτό, όμως αυτή τη στιγμή, όπως και είπατε εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Μογκερίνη, αλλά και εκπρόσωποι των κρατών μελών, θα πρέπει ε, να στηρίξουν την ειρηνευτική διαδικασία στη Συρία που είναι η μοναδική εγγύηση ε, για να ξαναβρούν τα σπίτια τους οι πρόσφυγες όταν έρθει αυτή η ώρα, όταν επιστρέψουν στη Συρία. Και θα πρέπει να βρεθεί και πολιτικός συμβασμός με τις χώρες από όπου έρχονται οι αιτούντες άσυλων. Γονζάλη Σπένια, ευχαριστώ πολύ. Αυτές τις μέρες, αυτό το καιρό θα πρέπει να θυμίσουμε την υπόθεση της Άννα Φράνκ που εάν είχε πάρει βίζα θα είχε μπορέσει να πάει να μεταναστεύσει στις Ηνωμένε Πολιτείες μαζί με την οικογένειά της. Ε, ε, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο σας θυμίζει κάτι η ιστορία με τους Ναζί. Ε, τώρα μέτρα όπως αυτά που εγκρίθηκαν στην Δανία και οι απειλές της Κομισιόν εναντίον της Ελλάδας είναι πραγματικά εξοργιστικές σε μια ένωση όπως η δική μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, παρολύσει ε, για τη Συρία, να κάνει μια αποτελεσματική πολιτική για την υποδοχή των προσφύγων τρίγωνο τόσο στην Τουρκία, το Λίβανο και την Ιορδανία, όσο και στην ίδια την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της να εγγυηθεί το δικαίωμα στο άσυλο και την κατάλληλη ένταξη των προσφύγων. Αυτό σημαίνει πόρους και αλλαγή πολιτικών προτεραιοτήτων. Σας ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Μπιτζότο. Α, υπάρχει μια γαλάζια... Α, διαδικαστικό, συγγνώμη. Μάλιστα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, λόγω των διάφορων επαναλήψεων θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην ακούμε συνεχώς κηρύγματα. Τρίτη φορά ακούμε κηρύγματα που περιγράφουν τραγικότατη την ε, ιστορία στα εξωτερικά σύνορα και προσπαθούν να τα δικαιολογήσουν τα πάντα με την περίοδο των Ναζί. Δύο φορές άκουσα σύγκριση το τι κάνουμε σήμερα με το ολοκαύτωμα. Πρόκειται για μια μοναδική περίπτωση το ολοκαύτωμα και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην κάνετε έτσι εύκολα αυτές τις συγκρίσεις. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπιτσότο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το 2015 ένα εκατομμύριο μετανάστες ε, έχουν συνταράξει την Ευρώπη. Η εισβολή συνεχίζει και θα συνεχιστεί. Τα ε, κράτη όπως η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν αφαιθεί μόνο τους να αντιμετωπίσουν αυτή την εισβολή και οι πολίτες μας έχουν αφαιθεί να αντιμετωπίσουν την μαζική αυτή μετανάστευση με την ανεξέλεγκτη αύξηση της βίας και της εγκληματικότητας της πόλης μας, με την ε, Ισλαμική τρομοκρατική τρέλα. Τα σύνορα της, της Ένωσης ε, είναι διαπερατά και η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη χωρίς τους σωστούς ελέγχους στη θάλασσα και στη στεριά, χωρίς σωστή πολιτική μετανάστευση και χωρίς υποχρεωτική καταγραφή των μεταναστών που ζουν στην πλάτη μας η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα επιβιώσει στις, ε, από τις κοινωνικές πιέσεις αυτής της επίγουσας μεταναστευτικής ροής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιμάται βαθύ ύπνο τα τελευταία χρόνια, ονειρεύεται μια ενωμένη και ισχυρή Ευρώπη, μα είναι ώρα να ξυπνήσουμε γιατί το όνειρο της, Ευρω... της Ενωμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μετατραπεί σε φιάλτη για τους πολίτες μας. Ε, Επόμενο ο ο κύριο Πέντε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ καταρχά θα ήθελα να χαιρετήσω αυτά που είπε τελευταία ομιλήτρια από του συντηρητικού, ότι δηλαδή θα πρέπει να ε, δίνουμε κάποιε αποχρώσει σε σχέση με του μετανάστε, πρόσφυγε και τι λέξει που χρησιμοποιούμε. Θα ήθελα να το επιστήσω την προσοχή στο γεγονό ότι ο πρώτο που καλλιεργεί αυτή τη σύγχυση είναι ο ε, Βρετανό Πρωθυπουργό David Cameron. Και γι' αυτό και έχουμε συχνά αυτό το πρόβλημα τώρα για να διαπραγματεύουμε πραγματευτούμε αυτή τη σχέση, σε σχέση με την Βρετανική πρόταση που είναι παράλογη. Είμαι ευτυχής που υπάρχουν ωστόσο συντηρητικοί που καταλαβαίνουν ποιο είναι η ουσία του προβλήματος. Κατά τα άλλα θα ήθελα να επιμείνω στην πτυχή των εξωτερικών υποθέσεων για το θέμα των προσφύγων και ιδιαίτερα στο γεγονός ότι πρέπει από τη στιγμή που θα ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις στη Γενέβη να προσπαθήσουμε να ασκήσουμε το κύρος μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση στις διαπραγματεύσεις. Ε, αποδυναμωνόμαστε σε αυτό το πλαίσιο, διότι είναι αλήθεια, πρέπει να το πούμε, δεν έχουμε ακούσει τις φωνές των Ιορδανών, των Συρίων, των Λιβανέζων που μας ε, μιλούσαν για τους πρόσφυγες και αυτούς που κάνει, και το τι κάνουν. Ε, αργήσαμε να αντιδράσουμε και αυτό θέλω να το πω γιατί ε, εδώ σε αυτή την αίθουσα έχουμε πολύ κόσμο που είναι τελείως ανεύθυνοι όταν πρόκειται για την Τουρκία για λόγους που έχουν να κάνουν με τα δικά τους κομματικά συμφέροντα είναι έτοιμοι να βάλουν την Τουρκία σε πολύ άσχημη θέση χωρίς να καταλαβαίνουν ότι χρειαζόμαστε αυτόν τον εταίρο για να λύσουμε το πρόβλημα των προσφύγων. Ευχαριστώ, κύριος Χάουιτ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πέρσι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποσχέθηκε να δώσει τρία δις στην, στην Τουρκία για να την βοηθήσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που έχει με τα 2,75 εκατομμύρια πρόσφυγες ε, που έχει. Το μέσον αυτό θα ήταν μια βοήθεια η οποία θα λειτουργούσε από πρώτης πρώτου και όμως ένα μήνα μετά ακόμα τα κράτη-μέλη της Ένωσης τσακών θα συνεισφέρουν. Η χώρα μου βεβαίως προσφέρθηκε να πληρώσει γρήγορα, αλλά απογοητεύτηκα ιδιαίτερα για το ότι δεν πήρε το μερίδιο που της αναλογούσε σε πρόσφυγες όσον αφορά την μετεκατάσταση. Μιλάμε για 0,5 δισεκατομμύριο το οποίο θα έπρεπε να δοθεί από τον κοινοτικό προπολογισμό και το υπόλοιπο από τα κράτη-μέλη και έχουμε φτάσει ήδη στο 1 δισεκατομμύριο από τον κοινοτικό προπολογισμό και δεν πρέπει να είναι άλλο. Ο πρόεδρος Γιούνκερ ε, είχε δίκιο όταν είπε ότι τα χρήματα αυτά είναι ζήτημα αξιοπιστίας και σήμερα όταν υπάρχουν κάποιοι και από τη δικιά μου τη χώρα που θέλουν να αποτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο τεστ αυτό της αξιοπιστίας πρέπει να φροντίσουμε να επιτύχει. Όπω τόνισε η πολιτική μου ομάδα, Όποια και αν είναι η κρίση, οι κοινέ μα αξίε πρέπει να παραμείνουν οι ίδιε. Και ζητάω από όλα τα μέλη να πάνε εδώ πέρα στι κυβερνήσει του και να του ζητήσουν να δώσουν τα χρήματα για να δοθεί ανθρωπιστική βοήθεια που τόσο απεγνωσμένα χρειάζεται. Σα ευχαριστώ, ο κύριο Τσαρνέτσκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, σέβομαι τους ε, προλαλήσαντες, αλλά εάν ρωτούσα εγώ πόσοι από εσά έχετε πάει σε στρατόπεδο προσφύγων, πώς θα σηκώναν το χέρι. Καλύτερα να μην ρωτήσω. Εγώ έχω πάει σε τέτοιο στρατόπεδο. Πέρασα έξι μέρες της άδειά μου εκεί πέρα, στο Κουρδιστάν. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν να πάνε, αρκετοί από αυτούς δεν θέλουν να πάνε στην Ευρώπη, αλλά πίσω στα σπίτια τους που τώρα βεβαίως τα ελέγχει το Ισλαμικό κράτος. Οπότε τα λεφτά δεν πρέπει να πάνε στην Τουρκία αλλά και στο Κουρδιστάν. Και τέλος, ας μην είμαστε υποκριτές. Μιλάμε για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Θυμάμαι τον πρόεδρο της Γαλλίας το Δεκέμβριο του 2007 ο οποίος είπε πως ε, το κλιματικό πακέτο ήταν ε, καλό για την παλιά Ευρώπη και όχι για ολόκληρη την Ευρώπη. Πού ήταν τότε η αλληλεγγύη. Πού είναι η αλληλεγγύη όταν η Γερμανία κάνει δικές συμφωνίες με τη Ρωσία. Σας ευχαριστώ. Κύριος Πέτερσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα διανύουμε μια περίοδο κρίσης αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γινόμαστε μάρτυρες αυτού του γεγονότος διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανίκανη να δράσει. Το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας, μία από τις βάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι κάτι που μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένο. Αποτύχαμε, εμείς οι πολιτικοί αποτύχαμε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα απότυχαν, δεν καταφέραμε να δώσουμε τις απαντήσεις που περίμεναν οι λαοί από εμάς. Και αυτό οφείλεται στην έλλειψη πολιτικής βούλησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το σημαντικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λύνονται τα προβλήματα. Αλλά δεν είναι ένα κουμπί το οποίο πατάει κανεί και ω διαμαγεία λύνεται το κάθε πρόβλημα. Εάν τα κράτη-μέλη δεν συμμετάσχουν, δεν συμβάλλουν στην κοινότητα, ε, τότε δεν έχουμε δεσμού, δεν υπάρχει αληθινή κοινότητα. Και αυτό το οποίο βιώνουμε αυτή τη στιγμή είναι το εξή. Όλε οι ευρωπαϊκέ κυβερνήσει μιλούν για κοινέ λύσει, αλλά πράττουν εξιδίων, ατομικά η καθεμία. Όλοι έχουμε ευθύνε, πρέπει να βρούμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα και πρέπει να καταλήξουμε σε κοινέ λύσεις, να τις διαμορφώσουμε μαζί. Πρέπει τα κράτη-μέλη να το κατανοήσουν αυτό και μια καλή ευκαιρία για να το συνειδητοποιήσουν όλοι αυτό είναι η επικείμενη σύνοδος κορυφής του Φεβρουαρίου. Καλό το Συμβούλιο να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις, το χρειαζόμαστε αυτό και όλοι γνωρίζουμε ότι για να καταλήξουμε σε κατάλληλες λύσεις πρέπει να μπορούμε να δράσουμε μαζί, από κοινού. Ο κύριος Χουαρίστια Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μετά από αρκετά χρόνια το Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι έλαβε τις κατάλληλες αποφάσεις και ότι τώρα έχει έρθει η ώρα τέλους για δράση. Η Επιτροπή υπονοεί και υπενήσεται ότι όσους περισσότερους εκδιώξουμε, τόσο περισσότερο ο κόσμος θα πιστέψει στο ευρωπαϊκό ε, κοινό άσυλο. Το ΕΛΚ περίπου τα ίδια και το Άλτε λέει ότι στις 18 Φεβρουαρίου είναι η σημαντική ημερομηνία. Χρειάστηκε χιλιάδες θάνατοι για να φτάσουν εκεί. Δείχνετε αλληλεγγύη από τη μία και τα κόμματά σας κάνουν το αντίθετο όταν είναι στην κυβέρνηση. Ε, για διαστροφικό παιχνίδι μίλησε μία Ιταλίδα συνάδελφος. Ένα μείγμα ανικανότητας, απουσία πολιτικής βούλησης. Ε, είναι θέατρο του παραλόγου, πιο παράλογο και από το θέατρο του Μπέκετ και των λοιπών. Πηγαίνετε στη Λέσβο, πηγαίνετε στη Θέουτα, στο Καλέ, να μάθετε ακριβώς τι συμβαίνει. Και η συζήτηση αυτή, αν πάτε, θα είναι τελείως διαφορετική. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέι, παρακαλώ. Προλίγο ακούσαμε τον πρόεδρο των σοσιαλιστών να λέει ότι το πρόβλημα της Ευρώπης ήταν ο ιός του φόβου έναντι της μεταναστευτικής καταστροφής και το, την ομιλία του αυτή τη χειροκρότησε ο πρόεδρος του ΕΛΚ εκπρόσωπος της κυρίας Μέρκελ. Ο κύριος Πιτέλε όμως καλό θα ήταν να έχει περισσότερη ψυχραιμία και να ε, υποδεχθεί στο σπίτι του τους πρόσφυγες όσους μπορεί. Υποτίθεται ότι υπερασπίζεστε μια κοινότητα αξιών. Οι αξίες σας όμως είναι αφηρημένες, αυθαίρετες και εξυπηρετούν ουτοπικές ιδεολογίες. Δεν είναι δικές μας οι αξίες αυτές. Εμείς έχουμε άλλες αξίες, άλλες αρχές. Εσείς θέλετε με κάθε τιμήμα να ε, βοηθήσετε τους παρανόμους σε βάρος των δικών μας Ευρωπαίων πολιτών. Δεν πληρώνετε όμως εσείς τις συνέπειες των τρελών σα αποφάσεων, αλλά είναι τα πιο ευπαθή τμήματα της ευρωπαϊκής κοινωνίας που υφίστανται αυτό το μεγάλο τίμημα. Οι, βιότι, οι βιαιότητες που διαπράττουν οι μετανάστες ε, στο ε, καλέ υπάρχουν, τις αρνείστε και δεν το κάνατε κατά λάθος. Πρόεδρε κυρίε και κύριοι συνάδελφοι σε ένα περιβάλλον απειλή κατά τη ζώνη σέγγεν οφείλουμε να είμαστε ειλικρινεί απέναντι στου εαυτού μα και τους πολίτε μα το κλείσιμο των συνόρων είναι πολιτική επιλογή όχι αναγκαιότητα επιλογή συγκεκριμένων κρατών που δεν θέλουν τους πρόσφυγες στο έδαφος τους αδιαφορούν για τις ευρωπαϊκές αξίες και τους διεθνείς κανόνες και πρωταγωνιστούν σε παιχνίδια μετάθεσης ευθυνών. η ελλάδα αγωνίζεται να ελέγξει κατά το δυνατόν μια απέραντη θαλάσσια έκταση στο αιγαίο εκεί όπου και οι ειδικοί της frontex κρίνουν ότι ο αποτελεσματικός έλεγχος είναι αδύνατος. σέβεται το διεθνές δίκαιο συνεργάζεται με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες και σώζει ανθρώπινες ζωές. η ευρωπαϊκή ένωση γνωρίζει πολύ καλά ότι στα παράλια της τουρκίας δρούν τα μεγαλύτερα δίκτυα διακίνησης ανθρώπων τεράστιου τζίρου το πιο απεχθές σύγχρονο οργανωμένο έγκλημα αλλά δεν ασκεί τις αναγκαίες πιέσεις για τη δημιουργία hot spots και εκτός ευρωπαϊκού εδάφους σύμφωνα με το ψήφισμα του συμβουλίου της ευρώπης. εμείς εμένουμε σε αυτό για να μην χαθούν άλλοι άνθρωποι και ζητούμε να υποχρεωθεί η τουρκία να σεβαστεί τις συμφωνίες που έχει υπογράψει και να τηρήσει τις δεσμεύσεις της δεν ωφελεί να απειλούμε την ελλάδα που λόγω της γεωγραφικής της θέσης έχει επομιστεί το βάρος της μεγαλύτερης προσφυγικής κρίσης από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας. τυχόν κατάρρευση της ζώνης σέγγεν θα είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη και δεν θα οφείλεται στη μεταναστευτική κρίση. ο μεγάλος χαμένος θα είναι η ίδια η ευρώπη και οι αξίες της. σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα είναι η μέρα της μαρμότας. Με αυτή την φανταστική ταινία του Bill Murray καταλαβαίνουμε ότι επαναλαμβάνονται ατέρμονα οι μέρες μας και οι διάλογοι μας και η συζήτησή μας. Δεν είναι όμως κομμωδία αυτό. Έφτασε ο χειμώνα, φεύγουν οι πρόσφυγες για να γλιτώσουν από τον πόλεμο. Πολλοί δεν καταφέρουν να φτάσουν στις ε, πόλεις μας γιατί πεθαίνουν στη διαδρομή. Η Europol μας είπε ότι υπάρχουν 10.000 προσφυγόπουλα εξαφανισμένα που έχουν περάσει τα ευρωπαϊκά σύνορα. Από τον Οκτώβριο μιλούμε για πρόγραμμα βοήθεια των προσφύγων στην Τουρκία, ελάχιστη πρόοδο έκτοτε. Ο αντιπρόεδρο κ. Τίμερμαν τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερασπίστηκε τη δημιουργία αυτού του εργαλείου και είπε ότι έτσι οι προθέσει μα θα μεταφραστούν σε πράξει. 24 ώρε μετά την παρουσίαση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε συγκεκριμένη πρόταση χρηματοδότηση έτοιμη να εφαρμοστεί από 1η Πρώτου του 2016 και το Συμβούλιο μετά από τόσου μήνε δεν έχει αποφασίσει ούτε τι θα χρηματοδοτήσει, ούτε πώ ούτε με ποιο τρόπο, ούτε τι θα κάνει. Τι περιμένετε κυρίες και κύριοι του Συμβουλίου, τι πρέπει να συμβεί επιτέλους για να ξεμπλοκαριστούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των 28. Δεν μπορούμε να έχουμε συνέχεια ατέρμονες και στήρες συζητήσεις για τη χρηματοδότηση, για την πολιτική ασύλου, για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το κύμα των προσφύγων. Εν πάση περιπτώσει κλείστε τις απαραίτητες συμφωνίες εσείς του Συμβουλίου. Συμβουλίου κάντε κάτι γιατί ο κόσμος πεθαίνει στις, ε, στις πύλες εισόδου της Ευρώπης. Ο κύριος Μπασίρ παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσο περισσότερο αλλάζουν τα πράγματα, τόσο περισσότερο ίδια μένουν. Συνεχίζουμε να μυρικάζουμε για το θέμα της μετανάστευσης και ενώ είναι πολύ μεγάλη απογοήτευση λόγω της έλλειψης προόδου, δεν είναι αρκετοί αυτοί που είναι έτοιμοι να δεχθούν ότι η στενή συνεργασία με τους γείτονές μας είναι απαραίτητη για να καταφέρουμε να ελέγξουμε κάπως την κατάσταση. Η Τουρκία είτε σε ορισμένους αρέσει αυτό είτε όχι, είναι βασικός εταίρος και παίκτη σε όλη αυτή την κίνηση ε, της μεταναστευτικής κρίσης που ε, μας επηρεάζει όλους. Και η γενικότερη πολιτική σχέση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί μέρος αυτής της συζήτησης. Πολύ απλά, ας μην λησμονούμε ότι η Τουρκία έχει επιδείξει καλή βούληση φροντίζοντας άνω των 2 εκατομμυρίων πρόσφυγες που έχουν ήδη πάει σε αυτή τη χώρα και μένουν. Προφανώς, οποιαδήποτε κονδύλια δοθούν ή δίνονται στην Τουρκία θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά. Όμως τα κέντρα καταγραφής, τα καταφύγια, τα, η τροφή, η εκπαίδευση εκεί ε, θα βοηθήσουν έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κύριος Πιμιέντα Λόπες παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Οι πολιτικές ε, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι στη ρίζα των συγκρούσεων στην Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική. Στηρίζονται ε, ακραίες δυνάμεις, πολλούνται όπλα και δικτατορίες όπως η Σαουδική Αραβία ανθίζουν. Αυτές είναι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Υπήρου και γι' αυτό έρχεται τόσος κόσμος προσπαθώντας να ξεφύγει από τη φτώχεια και από τον πόλεμο θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Τα τείχη και οι λύσεις οι φασιστικές απέναντι στους πρόσφυγες, η έννοια της Ευρώπης οχύρου για να μπορέσουν να συγκεντρωθούν σε πραγματικά στρατόπεδα συγκέντρωσης οι πρόσφυγες είναι ε, απάνθρωπες σε πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντί για αλληλεγγύη παραμένουμε σε άθλιες συνθήκες και προσπαθούμε να τους επαναπατρίσουμε. Η ιστορία οποία θα τιμωρήσει αυτούς που τώρα Σοπένων. Ευχαριστώ. Κυρία Μοντέλεφ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πόσο δύσκολο είναι το ξύπνημα. Παντού στην Ευρώπη η ιδεολογία υπέρ των ε, μεταναστών έχει διαλυθεί. Ε, τρομοκρατικές επιθέσεις, μαζικές κυβιασμοί, αντισημιτισμός και διάφορα άλλα είναι η συνέπεια της τύφλωσής σας. Παρά να ακούτε τα πατριωτικά κινήματα της Ευρώπης που είχε προβλέψει όλη αυτή την ε, κατάσταση, Ελπίζετε με, ότι με διάφορα ημίμετρα θα αντιμετωπίσετε το θέμα. Στηρίζοντας την Τουρκία που παίζει διπλό παιχνίδι με το Ισλαμικό κράτος, ε, θα το πληρώσετε. Το να μην αναλαμβάνετε τις ευθύνε σας σε μια τέτοια ένταση ε, που μεταξύ μεταναστών, προσφύγων και των τοπικών πληθυσμών αυτό, ε, και τις συγκρούσεις μεταξύ τους, παρακαλώ να το ακούσετε και να σταματήσετε αυτή τη συζήτηση κύριε Γιούνκερ, πριν είναι αργά. Ευχαριστώ. Η κυρία Κουντρίτσκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολλά παιδιά έχουν χαθεί καθοδόν προς ε, την Ευρώπη. Υπάρχουν άλλα σοβαρά, άρα σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια στα στρατόπεδα προσφύγων. Επίσης δεν ξέρουμε τίποτα για το ποιόν αυτών των ανθρώπων που έρχονται στην Ευρώπη. Τα παιδιά αυτά δεν έχουν έγγραφα, αλλά για τον ε, χύψη λόγο έχουν περάσει μια διαδικασία καταγραφής και τώρα αναγκάζονται να εκπορνευθούν ή να δουλεύουν ε, σε καταναγκαστική εργασία. Τι θα κάνουμε χωρίς βάσεις ε, δεδομένων και δεν λειτουργεί το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν και η Frontex ε, και η Europol και όλα αυτά εκεί πέρα τα όργανα δεν έχουν ακόμα πρόσβαση σε αυτές τις βάσεις δεδομένων που υπάρχουν. Πώς ε, μπορούμε να πολεμήσουμε τους ε, διακινητές αν τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να ανταλλάξουν πληροφορίες. Επιπλέον, πώς θα συντονίσει η Frontex την προστασία των εξωτερικών συνόρων αν δεν έχει πρόσβαση στην ε, βάση δεδομένων στη χώρα στην οποία κατευθύνεται το μεγαλύτερο κύμα ε, μεταναστών. Έχουμε λοιπόν τη Frontex, έχουμε το σύστημα πληροφοριών Schengen και μετά λέμε «Α, δεν μπορείτε να συνεργαστείτε μεταξύ σας, ούτε καν σε καιρό κρίσης». Σας ευχαριστώ, κυρία Γιώτοβα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαχειριστεί την κρίση των μεταναστών ή να ασχοληθεί μόνο με τις συνέπειες αυτής. Εάν η απάντηση είναι το πρώτο, τότε έχουμε αποτύχει. Ο συσήφιος μύθος θα μπορούσε να είναι το σύμβολο της πολιτικής που ακολουθεί η Ευρώπη για το θέμα αυτό, γιατί δεν λύσαμε κανένα από τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων που προσπαθούν να ξεφύγουν από το θάνατο και τον πόλεμο. Ούτε καθησυχάσαμε τις ανησυχίες των δικών μας Ευρωπαίων πολιτών. Αντί να λαμβάνουμε αλληλέγγυες αποφάσεις, θέλουμε ε, ξεχωριστές κινήσεις ε, σε κάθε κράτος μέλος και ύψωμα ε, φραχτών πρέπει να υιοθετήσουμε εξαιρετικά μέτρα σε εξαιρετικές προθεσμίες ενώπιον εξαιρετικής κατάστασης. Θα πρέπει να σεβαστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο. Αυτό θέλουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθυστερεί την έγκριση του κανονισμού σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Σώμα Φύλαξη Συνόρων. Η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Κροατία αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής. Προσπαθούμε να έχουμε ζώνες προφυλακτήρα μεταξύ των χωρών Σέγγεν και των χωρών διέλευσης. Αυτό προσπαθείτε να κάνετε. Ένας μόνιμος μηχανισμός με την εγκατάσταση κατάστασης πώς θα λειτουργήσει ε, ε, εάν ο προσωρινός μηχανισμός δεν δίνει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. η Τα Βαλκάνια είναι ιδιαίτερη περιοχή κύριε Επίτροπε. Ας μην ε, παίζουμε με τη φωτιά. Και δεν φταίει η Ελλάδα εάν η συμφωνία με την Τουρκία ουσιαστικά δεν δούλεψε. Είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα και όχι ελληνικό. Έχει έρθει πλέον η ώρα το Συμβούλιο να υιοθετήσει συγκεκριμένο πρόγραμμα με συγκεκριμένη δράση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τζαμπάσκι. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, εκπρόσωποι του ΕΛΚ των Σοσιαλιστών και της ΓΚΟΕ, Όλα αυτά δείχνουν την πλήρη αποτυχία της πολιτικής σας, την, της πολιτικής που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και χρόνια σε θέματα μεταναστευσής. Η Τουρκία στηρίζει τους ελαφιστές και εσείς στηρίζετε την Τουρκία και τις προσφέρετε συμφωνίες. Προσπαθείτε να προλάβετε τα πράγματα, αλλά δεν μας ακούσατε ποτέ. Η ολοκλήρωση αποτυγχάνει η ευρωπαϊκή, η πολυπολιτισμικότητα αποτυγχάνει, οι ποσοστώσεις αποτυγχάνουν, η βία στην κολονία τα δικήματα που διαπράττονται, ο υψηλός αριθμός των μεταναστών, ο υψηλός αριθμός των προσφυγόπουλων που έχουν εξαφανιστεί, όλα αυτά είναι δικά σας λάθη και οφείλονται σε εσά και μόνο εσάς. Σταματήστε με τις δικαιολογίες και τα κενά περιεχομένου λόγια. Ο κύριος Μπέγκε. ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, ε, πρέπει να ομολογήσουμε πως οι μηχανισμοί που είχαμε δημιουργήσει ήταν για φυσιολογικούς καιρούς και δεν άντεξαν στην κρίση. Πρέπει να πούμε εδώ πέρα πως πρέπει να γίνει κοινή μας υπόθεση η προστασία των εξωτερικών συνόρων όπως και η κατανομή των βαρών όπως προβλέπει το άρθρο 80 της συνθήκης. Επίσης πρέπει να καθοριστούν ε, σίγουρες και ασφαλείς χώρες ε, προ ε, με συγχωρείτε, προέλευση Αλλά βεβαίω ε, θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, αλλιώ δεν θα σταματήσει η ροή. Θα πρέπει λοιπόν γενικά να δούμε την πολιτική μας όσον αφορά την γειτονία. Τώρα μιλάμε για ένα μέσο για την Τουρκία. Η αρχική πρόταση της Κομισιόν ήταν 500 εκατομμύρια από τον προπολογισμό, 2,5 δισεκατομμύρια από τα κράτη-μέλη. Χωρίς συμμετοχή του Κοινοβουλίου ε, ξαφνικά λέτε ένα δισεκατομμύριο από τον κοινωνικό προπολογισμό. Ε, δεν γίνεται έτσι όμως. Πρέπει να το πω, δεν είναι αυτή η συνεργασία εταίρων. Και μετά έχουμε την Πέμπτη στο Λονδίνο την διάσκεψη των δωρητών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μου λέτε θα δεσμευτεί για 2,2 δισεκατομμύρια. Σας παρακαλώ να διπλασιάζετε τις δεσμεύσεις σας. Επίσης είναι νέα λεφτά ή είναι το πακέτο του Οκτωβρίου 2015 2016 και μετά κυρία Πρόεδρε λέτε για Μακεδονία και Σερβία που θα πρέπει επίσης ε, να ενισχυθούν αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουν πάρει ήδη 500 εκατομμύρια από τον κοινοτικό προϋπολογισμό τα οποία θα πήγαιναν ακριβώς ε, και σε αυτές τις χώρες. Ε, εδώ πέρα μιλάμε δηλαδή για ακροβατικά με τον προϋπολογισμό και δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση της κρίσης των προσφύγων. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πύρη. Ευχαριστώ. Κύρια Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλει προσπάθεια για να αντιμετωπίσει το ζήτημα, αλλά στην πραγματικότητα δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι. Η έλλειψη αλληλεγγύης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η αιτία. Η Ευρώπη του Βίκτορ Όρμπαν έρχεται κάθε μέρα όλο και πιο κοντά. Την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε και άλλα τέτοια ανάλογα. Η Ολλανδική κυβέρνηση ετοιμάζει εναλλακτικά σχέδια ε, για να υπάρξουν ασφαλές ε, δίωδοι για τους ε, πρόσφυγες στην Ευρώπη. Μιλάει για 250.000 άτομα το χρόνο. Και τώρα μας λένε πως θα ακολουθήσουν μόνο όσες χώρες θέλουν. Οι παράνομες δίωδοι θα πρέπει να μην είναι η πιο ελκυστική μέθοδος. Πόσες εναλλακτικές θεωρείτε πως ε, υπάρχουν απέναντι στην ε, Ευρώπη της ε, ιστερίας. Κύριε Αβραμόπουλε, θα πρέπει να αλλάξετε νοοτροπία και νομίζω πως θα βρείτε και περισσότερη στήριξη εντός του Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ κύριε Σφαντάλεν. Κυρία Πρόεδρε, Και κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε, σας ε, καλωσορίζω. Ακούσαμε πως πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Θα πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε συνεχώς σχέδια. Πρέπει κάποια στιγμή να περάσουμε στις πράξεις. Η Ολλανδία που έχει την ε, Προεδρία του Συμβουλίου θα πρέπει να κάνει ένα έκτακτο συμβούλιο και το λέει ως προτεστάντης να ακολουθήσει το μοντέλο της εκλογής του Πάπα στο Βατικανό. Να μην βγείτε αν δεν βρείτε λύση από εκεί μέσα. Η Ευρώπη πραγματικά υποδέχεται ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν από τον πόλεμο με ανοιχτά τα χέρια. Αλλά για ανθρώπους οι οποίοι ζητάνε άσυλο και είναι από Αλβανία, Μαρόκο και οπουδήποτε αλλού δεν υπάρχει χώρος. Πρέπει να επιστρέψουν στις χώρες τους και είναι μια χαρά. Και τέλος δεν πρέπει η, Ευρωπαϊκή, η Τουρκία να βρει ε, τον τρόπο να εμπλακεί περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ πως ένα πρόγραμμα γειτονίας είναι η καλύτερη λύση. Ευχαριστώ κύριο Σκοέλιο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, από την αρχή αυτής της κρίσης των, της προσφυγικής ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να δράσει σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Το ένα άμεσο, το άλλο μακροπρόθεσμο. Το ένα για να αντιμετωπίσει την επίγουσα ανάγκη και το άλλο για να αντιμετωπίσει τη ρίζα του προβλήματος. Ανακοινώνοντας ε, ε, νομοθετικές, νομοθετικά μέτρα δεν αντιμετωπίζονται οι επίγουσες καταστάσεις. Τα κράτη δεν θέλησαν να να βρουν λύσεις από την αρχή και αντιμετωπίζουν συνεχιζόμενες τραγωδίες στη Μεσόγειο και το ίδιο γίνεται τώρα με το Σέγγεν. Ο μηχανισμός ε, σα ανάκλησης ε, είναι αδύναμος οι επιχειρήσεις επιστροφής ε, συνεχίζουν να συμβαίνουν και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά ε, ξαπλώνονται εθνικά ε, μέτρα απομονωμένα και εγωιστικά τι αντιμετωπίζουν τα κράτη και τα κράτη μάλλον θέτουν σε κίνδυνο το Σέγγιν όχι οι πρόσφυγες το να μπορούν να ανακαλέσουν αυτά τα μέτρα τα κράτη μπορούν προσωρινά αλλά είναι προσωρινά δεν λύνει κανένα πρόβλημα αυτό ο χώρος ε, Σέγγεν ανέκαθεν ε, σήμαινε ενισχυμένα εξωτερικά σύνορα. Ο νέος μηχανισμός του Σέγγεν, τον οποίο εγκρίναμε το 2013, δείχνει ότι η Ένωση έχει δυνατότητα να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Όμως, από αυτή την κρίση προκύπτει σαφώς ότι η Ευρώπη δεν ε, χρειάζεται κι άλλα μέσα για να λύσει προβλήματα που τα ευρωπαϊκά κράτη δεν θέλουν να λύσουν. Γι' αυτό θα πρέπει το Frontex να ενισχυθεί. Ευχαριστώ. Γκάιερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Για τον προπολογισμό του 2016 η Ευρωπαϊκή ότι υπήρχε διαθέσιμο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των προσφύγων η Δημοσιονομική Αρχή της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, διέθεσε τα trust funds τα οποία υπήρχαν διαθέσιμα και τα κράτη-μέλη δεν έχουν κάνει ακόμη κάτι τέτοιο. Το ερώτημά μου είναι γιατί ε, συνεννοείστε για τέτοια πράγματα όταν προφανώς δεν είστε διατεθειμένοι να τα χρησιμοποιήσετε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αποδείχτηκε πως ε, στην αντιμετώπιση της κρίσης αυτής η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει έναν επικοδομητικό ρόλο. Γι' αυτό βρίσκω περίεργο Ε, το να μαθαίνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την χρηματοδότηση της Τουρκίας από τις εφημερίδες. Θα έπρεπε να είχατε διαβουλευτεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρέπει να κάνετε κάτι για να διορθώσετε την κατάσταση. Σας ευχαριστώ κύριος Μαριάς. Ορισμένοι κατηγορούν εντελώς άδικα βεβαίως στην Ελλάδα ότι δήθεν δεν περιορίζει τις προσφυγικές ροές στο Αιγαίο. Μάλιστα απειλούν την Ελλάδα με αποβολή από το Σέγγεν, παρότι βέβαια γνωρίζουν ότι αυτό δεν προβλέπεται νομίζετε συνάδελφοι ότι το θέμα της ανάσχεσης των χιλιάδων προσφύγων που φέρνουν τα τουρκικά δουλεμπορικά κυκλώματα στο αιγαίο θα το λύσει η νέα frontex που θα κάνει τι θα βυθίζει βάρκες γεμάτους πρόσφυγες. δεν έχετε άραγε διερωτηθεί γιατί χιλιάδες πρόσφυγες διακινδυνεύουν να πνιγούν στο αιγαίο για να έρθουν στην ελλάδα και δεν επιλέγουν να πάνε από την τουρκία στη βουλγαρία. γιατί άραγε η ελλάδα έχει μετατραπεί σε μαγνήτη για τους πρόσφυγες; μα γιατί είναι η μοναδική χώρα σέγγεν που γετνιάζει με την τουρκία και ως χώρα σέγγεν χορηγεί ταξιδιωτικά έγγραφα που τα παίρνουν οι πρόσφυγες για να πάνε στη γερμανία. εάν η ελλάδα αποχωρήσει από τη σέγγεν τότε το 90% των προσφύγων δεν θα έρχεται στην ελλάδα. Γι' αυτό έχω προτείνει ήδη από τις 11 Δεκεμβρίου η Ελλάδα να κλείσει τα σύνορα και να αποχωρήσει από τη συνθήκη Σέγγεν. Οι αρνητικές συνέπειες για την πατρίδα μου θα είναι ελάχιστες και τα ωφέλη τεράστια. Αφήστε λοιπόν τη διγλωσία άλλωστε η σέγγεν έχει ανασταλεί στη γερμανία τη γαλλία τη σουηδία την αυστρία και τη δανία. εφαρμόστε την πεντεκατάσταση των προσφύγων σταματήστε να θοπεύετε την άγκυρα δημιουργήστε hot spots στην τουρκία. ευχαριστώ. Now, Πρόεδρε, παρά τις δικαιολογημένες επιφυλάξεις πρέπει να προωθήσουμε στην τουρκία τα χρήματα που έχουν εγκριθεί για να καλυφθούν οι ανάγκες των 2,5 έως τριών εκατομμυρίων προσφύγων που έχουν καταφύγει σε αυτήν. Όσο καθυστερούμε, τόσο πιο γρήγορα θα ξεφύγει το προσφυγικό από κάθε έλεγχο. Έχουμε μπροστά μας δύο μήνες δύσκολου καιρού στο Αιγαίο, που σημαίνει ότι οι ροές θα είναι 50 έως 60 χιλιάδες άτομα το μήνα. Από τον Απρίλιο όμως και με τη βοήθεια του καλού καιρού, οι ροές μπορεί να φτάσουν τις 150.000 άτομα το μήνα, αποσταθεροποιώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο εάν αλλάξει η πολιτική της άγκυρας και γίνει πιο περιοριστική θα μειωθούν δραστικά οι προσφυγικές ροές. για να δούμε όμως αν η κυβέρνηση της τουρκίας είναι συνεργάσιμη θα πρέπει πρώτοι εμείς να καλύψουμε τις βασικές οικονομικές ανάγκες των προσφύγων που βρίσκονται στην τουρκία. άλλωστε εμείς επιγόμαστε για γρήγορη μείωση των προσφυγικών ροών. εάν στηρίξουμε οικονομικά τους πρόσφυγες στην τουρκία και αυτή δεν ανταποκριθεί τότε θα κάνουμε αυστηρή την πολιτική απέναντί της. Πρέπει όμως πρώτα να στείλουμε τα χρήματα για να αξιολογήσουμε την αντίδραση της Άγκυρας και να πάρουμε οριστικές αποφάσεις. Πολλοί από τους συναδέλφους πιστεύουν ότι καθυστερώντας την αποστολή ή ματαιώνοντας την αποστολή των χρημάτων θα τιμωρήσουμε το καθεστώς της Τουρκίας για το οποίο εγώ δεν έχω ιδιαίτερα θετική άποψη. Πιστεύω όμως ότι καθυστερώντας την αποστολή των χρημάτων Τιμωρούμε 2,5 έω 3 εκατομμύρια πρόσφυγε και του εαυτού μα. Ευχαριστώ. Ακούω αυτή τη συζήτηση που γίνεται αυτές τις ώρες και αυτές τις εβδομάδες και μήνες, αυτή τη συζήτηση που έχει να κάνει με τις αξίες της Ευρώπη. Παράλληλα όμως γίνεται άλλη μια συζήτηση που μόνος του την κάνει ο πρόεδρος Βέμπερ έναντι της ε, Ιταλικής κυβέρνησης. Εμείς όμως χρειαζόμαστε πολιτική και όχι λογικές ε, ε, τέτοιου τύπου που πάντα παρουσιάζει ο πρόεδρος Βέμπερ. Διερωτώ με, ας πούμε, γιατί σήμερα δεν υπόθηκε ούτε μια λέξη για το δικό του συνάδελφο στο κόμμα του, τον κύριο Όρμπαν, ο οποίος ε, κλείνει με σειρματοπλέγματα τις, τα σύνορά του. Είναι ένα πολύ περίπλοκο πρόβλημα και γι' αυτό χρειάζεται να μιλήσουμε για πολιτική. Χρειάζεται να ξαναδούμε τις αξίες μας, να δούμε το Σέγγεν, πώς θα πρέπει να το ε, προσαρμόσουμε, πώς θα υποδεχτούμε τους πρόσφυγες στην Ήπειρό μας, πώς θα βοηθηθεί η Ιταλία και η Ελλάδα, πώς θα βοηθηθούν τα στρατόπεδα των προσφύγων στη Τουρκία. Και αντί γι' αυτό μιλάμε με τέτοιους όρους. Ε, ε, ίσως Ίσως και είναι μια, ένα ερώτημα που θέλω να θέσω. Η πραγματική επίθεση που κάνει ο Βέμπερ δεν είναι αντίον του Προέδρου Ρέντζη, αλλά ίσως να είναι μια ε, επίθεση κατά της Κομισιόν και του Προέδρου Γιούνκερ. Ο κύριος Μπαρέκοφ. Ε, ευχαριστώ. Είμαι Ευρωπαίος, αλλά καταρχάς είμαι, πάνω απ' όλα είμαι Βούλγαρος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη φάση ε, οδεύει προς την καταστροφή. Το Σέγγεν δεν υπάρχει πλέον. Υπάρχουν νέα σύνορα και η Ευρώπη πολλαπλών ταχυτήτων που έχει καταστήσει τις χώρες τις πιο φτωχές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις έχει μετατρέψει σε γκέτο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να λάβει ούτε καν μια απλή απόφαση. Ε, κάνουμε πολλές υποχωρήσεις απέναντι στο καθεστώς του Ερντογάν που αγοράζει το πετρέλαιο του Νταέσου το να γίνουν οι φτωχές χώρες της Ένωσης όπως η Ελλάδα και η Βουλγαρία χώρες ε, απορρόφησης των σοκ είναι έγκλημα κατά των λαών αυτών. Θα πρέπει να στηριχθούν οι χώρες αυτές όπως και η Βουλγαρία για να στηρίξουν τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Τα χρήματα αυτά θα έπρεπε να δοθούν στους ε, συνοριοφύλακες της Βουλγαρίας και της Ελλάδας και στον Ερντογάν. Θα ήθελα να πω δύο λόγια, λέει ο κ. Βέρκ. Πρώτα απ' όλα, το θέμα της βίας κατά των προσφύγων είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν θα πρέπει καθόλου να παραμεληθεί, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για παιδιά. Χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες παιδιά. Το οργανωμένο έγκλημα δεν περιμένει ούτε σταυρώνει τα χέρια. Ε, Εποφελείται από την κατάσταση και θα πρέπει να φροντίσουμε και τις, ε, τα τις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι γνωρίζουμε το γιατί. Πρέπει να βρούμε απαντήσεις για όλα αυτά τα θέματα. Και επίση πώ θα οργανωθούν και θα περιοριστούν οι μεταναστευτικέ ροέ. Αλλά δεν μπορούμε αυτό να το λύσουμε άμα τσακωνόμαστε μεταξύ μα. Πρέπει να βασιστούμε στι δυνάμει μα και να ενισχύσουμε το Σέγγεν. Αυτή είναι μια δοκιμασία που έχουμε μπροστά μα και είναι δοκιμασία για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δόξα ο Θεό, το τμήμα τη λύση βρίσκεται στου συνοριοφύλακε και το τέταρτο θέμα που θέλω να τονίσω είναι ότι θα πρέπει να χορηγήσουμε το καθεστώς του πρόσφυγα, θα πρέπει να σώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με κάθε τίμημα και γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σωστά τις μεταναστευτικές ροές. Να βοηθήσουμε την Αλβανία, τη Μακεδονία και τη Βουλγαρία που το χρειάζονται. Διαφορετικά θα, θα αρχίσει να ε, επιστρέφουμε τους οικονομικούς μετανάστες. Ευχαριστώ κύριος Λόπες Αγγιγιάρ. Κύριε Πέτροπε, για άλλη μια φορά κάνουμε αυτή τη θλιβερή συζήτηση η οποία δεν έχει αντικείμενο τους πρόσφυγες, έχει αντικείμενο την πληγωμένη Ευρώπη. Παιδιά όπως ο Ιαϊλάν δεν είναι μόνο εικόνα για τα ΜΜΕ, μιλούμε για πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν πνιγεί στις ακτές μας. Έχουμε το ΣΕΚΕΝ, έχουμε αποφάσεις ντροπή στο Συμβούλιο το οποίο το μόνο που κάνει να παρατείνει την αναστολή της ελεύθερης κυκλοφορίας για δύο χρόνια, ενώ μέλη του Συμβουλίου δεσμεύουν τα αγαθά των προσφύγων για να χρηματοδοτήσουν την παραμονή τους, όταν αυτοί έρχονται εδώ προσφεύγοντας ακριβώς και καταφεύγοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση. 10.000 παιδιά προσφυγόπουλα έχουν εξαφανιστεί έχοντας περάσει τα σύνορά μας. Είναι απαραίτητο να ληφθούν αποφάσεις. Ο Ζακ Ντελόρ είπε για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι σαν ένα ποδήλατο το οποίο αν δεν κάνει κανείς ποδήλατο και δεν κουνάει τα πετάλια τότε θα πέσει. Δεν πρέπει να γίνει έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να οπισθοχωρήσουμε στην αποσύνθεση. Πρέπει να έχουμε αλληλεγγύη. Δεν μπορούμε να εγκαταλείπουμε τα εξωτερικά σύνορα, τα πιο αδύναμα που είναι η Ελλάδα. Ο κύριος Γιούρεκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ακούσα πάρα πολλές όμορφες δηλώσεις και όμορφα λόγια για τη μετανάστευση. Όμως από όλα αυτά απουσιάζει η αξιοπιστία. Γιατί σιωπούμε όταν κάποιος ζητά βοήθεια. Γιατί σιωπούμε όταν ακούμε πράγματα που δεν μας αρέσουν. Π.χ. την εξής αλήθεια η βία εναντίον χριστιανών προσφύγων από άλλους μετανάστες στα, στους του προσφύγων και στις δικές μας πόλεις υπάρχει. Έχουμε συγκεκριμένα γεγονότα και τα γνωρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για παράδειγμα, ε, είναι τέτοια περιστατικά που είναι ψηφίσματα για τέτοια περιστατικά που καθυστερεί το Κοινοβούλιο και εβδομάδες να τα συζητήσει δεν είναι διαφορετικές, ξέρετε, οι έννοιες αυτές. Μερικές φορές είναι αντίθετες. Δεν είναι θέμα μόνο αλληλεγγύης, είναι και θέμα της επιβολής της πολυπολιτισμικότητας σε χώρες που επιθυμούν να την αποφύγουν και μπόρεσαν να την αποφύγουν. Η κυρία Ματέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τεράστια μεταναστευτική πίεση στα εξωτερικά τη σύνορα που θέτει σε πολύ δύσκολη δοκιμασία του ε, ε διάφορες συνθήκες μεταξύ των οποίων και τη Σέγγεν. Παρά τη δύσκολη κατάσταση θα πρέπει να είμαστε σε θέση να βρούμε μια σωστή εξισορρόπηση ανάμεσα στις απαιτήσει προστασία των ερωτών ΕΕ, άσυλων, σεβόμενοι έτσι τις υποχρεώσεις μας ε, τη διεθνή, αλλά και την αδυναμία να υποδεχτούμε οικονομικού μετανάστε. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που λάβαμε, που δυστυχώς δεν είναι πάρα πολύ ακριβή, ανάμεσα γύρω στους 500 με 5.000 μετανάστες φτάνουν καθημερινά από την Τουρκία στην Ελλάδα. Είμαστε ευγνώμονες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις νομοθετικές προτάσεις που υπέβαλε τελευταία, αλλά θα πρέπει να δουλέψουμε για να βρούμε πολύ σύντομα μια λύση. Είμαι πεπισμένη πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ένα νομοθετικό και εκτιμένο χρήσιμο και ότι αυτοί οι κανόνες θα πρέπει να εφαρμοστούν μέχρι ε, τέλους και Είμαι πεπισμένη επίσης πως το Σέγγεν θα πρέπει να το υπερασπιστούμε, αλλά όχι να ξεπερνάμε ένα πιο προκαθορισμένο όριο. Η δημιουργία των hot spot και ο μηχανισμών των ποσοστώσεων που όπως είναι φαίνεται να είναι λυπής είναι δύο από τις προτεραιότητες με τις οποίες θα πρέπει να ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να φτάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια οριστική συνεννόηση όσον αφορά τη χρηματοδότηση των τριών δις ευρώ προς την Τουρκία ώστε να ελέγξει τις μεταναστευτικές ροές για την περίοδο 2016-2017. Η Τουρκία μπορεί να είναι ένας εταίρος γεωγραφικός σημαντικός για να επιτύχουμε το στόχο του ελέγχου των ροών. Σε αυτή την ιστορική στιγμή η Ευρώπη δεν δεν μπορεί να ε, δεχτεί τους πάντες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τώρα ο κύριος Ντενανό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντως, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες, κυρίως ε, Σύριοι, έχουν ε, γίνει δεχτεί επισήμως στη τουρκική επικράτεια. Αυτό δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους, γιατί αυτοί οι μετανάστες αργά ή γρήγορα θα έρθουν στις χώρες μας ή θα πάνε σε μια σε κάποια από τις χώρες της Ένωσης. Η Τουρκία όντως ε, βρίσκεται σε πολύ σημαντική γεωστρατηγική θέση και θα πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη συνέχεια. Ε, αυτή η κατάσταση δημιουργεί υποχρεώσει στην ίδια την Τουρκία αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθάει την Τουρκία είναι μια έξυπνη ιδέα την οποία στηρίζω αλλά θα πρέπει αυτό να γίνει με διαφάνεια Ποιο πληρώνει αυτή τη βοήθεια, είναι τα κράτη ή είναι ο προπολογισμό της ενωση ή και οι δύο. ποιο ε, λαμβάνει αυτή τη βοήθεια, είναι η τουρκική κυβέρνηση ή είναι η ΜΚΟ, ποιος ελέγχει τη χρήση αυτών των κονδυλίων, ένα σωρό ερωτήματα στα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να απαντήσουμε, θα πρέπει να γίνει να γίνουν προσπάθειες ώστε αυτή η Τουρκία να μπορέσει αξιοπρεπώς να δεχτεί τους πρόσφυγες στην επικράτειά της. Ο κύριος Χριστοφόρου. Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι το προσφυγικό μας αγγίζει όλους. Και πρωτίστως οφείλω να πω ότι άγγιξε την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όσο και αν ασκούμε κριτική ή αυτοκριτική, πρέπει να λέμε ναι, μπορεί να μην έγιναν όσα έπρεπε να γίνουν, όμως εάν όλοι έκαναν ό,τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, σήμερα πιθανόν να μην συζητούσαμε για προσφυγικό τι έκαναν άλλοι όταν η ευρωπαϊκή ένωση μόνο μέσα στο 2015 έδωσε οικονομική βοήθεια για το ευρύτερο θέμα περίπου 18 δισεκατομμύρια. Πόσες συζητήσεις, πόσες προσπάθειες, πόσες ενέργειες και πόσες δράσεις ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ο Αραβικός Σύνδεσμος, οι Ηνωμένε Πολιτείες της Αμερικής, η Ρωσία, άλλες χώρες ευρωπαϊκές που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά δεν έκαναν τίποτε και βλέπουν με απάθεια ή πολλές φορές ασκούν και κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως πρέπει να πούμε κάτι πολύ σημαντικό τους πρόσφυγες δεν τους δημιουργεί η ελλάδα. η ελλάδα υποδέχεται τους πρόσφυγες. την ίδια στιγμή που κάποιες άλλες χώρες υψώνουν τείχη και φράγματα η ελλάδα υψώνει τον πύχη της αλληλεγγύης και ο δοκιμασμένος ελληνικός λαός με δοκιμασμένη την οικονομία του με λιγοστά μέσα στη διάθεσή του αποδείχθηκε πρότυπο και παράδειγμα και πιστεύω ότι αυτοί που συνεχίζουν να πυροβολούν την ελλάδα δεν αγαπούν την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτοί που θεωρούν ότι η Ελλάδα πρέπει να μείνει εκτό Σέγγεν είναι γιατί θέλουν να υποσκάψουν και να τεινάξουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στον αέρα. Πιστεύω ότι αν θέλουμε να αναζητήσουμε ευθύνε πρέπει να κοιτάξουμε στην Τουρκία, η οποία Τουρκία ουσιαστικά αφήνει του πρόσφυγε και του στέλνει στην Ελλάδα. Τι θέλουν κάποιοι, η Ελλάδα να ξαναστέλνει πίσω στην Τουρκία του πρόσφυγε και ένα τελευταίο, κυρία Πρόεδρε, να πω ότι αξίζει ο ελληνικός λαός και οι έλληνες των νησιών να στηριχθεί πρωτοβουλία και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Επίτροπε, για να πάρουν τον όμπελ ειρήνη για την προσπάθεια και τον ηρωισμό που επέδειξαν απέναντι στους πρόσφυγες. Er Ευχαριστώ. Post. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Από τις τρεις είμαι στην αίθουσα και παρακολουθώ τη συζήτηση. Διαπιστώνω ότι το επίπεδο της συζήτησης είναι πολύ χαμηλό και αυτό είναι κάτι που με απογοητεύει ιδιαιτέρως. Ντρέπομαι γι' αυτό και τρομοκρατούμε κιόλα. Ε, αν λάβω υπόψη μου αυτά που άκουσα να λέγονται σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Διατρέχουμε ένα μεγάλο κίνδυνο σήμερα αυτό το οποίο διακυβεύεται είναι όλο το ευρωπαϊκό εχείρημα. Αυτό το οποίο θέτουμε σε κίνδυνο είναι η πίστη, η εμπιστοσύνη που έχει στο ευρωπαϊκό εγχείρημα η διεθνής κοινότητα. Αν δεν καταφέρουμε εμείς να προασπίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, αν δεν καταφέρουμε εμείς να δείξουμε ουμανισμό, ποιος θα το κάνει. Μιλούμε για το Ισλαμικό κράτος, μιλούμε για το ρατσισμό και λέμε ότι αυτά τα δύο βασίζονται, έχουν τις ίδιες βάσεις. Πρέπει να καταπολεμήσουμε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί. Η έλλειψη σεβασμού που επικρατεί έναντι του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πράγματα απαράδεκτα. Βάσει της τελευταίας έκθεσης της Διεθνούς Αμνηστίας, οι γυναίκες και τα παιδιά είναι αυτοί που υφίστανται κακή μεταχείριση από Ευρωπαίους ε, δημοσίους υπαλλήλους. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να δράσουμε είναι πολύ σημαντική η αξιοπρέπεια. Αλλιώς θέτουμε σε κίνδυνο το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ο, ο κύριος Ράντεφ. Κοιτάξτε κυρίες και κύριοι. Είναι σαφή θες ποια κατεύθυνση πρέπει να πάρει η δική μας μεταναστευτική πολιτική. Θα συνεχίσουμε να εφαρμόσουμε την πολιτική των ανοιχτών θυρών ή θα μειώσουμε τις μεταναστευτικές ροές και θα εγγυηθούμε την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών χωρίς να παραβούμε το διεθνές δίκαιο. Εγώ είμαι υπέρ του ενισχυμένου ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επανειλημμένος. Ε, η Βουλγαρία το κάνει αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εάν τα κράτη-μέλη επενδύσουν στη φύλαξη των συνόρων τους, η αμοιβαία εμπιστοσύνη θα ενισχυθεί και η ελεύθερη κυκλοφορία εντός των συνόρων θα διατηρηθεί. Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ απαραίτητο η νέα υπηρεσία για την ε, φύλαξη των συνόρων, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής, να ασχοληθεί όχι μόνο με τα σύνορα Σέγγεν, αλλά και με όλα τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό θα δείξει ότι επιζητούμε μια ευρωπαϊκή λύση στην μεταναστευτική κρίση. Δυστυχώς, οι βούλγαροι συνοριοφύλακες που πρέπει να αναλάβουν το δύσκολο εγχείρημα να φυλάξουν τα σύνορα με την Τουρκία δέχονται πολύ συχνά την κριτική από ξένες μη κυβερνητικέ οργανώσεις και αυτό είναι κατά την άποψή μου απαράδεκτο. Πόσο μάλλον που ε, όλες οι έρευνες που έχουν λάβει χώρα για να ε, διαπιστώσουν κατά πόσο υπάρχει παράβαση κοινοτική νομοθεσία έχουν καταλήξει στο αντίθετο, στο ότι δηλαδή δεν έχει υπάρξει παράβαση ε, κοινοτική νομοθεσία. Και θα ήθελα να σα ευχηστήσω την προσοχή στην ανάγκη συνεργασία με τις γειτονικέ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωση και κυρίως με αυτές που υποδέχονται τον ε, υψηλότερο αριθμό μεταναστών και που είναι χώρες διέλευση. Μία εταιρική σχέση με τις χώρες αυτές θα κάνει πιο αποτελεσματικό τον αγώνα για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και, ε, και των διακινητών. Η κυρία Νταλή παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συναδελφοί. Δυστυχώ είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία αντί να μιλάμε για τη μεταναστευτική κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρονοτριβεί με πολιτικέ που ασχολούνται μόνο με τι συνέπειε. Είναι ένα ζήτημα το οποίο υπερβαίνει τα ευρωπαϊκά σύνορα και απαιτεί συντονισμένη δράση με διάφορε χώρε Οι προκλήσεις ε, που αντιμετωπίζουμε υποβαθμίζουν τα σύνορά μας ε, αλλά και ευρωπαϊκούς νόμους που ποτέ δεν είχαν στόχο την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα, δηλαδή τις συμφωνίες Δουβλίνου και Σέγγεν. Το σχέδιο μεταγκατάστασης ακόμα δεν λειτουργεί και το μεγαλύτερο βάρος το φέρουν οι χώρες που είναι στην πρώτη γραμμή. Δεν έχει νόημα να δείχνουμε χώρες με το δάχτυλο. Η πραγματικότητα είναι πως οι χώρες, οι μεθοριακές, ε, δεν μπορούν να εγκαταληφθούν χωρίς καθόλου στήριξη. Απαιτούμε ευρωπαϊκές πολιτικές που θα καταδείξουν ότι το πρόβλημα το διαχειρίζονται όλες οι χώρες μαζί. Αλλιώς θα συνεχίσουμε να κάνουμε κύκλους χωρίς να ασχοληθούμε σοβαρά με το ζήτημα και θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Ζόμερ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω πως εγώ τις τελευταίες εβδομάδες ε, εκνευρίζομαι για αυτά τα οποία που ακούω ότι θέμε ευρωπαϊκή λύση. Μα έχουμε ευρωπαϊκή λύση. Έχουμε πάρα πολύ καλούς νόμους. Εντάξει, κάποια πράγματα πρέπει να ρυθμιστούν, είναι εξαιρετικές οι καταστάσεις, αλλά οι νόμοι που έχουμε νομίζω για άσυλο και μετανάστευση δεν είναι άσχημοι, αλλά απλούστατα κάποια καρδιμέλη δεν τους στηρούν. Αυτό πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να αγνοούμε νόμους και κανόνες. Δεν είναι δυνατόν κράτη-μέλη να μην τηρούν ούτε τους νόμους ούτε τις δεσμεύσεις τους. Η αρμοστία του ΟΗΕ δεν λαμβάνει τα χρήματα που τους έχουν προσχεθεί, δεν μπορεί να φροντίσει πρόσφυγες, η Frontex δεν λαμβάνει το επιπλέον προσωπικό κονδύλια και μέσα που έχει ε, ζητήσει. Η Τουρκία δεν λαμβάνει τα υπεσχημένα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τι είναι 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακούγονται πολλά, αλλά σκεφτούμε πόσα έχουμε δώσει ήδη στην Ελλάδα και πόσο πιο φτηνό θα ήταν εντό εισαγωγικών ε, για τα κράτη-μέλη να πληρώσουν αυτά τα τρία δις αντί για να δεχτούν όλους τους ε, πρόσφυγες οι οποίοι ε, πράγματι μπορεί να μην θέλουν όλοι να έρθουν στην Ευρώπη αλλά να είναι πιο κοντά στην πατρίδα τους για να επιστρέψουν. Πού είναι λοιπόν αυτή η περίφημη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Από ό,τι φαίνεται για κάποια κράτη-μέλη ισχύει η αλληλεγγύη μόνο όταν είναι να εισπράξουν λεφτά από τον προπολογισμό. Τότε μιλάνε για αλληλεγγύη. Αλλά δεν είναι δυνατόν αυτό. Δεν είναι δυνατόν να αρνούνται τα κράτη-μέλη απλούστατα και να αφήνουν άλλα να κουβαλάνε το βάρος μόνα τους. Πρέπει τα κράτη-μέλη κάποια στιγμή να ε, δώσουν και κάποιο λόγο. Και η Κομισιόν θα πρέπει να κινηθεί. Μιλάω εδώ πέρα για διαδικασίες επί παραβάση. Ε, κράτη-μέλη θα πρέπει κάποια στιγμή να μην λαμβάνουν πλέον χρήματα τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Σα ευχαριστώ. Κόφοντ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών. Χαίρομαι που σα ξαναβλέπω. όπω ξέρουμε όλοι, το σύστημα του Δουβλίνου κατέρευσε νομίζω. Και ακολουθεί η Σέγγεν αν δεν κάνουμε κάτι. Όλα αυτά είναι άμεσο αποτέλεσμα της έλλειψης αλληλεγγύης μιας κοινή ευρωπαϊκής προσέγγισης έλλειψης αποτελεσματικού ελέγχου των εξωτερικών συνόρων. Και πάρα πολλά κράτη-μέλη δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και δεν παίρνουν το μερίδιο προσφύγων που τους αναλογεί. Κάποια έχουν δεκάδες χιλιάδες αιτήσει, κάποια άλλα εκατοντάδες ή και λιγότερα. Τα κράτη-μέλη που φέρουν το βάρος της εισρωής όπως η Γερμανία, η Σουηδία, η Δανία, η Αυστρία ε, δυστυχώς εξαναγκάζονται να επιβάλλουν σκληρούς νόμους ε, ασύλου. Αυτό είναι μια προσπάθεια να ανταποκριθούμε στον τεράστιο αριθμό προσφύγων δυστυχώ. Ο λόγος για όλα αυτά είναι ότι η Ευρώπη πρώτα απ' όλα δεν αντιμετωπίζει τις ρίζες ε, του προβλήματος και βέβαιω ε, δεν συνεργάζεται με αλληλεγγύη. Τέσσερα μόνο κράτη-μέλη δίνουν 0,7% σε αναπτυξιακή βοήθεια. Απαιτούνται λεφτά για την υπατιαρμοσία του για τους πρόσφυγες και άλλες υπηρεσίες και σας παρακαλώ Κάντε κάτι γι' αυτό. Ενθαρρύνετε τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις ευθύνε τους για πρόσφυγες ε, και για να αντιμετωπίσουν τις αιτίες. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ, μέρα. Σενιόρα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η συνθήκη Σέγγεν είναι σε κίνδυνο και πρέπει να την προστατεύσουμε. Οποιοδήποτε πρόβλημα, όσο περίπλοκο και αν είναι, δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο την ελεύθερη κυκλοφορία μας. Αυτό μάλιστα και πρέπει να σώσουμε και ζωές και να διατηρήσουμε την αρχή της μη επιστροφής. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε τον πόλεμο στη Συρία και δεύτερον θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες και τις δεσμεύσεις που είναι οι δικές μας σε θέματα μετεγκατάστασης υποδομών οικονομικής ενίσχυσης. Μιλώ για αλληλεγγύη και απευθύνομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο επιτέλους να ε, υιοθετήσουν ε, οριστική συμφωνία για τη χρηματοδότηση των τριών δις που δεσμεύτηκαν με την Τουρκία ορίζοντας ε, την ερεσιμότητα ε, της προϋποθέσεις που συνοδεύουν αυτά τα χρήματα και τους όρους. Να σταματήσει το μπλοκάρισμα στο Συμβούλιο επιτέλους, το τέλμα. Τα hot spot πρέπει να γίνουν για να υπάρξει τακτική άφηξη μετακτικότητα στη δική μας επικράτεια. Πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους και αυτά που κάνουν την καταγραφή, αλλά και οι υπόλοιποι που ασχολούνται με την κοινωνική ενσωμάτωση, ένταξη, την οικονομική ενίσχυση και που εγγυώνται ότι θα υπάρξει αφομοίωση και θα σταματήσουν οι συγκρούσεις. Γιατί ξέρετε, οι πρόσφυγες θέλουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους όταν τελειώσει ο πόλεμος. Μιλώ για μια κατάσταση η οποία είναι επίγουσα, αλλά μεταβατικά επίγουσα. Θα πρέπει να προστατεύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα εξωτερικά σύνορα και να επιστρέψουμε όλους αυτούς που δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Και όλα αυτά ε, σεβόμενη ε, τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κιέγκε παρακαλώ. Συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε η Κομισιόν και το Συμβούλιο. Ωστόσο, είμαστε ακόμα πολύ μακριά από την εξέβρεση κοινών απαντήσεων και φοβούμε πως δεν θα τις βρούμε, τουλάχιστον μέχρι ισότου. Σε αυτές τις κοινέ συζητήσει ε, δεν ε, ε, ληφθούν κοινέ πολιτικές αποφάσεις που να είναι φιλόδοξες, καθώς και εφαρμοστικά μέτρα. Είναι, σκανδαλώδες το γεγονός ότι Μέχρι σήμερα μόνο 400 αιτήματα ε, μετεγκατάσταση έχουν γίνει δεκτές από ε, τα κράτη-μέλη. Οι μεταναστευτικέ ροέ ε, δεν γίνεται να σταματήσουν εάν δεν ληφθούν πήγοντα μέτρα και πολιτικές διορατικές και μακροπρόθεσμες. Είναι αλήθεια κύριε Επίτροπε ότι η διάσωση ανθρωπίνων ζωών και η αρχή της μη επαναπρόθεση δεν είναι διαπραγματεύσιμες αξίε. Χωρί μια μακροπρόθεσμη και διορατική οπτική από πλευρά της Ευρώπης θα γίνουμε θύματα πολιτικής αποτυχίας άνευ προηγουμένου και θα πέσουμε στα χέρια δυνάμων ακραίων, ξενοφοβών και λαϊκιστικών. Η ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων, της οποίας, στο στόχος, το τέλος θα σήμαινε την παρακμή του, του σχεδίου ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε Ήσασταν πραγματικά εξαιρετικός ε, το μεσημέρι με τα όσα έχετε ήδη κάνει. Μας εξηγήσετε γιατί ε, τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύουν ε, της, την δημοκρατία, γιατί υπάρχουν οι καθυστερήσεις αυτές που επηρεάζουν το 80% των κονδυλίων σε, ένα κόσμο σε μια περιοχή που χρειάζεται επενδύσεις. Και βέβαια ένα ερώτημα πόσα λεφτά φτάνουν όντως στους πρόσφυγες και δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε γιατί βρίσκονται καινούργια λεφτά από Trust Funds. Θα προσπαθήσουμε εμείς εδώ με συναδέλφους να βρούμε κάποιες ε, κοινέ λύσεις. Υποστηρίζω τις προτάσεις που κάνατε, τις προτάσεις της ε, Κομισιόν και θα ήθελα να ζητήσω και άλλες, ε, δηλαδή συγκεκριμένα να μπορέσουν όλα τα κράτη-μέλη να επιδείξουν τον ίδιο βαθμό αλληλεγγύης που επιζητούν όταν είναι να εισπράξουν κονδύλια. Και θεωρώ πως ε, πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο μας αφορά όλους, ε, δεν είναι θέμα Γερμανίας, Ιταλίας, Τουρκίας, Ελλάδας, Γι' αυτό θεωρώ πως θα πρέπει να πούμε στους ε, συναδέλφους ε, που ζητάνε κάποια αλληλεγγύη και ανήκουν σε κόμματα ε, που οι κυβερνήσεις μετά στις χώρες τους κάνουν τα αντίθετα, θα έπρεπε να πω πως καλύτερα ήταν να μην μιλάνε τόσο πολύ και τόσο μεγαλόφωνα, γιατί η συζήτηση αυτή έπρεπε να γίνει για να ακουστούν κάποια πράγματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Μετσόλα. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, 4,5 ώρες είμαι σε αυτή την αίθουσα και συνεχίζω να πιστεύω ότι καλώς έχουμε αυτή τη συζήτηση. Συμφωνούμε όμως όλοι στο ότι οι πολίτες μας ζητούν συγκεκριμένη δράση από τα κράτη-μέλη. Αρκετά λόγια έχουν ακούσει. Όλοι μας έχουμε ακούσει αρκετά. Πρέπει τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν για τα πιεστικά αυτά ζητήματα του καιρού μας. Ήδη ο κόσμος θα χάσει την πίστη του στην πολιτική αυτή τη διαδικασία. Δεν έχει κανένα νόημα να συμφωνούμε επί όταν απουσιάζει η εφαρμογή, η υλοποίηση και η πολιτική βούληση. Ω προ το Σέγγεν, να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν εσωτερικά σύνορα, γιατί υποσχεθήκαμε ότι τα εξωτερικά σύνορα θα είναι πιο ασφαλή. Το ένα εξαρτάται από το άλλο. Εμπιστευθήκαμε στα κράτη-μέλη το καθήκον να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και μας απαγοήτευσαν σε ορισμένες περιπτώσεις. Άρα χρειαζόμαστε περισσότερα μέτρα και πιο ισχυρά. Αλλά δεν θα αρκέσουν αυτά από μόνα τους. Χρειαζόμαστε μια ολική, συνολική προσέγγιση που θα εξετάζει όλες τις πτυχές. Ναι, πρέπει να επιστρέφεται ο κόσμος τηρώντας πλήρως την αρχή της μη επαναπροώθησης και θα πρέπει όσοι ε, δικαιούνται προστασίες να έχουν την ευκαιρία να τη ζητήσουν. Αν όμως είναι επιλέξιμος θα πρέπει να αποσταλεί πίσω με ασφάλεια και γρήγορα. Όσοι δικαιούνται προστασία θα πρέπει να τη βρουν στην Ευρώπη και σε άλλε ασφαλεί χώρε. Υπάρχουν προκλήσει, αλλά πρέπει να έχουμε διτή προσέγγιση. Όποιο φεύγει από τον πόλεμο πρέπει να έχει τα δικαιώματα τα οποία δικαιούται. Είναι όμω δίκαιο να περιμένουμε να σέβεται τι αρχέ πάνω στι οποίε εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλο η άνοδος ε, του λαϊκισμού και της ξενοφοβίας στην Ευρώπη είναι πολύ ανασυχητική. Τα γεγονότα στην κολονία και οι πρόσφατες ρατσιστικές επιθέσεις δείχνουν ζητήματα που υποβόσκουν και θα πρέπει να λύσουμε. Θα πρέπει να καταστήλουμε το μίσος και ως πολιτικοί έχουμε ιδιαίτερη ευθύνη και δεν πρέπει να την παραγνωρίσουμε. Ο κύριος Φερνάντες, Χωσέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ Κύριε Πίτροπε, κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου, για να μιλήσω για το θέμα των προσφύγων θα σας δώσω μια πολύ εύκολη συνταγή, μια έκκληση. Σεβαστείτε τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάλτε στην πράξη την αλληλεγγύη και ε, υλοποιήστε συγκεκριμένες δράσεις. Αυτό που έλεγε ο Ρόμπερ Σούμεν στην περίφημη δήλωση της 9ης Μαΐου 1950, για τα κοινά προβλήματα μόνο με κοινέ δράσεις και κοινέ ε, λύσει μπορούμε να τα επιλύσουμε. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε ειρήνη, θα υπερνικήσουμε τις προκλήσεις και αυτή ε, ακόμα την κρίση την προσφυγική. Όμως μια αλληλεγγύη δεν σημαίνει μόνο να παίρνει κανείς. Η αλληλεγγύη σημαίνει και να δίνεις. Και είναι απαράδεκτο τα κράτη-μέλη που παίρνουν ε, εκατοντάδες εκατομμύρια, ε, δισεκατομμύρια από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ικανά στη συνέχεια να δώσουν ένα σέντζι για να λύσουν αυτή αυτό το πρόβλημα. Απέναντι σε αυτό το πρόβλημα που έχουμε λοιπόν, θα σας ε, υποβάλω κάποια ερωτήματα. Υπάρχει κάποιο κάτω μέρος που αρνείται να συμβάλλει. Ε, υπάρχουν συγκεκριμένα ποσά για κάθε κάτω μέλος και αυτή η συστήριξη μπορεί να επεκταθεί για την Ιορδανία και το Λίβανο. Ποιος ε, δεν θα εγκρίνει ε, για να υπάρξει βοήθεια επιτόπου. Είναι σημαντικό να δράσουμε με διαφάνεια, με αξιοπιστία και πριν αργά να δράμε ε, να, να, πριν αναργά και να προκύξουν τα, οι διάφοροι ισμοί, εθνικισμοί κτλ. Κύριε Κοράζα Πίλτ, Πρόεδρε, ενώ τα κράτη-μέλη έχουν δείξει διχασμό, δείχνουν μάλλον τσακώνται μεταξύ τους, τα παιδιά πνίγονται στη θάλασσα. Πρέπει να τους λύσουμε και να αντιμετωπίσουμε όλους όσους φτάνουν στην Ευρώπη με αξιοπρέπεια. Οι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν κρίση, όχι εμείς και για τα παιδιά η Ευρώπη θα πρέπει να σημαίνει ασφάλεια και προστασία. Και ξέρετε τι πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχουν εθνικές λύσεις. Έχουμε κοινού κανόνες για την υποδοχή, καταγραφή, εγκατάσταση, επανεγκατάσταση και επιστροφή. Αυτό που λείπει, πούληση από τα κράτη-μέλη. Το Συμβούλιο πρέπει να ενεργήσει, να μοιραστεί τις ευθύνες ή τουλάχιστον δώστε κάποια χρήματα για να βελτιωθούν οι συνθήκες για τους πρόσφυγες και η προστασία τους στην Ιορδανία, στο Λίβανο, στην Τουρκία και, να επιτείνετε τον αγώνα κατά των λαθρε... λαθροδιακινητών. Αυτοί θα πρέπει να φοβούνται, όχι οι πρόσφυγες. Και Κυρία Πρόεδρε, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με αυτό. Η Τουρκία είναι κομμάτι της λύσης, της βραχυπρόθεσμης και της μακροπρόθεσμης. Όλοι όσοι έρχονται στην Ευρώπη δεν έχουν το δικαίωμα να μείνουν εδώ. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε δαχτυλικά αποτυπώματα για να διακρίνουμε ανάμεσα σε αυτούς που έχουν το δικαίωμα διεθνούς προστασίας και, τους και τους, των οικονομικών μεταναστών. Και οι αποτελεσματικέ εξωτερική έλεγχοι στα σύνορα είναι προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη. Η εσωτερική έλεγχη θα είναι το τελευταίο καταφύγιο. Θα πρέπει πια τα κάτι μέλη να σοβαρέψουν για το κόστος ε, κατάργησης του Σέγγεν και το Συμβούλιο παίζει με τη φωτιά αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα περνάμε στην αγαπημένη μου διαδικασία, το Κετσιάνι. Είναι αργά, έχουμε καθυστερήσει. Οπότε ζητώ συγγνώμη, απλά θα, ε, πρέπει να διαλέξω κάποιους ε, βουλευτές, δεν θα μπορέσουν να μιλήσουν όλοι. Η κυρία Σόιντροβα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αντιπρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ. Θεωρώ πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει γρηγορότερα γιατί η κατάσταση δεν βελτιώνεται. Τρία σχόλια έχω, πολύ σοβαρά. Θεωρώ πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να φροντίσει τα παιδιά. Τα παιδιά απειλούνται περισσότερο, είναι η πιο ευπαθής ομάδα. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα μέσο για να είναι ασφαλή τα παιδιά, τα ασυνόδευτα να πάνε σε κάποια σίγουρα κέντρα να μην κυκλοφορούν άστεγα στους ε, δρόμους. Νομίζω αυτό πρέπει να γίνει άμεσα από τη Frontex. Δεύτερον, η προστασία των ε, συνόρων και ειδικότερα των ε, θαλασσίων συνόρων. 18 Φεβρουαρίου πρέπει κάτι να κάνει το Συμβούλιο αυτό είναι προϋπόθεση για την ε, περαιτέρω ελεγγύη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άννα Χέντ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χιλιάδες άνθρωποι προσπαθούν να φύγουν από τον πόλεμο, να ξεφύγουν από το πόλεμο και έρχονται στην Ευρώπη. Καθήκον μας ως άνθρωποι είναι να έχουμε ξεκάθαρη στάση οι ευρωπαϊκές συνθήκες υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα στο άσυλο. Εάν κάποιος ψάχνει καταφύγιο στην Ευρώπη, έχει δικαίωμα να του δοθεί άσυλο. Ορισμένοι όπως ο Ρόμπερτ Φίκο στη Σλοβακία αρνούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους και έχουν ρατσιστικά λόγια εκφέρει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει αποφάσεις ως προς την κατανομή ειδικότερα ως προς τις χώρες ε, που δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Μπορεί η Επιτροπή να μας πει τι θα κάνει τελικά. Ευχαριστώ. Χίλτε Βάτμαν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη να αντιδράσω στον κύριο Κέρκοπ που αναφέρθηκε στο ότι ο Λουί Μισελ εκνευρίστηκε για το ότι κάποιοι δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους και αυτό το παρομοίασε με το να σκοτώνουν κάποιοι τους πρόσφυγες. Ε, κοιτάξτε, δεν υπάρχουν χίλιες λύσεις. Ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει να ξεκουραστούμε καθόλου να μην πάρουμε άδεια κάθε μέρα να ασχολούμαστε με αυτό το ζήτημα. Ξέρουμε ποιες είναι οι λύσεις. Δύο, 10.000 αγνοούμενα παιδιά. Τι σκοπεύετε να κάνετε, ποιο είναι το σχέδιο δράσης για να τα εντοπίσετε. Δεύτερον, ο σύζυγός μου έχει άλλο χρώμα δέρματος και τα παιδιά μου το ίδιο. Νιώθω τον ρατσισμό να αυξάνεται και στη χώρα μου. Τι θα κάνετε για να σταματήσετε τον ρατσισμό. Φροντίστε να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση και να έχουν οι άνθρωποι με διαφορετικό χρώμα μέλλον εδώ στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Χρυσόγονος ακούσαμε επικρίσεις κατά της ελλάδας για την καθυστέρηση λειτουργίας των κέντρων καταγραφής προσφύγων και μεταναστών στα νησιά του αιγαίου. πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι μια χώρα που αντιμετωπίζει μια χωρίς προηγούμενο οικονομική κρίση έχει αντικειμενικές δυσχέρειες να υποδεχθεί και να ελέγξει ένα κύμα προσφύγων και μεταναστών που υπερδεκαπλασιάστηκε το 2015 σε σχέση με το 2014 αντί να κατηγορείτε την ελλάδα παραγνωρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλει με τα πενιχρά της μέσα ασχοληθείτε με το καθεστώς ερντογάν το οποίο παραβιάζει συστηματικά όσα συμφώνησε με την ευρωπαϊκή ένωση και διοχετεύει κατά βούληση τους ανθρώπους στο ελληνικό έδαφος εκβιάζοντας για ακόμη περισσότερα χρήματα από την ευρώπη. ταυτόχρονα η τουρκία επωφελείται από το δουλεμπόριο αφού τα κέρδη των διακινητών εισραίουν στην οικονομία της και τα ενθυλακώνουν και στελέχη του καθεστώτος η ευρώπη οφείλει να επιδείξει πραγματική αλληλεγγύη προς την ελλάδα και να μιλήσει στη γλώσσα των κυρώσεων προς τον κύριο ερντογάν. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Gianluca Vorano. Elnök Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Πρέπει να το συζητήσουμε το θέμα αυτό της μετανάστευσης, αλλά ο τίτλος εδώ πέρα της συζήτησης αφορά την ε, προσφυγική κρίση. Θα ήθελα τώρα να σας πω αυτά τα οποία είπε ένας καθολικός επίσκοπος. Είπε, οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι πρόσφυγες, είναι μετανάστες, είναι δεν είναι οικογένειες, είναι άνδρες, μουσουλμάνοι, δεν θέλουν να προσαρμοστούν. Πρέπει να τα δουν αυτά τα κράτη-μέλη και δεν ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα αλλά με εγκλήματα κατά των προσφύγων. Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι πως το κοινοβούλιο σφάλει ίσως και ηθελημένα και θέλετε να προσφέρετε μια νέα πατρίδα σε αυτούς τους ανθρώπους. Κάνουμε λάθος, δεν περίμεναν αυτό από εμά οι ψηφοφόροι, δεν μα ψήφισαν γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στον χώρο Σέγγεν είναι ένα κεκτημένο εξαιρετικά σημαντικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να το διατηρήσουμε. Δυσκολεύομαι να καταλάβω τις δηλώσεις ορισμένων πολιτικών ανδρών, οι οποίοι λένε ότι δεν πρέπει να δώσουμε κονδύλια για την επίλυση της μεταναστευτικής κρίσης. Και αυτή οι πολιτικοί μιλούν για την αναστολή του χώρου Σέγγεν για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και λένε ότι δεν θα μας αυτό. Εγώ σε ό,τι με αφορά θέλω να πω ότι χωρίς οικονομική ε, ενίσχυση και χρηματοδότηση δεν θα επιλύσουμε αυτή την κρίση. Οφείλουμε όλοι να καταλάβουμε ότι αν δεν το πράξουμε το τίμημα που θα πληρώσουμε θα είναι ακόμα πιο υψηλό. Είναι υποχρέωσή μας επίσης να προβλέψουμε δυνατότητα σε κάθε κράτος μέλος να επαναφέρει τον έλεγχο στα εσωτερικά της σύνορα προσωρινά όμως μόνο. Και καταλαβαίνω γιατί ορισμένες χώρες θέλουν να ενισχύσουν αυτούς τους ελέγχους. Όμως το προσωρινό είναι η λέξη κλειδί σε όλα αυτά. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Χέτμαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να αναφερθώ στην συνθήκη Σέγγεν που είναι το δικό μας και εκτιμένο όλων ημών. Θα πρέπει όλοι να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό και να το υπερασπιζόμαστε. Είναι ένα σχέδιο θαραλέο, καινοτόμο, και ήταν ε, το διαπιστευτήριο, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον υπόλοιπο κόσμο. Είναι το θεμέλιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων και των αγαθών. Το να καταργήσουμε τη συνθήκη του Σέγγεν σημαίνει ότι θα επιβάλλουμε στους εαυτούς μας ένα τεράστιο κόστος το οποίο δεν είμαστε σε θέση να αναλάβουμε. Αντιθέτως πρέπει να ενισχύσουμε το σύστημα, πρέπει να προστατεύσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα και να κάνουμε γρήγορα και αποτελεσματικά βήματα προς αυτό το στόχο. Θα θέλουμε επίσης να εφιστήσουμε την προσοχή όλων στην εταιρική σχέση, στη συνεργασία με την Τουρκία. Έχουν γίνει τα κατάλληλα βήματα και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι την συμφωνία θα εφαρμόσουν αμφότερα τα μέρη. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκόμες παρακαλώ. Την περασμένη Τετάρτη αισθάνθηκα περήφανη που είμαι Πορτογαλίδα. Το Εθνικό μας Κοινοβούλιο με ομοφωνία κατέριψε την πρόταση της Δανίας για την κατάσχεση των τιμαλφών. Ε, τέτοιες πολιτικές ε, θυμίζουν ε, παλιές καθεστώτα αλλά παίζουν και το παιχνίδι των τρομοκρατών. Η Πορτογαλία είναι έτοιμη και περιμένει πρόσφυγες αλλά δεν καταφθάνουν γιατί το σύστημα με δεν δεν λειτουργεί. Ε, η Ελλάδα και η Ιταλία δεν είναι καταλληλώ εξοπλισμένε για να μπορέσουν να διεκπαιρεώσουν όλα ε, τα απαραίτητα. Μόνο από κοινού θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Το να καταστρέψουμε το Σέγγεν δεν θα βελτιώσει του ελέγχου στα σύνορα, ούτε θα λιγοστέψουν οι πρόσφυγες, θα υποφεληθούν μόνο οι διακινητέ. Ε, δεν πρέπει να ανεχόμαστε αυτού του υπουργού που μας γεμίζουν ντροπή και που λένε να, πνίξουμε τους πρόσφυγες που φτάνουν στις πλαγιές μας. Οι υπουργοί που φτιάχνουν ε, νόμους για να καταστήσουν εγκληματίες της ΜΚΟ που βοηθάνε. Ε, δεν μπορούμε ε, να επιτρέψουμε οι κυβερνήσεις μας να εξακολουθήσουν να τροφοδοτούν το λαθρομετανάστευση των προσφύγων να τροφοδοτούν τους διακινητές και να παράγουν τους πρόσφυγες και πρέπει εμείς να τους υποδεχτούμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Επίτροπος Χάν, παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες μου και κύριοι. Κύριε Γκρέσλε, Αντιλαμβάνομαι την ε, σκέψη σας ε, πως θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει κάτι το διαφορετικό. Παρόλα αυτά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σχεδόν 150 ομιλητές για αυτή την ε, συζήτηση και για την παρουσία της. Νομίζω ότι συμφωνούμε πως είναι σωστό οι χώρες οι οποίες είναι πάρα πολύ κοντά στην Συρία και δέχονται το μεγαλύτερο κομμάτι των προσφύγων να βοηθηθούν. Να βοηθηθούν όχι για κάποια, με κάποια κοινική ιστεροβουλία αλλά για ανθρώπινους λόγους. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι παραμένουν στην περιοχή και αυτοί επίσης οι οποίοι είναι πρόσφυγες εντός της ε, Συρίας, ε, μιλάμε για 8 εκατομμύρια, να στηριχθούν και οικονομικά, να παραμείνουν στην ευρύτερη περιοχή έτσι ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν στην χώρα τους ε, όταν επιστρέψει η ειρήνη και να την ανοικοδομήσουν γιατί αυτή την σταθερότητα ε, χρειαζόμαστε στην περιοχή να ανοικοδομηθεί αυτή η καταστραμμένη χώρα των 23 εκατομμυρίων και να επιστρέψει τουλάχιστον ε, ένα κομμάτι της ειρήνης εκεί πέρα. Και εκεί πέρα κάθε ευρώ που επενδύουμε όχι μόνο στην Τουρκία αλλά και στο Λίβανο και στην Ιορδανία και σε μέρη της Συρίας και του Ιράκ θεωρώ πως είναι λεφτά τα οποία εξοδεύουμε σωστά και προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό το λέω απευθυνόμενο σε κάποιους υπουργούς οικονομικών που ίσως τα βλέπουν διαφορετικά. Για το μέσο για την Τουρκία τα γνωστά 3 δισεκατομμύρια. Είναι γνωστό ότι η Κομισιόν μετά τις δυσκολίες που υπήρχαν μεταξύ των κρατών διαφορετικές σκέψεις τελικά καταφέραμε και θα έρθω κύριε Μπέγκε στην κριτική σας να διαθέσουμε ένα δισεκατομμύριο για δύο έτη για να διευκολύνουμε τα κράτη-μέλη να βρουν τα άλλα δύο δισεκατομμύρια. Δεν είναι λοιπόν ότι θα δοθούν αμέσως τα τρία δισεκατομμύρια αυτά στην Τουρκία. Είναι ένα μάξιμουμ ποσό για τρία χρόνια με στόχο να βοηθήσουν τις υπαρκτές οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Τουρκία με το πρόβλημα αυτό. Τα λεφτά αυτά θα πρέπει να πάνε αποκλειστικά σε στρατόπεδα Συρίων προσφύγων για, μέσα, για μέτρα εκπαίδευσης, υγείας, ε, διαμονής. Ε, τα λεφτά αυτά θα τα διαχειριζόμαστε εμείς η δική μου η υπάλληλη. Η Τουρκία βεβαίως έχει το καθεστώς της διαβούλευσης, ε, βεβαίως μας λέει που θα χρησιμεύσουν περισσότερο αυτά τα λεφτά, αλλά θεωρώ πως ε, η διοίκηση είναι δική μας και βεβαίως πάει χέρι-χέρι με μια αξιολόγηση των αναγκών. Να δούμε δηλαδή πού και πώς και σε ποιο βαθμό πραγματικά χρειάζονται τα λεφτά. Τα 3 δισεκατομμύρια λοιπόν όπως είπα είναι ένα στοιχείο μόνο σε ένα action plan το οποίο έχει στόχο να θέσει τη σχέση με την Τουρκία σε μια νέα βάση και αυτό το λέω γιατί εντάξει, δεν είναι ε, η σημερινή συζήτηση αλλά συνεχώς μας ασκείται κριτική για το ότι δεν δίνουμε βάρος στις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή των ε, θεμελιωδών ε, θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας διαβεβαιώ ότι ειδικά στις ε, διαπραγματεύσεις για τα κεφάλαια 23 και 24 δεν θα υπάρξει ούτε ένα χιλιοστό απόκληση από τα θεμελιώδη, από το κράτος δικαίου. Δεν είναι διαπραγματεύσιμα αυτά τα πράγματα, πρέπει να γίνουν σεβαστά και τελείωσε. Ναι κύριε Μπέκε έχετε δίκιο και εγώ θα ήθελα να έχουμε απλούστερους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς αλλά ειλικρινά σας λέω ε, αντιμετωπίζουμε μια πρόκληση. Θα βοηθήσουμε ή θα χαθούμε σε θεσμικές συζητήσεις, ε, σε συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς ε, κτλ. Δηλαδή το θέμα είναι τώρα να φύγει πυροσβεστική να σβήσει τη φωτιά ή να προκηρυχθεί διαγωνισμός για πυροσβεστικά οχήματα. Πραγματικά. Ε, το θέμα λοιπόν είναι να πούμε ναι εντάξει να δώσουμε τα λεφτά και πραγματικά θα ήθελα εδώ πέρα να ευχαριστήσω την ε, συνάδελφο τον Κρυσταλίνα Γεωργιέβα για το ότι τα κατάφερε ένα σημείο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ και αναφέρθηκε και ο φίλος ο Δημήτρης Αβραμόπουλος η σύνθεση των ροών στα Δυτικά Βαλκάνια άλλαξε τις τελευταίες εβδομάδες και σήμερα μπορούμε να πούμε πως 40% ή και λιγότερο ε, των ανθρώπων αυτών είναι όντως Σύριοι και οι υπόλοιποι είναι από άλλες ε, χώρες. Η, η πατιαρμοστία του ΟΗΕ για τους ε, πρόσφυγες την Τετάρτη που μας πέρασε μου είπε πως 45% ε, των ε, αφήξεων ε, στην Ελλάδα γεννήθηκαν στο Ιράν και βεβαίως δεν μπορούμε να μιλήσουμε μόνο για μόρα. Οπότε έχουμε διάφορα πολιτικά ζητήματα. Τέλος. Θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε στιβαρά, εάν μόνο μπορούμε να διασφαλίσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα. Αυτό πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα, γιατί μόνο έτσι θα διατηρηθεί η Σέγγεν. Η Σέγγεν από την οποία αποφελούνται οι πολίτες μας και ήδη στην ε, κεντρική Ευρώπη υπάρχει ένας χώρος ε, κινητικότητας χωρίς σύνορα. Κάτι το οποίο αποτελεί πλέον καθημερινή πρακτική. Πρώτη προτεραιότητα λοιπόν πρέπει να έχει η διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων και ελπίζω οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο να οδηγήσουν πράγματι στο αποτέλεσμα το οποίο προτείνει η Κομισιόν και προσεχώς να έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Mr. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Και τώρα ο Επίτροπος Δημήτρης Σεβραμόπουλος, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας για αυτή την καρποφόρα μαραθώνια συζήτηση ως προς το μάκρος και ως προς την αντοχή έπρεπε κανείς να έχει. Ήταν όμως πάρα πολύ χρήσιμα. Καλωσορίζω το γεγονός ότι όλοι έχουμε κοινούς στόχους. Να τιμήσουμε τις αξίες της Ευρώπης, σεβόμενοι το δικαίωμα των προσφύγων και εξασφαλίζοντας ότι θα διατηρήσουμε, ε, θα προστατεύσουμε τον χώρο Σέγγεν. Ένα, ε, ε, το πιο, από τα πιο απτά επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πρέπει να διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας για να το επιτύχουμε αυτό, όπως κατέστη σαφέστατο και σήμερα. Και τώρα δύο λόγια στα ελληνικά. Για τους φίλους μου ευρωβουλευτές. Ότι όλες οι χώρες μέλη της ε, ζώνης Σέγγεν οφείλουν να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα από το συνοριακό κώδικα. είναι μια βασική αρχή που όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να σέβονται. όμως θέλω να είμαι σαφής για μια ακόμα φορά ποτέ δεν τέθηκε ούτε τίθεται θέμα αποκλεισμού χώρας μέλους της σέγγεν από τη ζώνη σέγγεν. αυτό ούτε καν προβλέπεται πολλές δε από τις ελλείψεις που παρατηρούνται που σημειώνονται σχετίζονται αναπόφευκτα και με τις μεταναστευτικές ροές. αυτό αναγνωρίζεται από όλους και αυτές καλύπτονται και από τη συνδρομή των κρατών μελών αλλά και της ίδιας της επιτροπής. η επιτροπή άμεσα και έμεσα στέκεται στο πλευρό της ελλάδος και όλων των κρατών μελών που είναι αυτόν τον καιρό υποποίηση και θα μου επιτρέψετε τώρα αφού έκανα αυτή την επισήμανση την τόσο ξεκάθαρη να συνεχίσω και πάλι στα αγγλικά. Ε, και θα ήθελα να πω δύο λόγια και να απαντήσω στα όσα είπε ο Γκίφερ Χόφστατ στην αρχή. Αυτό που προσπαθούμε να επιτύχουμε με την δημιουργία hotspots ε, έχει πολλά κοινά στοιχεία με την έννοια της Ευρωπαϊκής Δύναμης Γρήγορης Αντίδρασης για τους πρόσφυγες που πρότεινε ο κύριος Φερχόφστατ. Η ΑΖΟ, η Frontex, η Europol και όπου είναι απαραίτητο και η Eurojust συνεργάζονται επί τόπου μαζί με διεθνείς οργανισμούς ώστε να επιταχυνθεί η αναγνώριση, η καταγραφή και η ε, λήψη δεχτυλικών αποτυπωμάτων από τους ε, πρόσφυγες. Ε, η Κομισιόν έχει στείλει ομάδες επιτόπου για να βελτιωθεί ο συντονισμός. Κανένας δεν μπορεί ούτε δεν θα καταλάβει τα σύνορα οποιοδήποτε κράτους μέλους. Αυτό πρέπει να είναι σαφές. Αλλά όλα τα κράτη-μέλη σύμφωνα με την αρχή της ελληνικής οφείλουν να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη που βρίσκονται στο μέτωπο για να αντιμετωπίσουν αυτή την ανεφρεγουμένου πίεση. Η κυριαρχία των κρατών μελών εξασφαλίζεται από τις συνθήκες. Μάλιστα, καθυστερήσεις έγιναν. Αλλά είναι λάθος στρατηγική να αλλάζουμε στρατηγική μόνο και μόνο λόγω πανικού. Και σε αυτό το σημείο συμφωνώ με την παρέμβαση του Προέδρου της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, του Κλόντ Μωράες, ότι θα επιτύχουμε και μπορούμε μόνο να επιτύχουμε μαζί. Η Ελλάδα επιταχύνει την εφαρμογή και οι συζητήσεις όπως η σημερινή εδώ στέλνουν τη σωστά μηνύματα σε όλες τις κυβερνήσεις ώστε να αναλάβουν και να εφαρμόσουν, να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους. Η Κομισιόν είναι έτοιμη να κάνει ακόμα περισσότερο και δεν σταματάμε στην εφαρμογή μιας συνολικής καθολικής προσέγγισης ε, για το μεταναστευτικό. Το Μάρτιο ήδη θα εκδώσουμε ανακοίνωση για τη διαχείριση της μετανάστευσης ε, ανακοινώντας περαιτέρω βήματα. Επίσης τον Μάρτιο σκοπεύουμε να καταθέσουμε τροποποιημένη πρόταση για τα ΕΦΗ e e σύνορα. Επίσης σκοπεύουμε να υποβάλουμε φιλόδοξο πακέτο διαχείρισης της μετανάστευσης με πρόταση για μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου. Τώρα, ένα διορθωτικό πρόγραμμα επανεγκατάστασης καθώς και πρωτοβουλίες νομικής ε, εγκατάστασης όπως η αναθεώρηση της μπλε κάρτας θα είναι το τμήμα του πακέτου. Βασίζομαι στην πλήρη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην προετοιμασία αυτών των προτάσεων. Όπως έχω ήδη πει, όλοι πρέπει να κάνουμε το μερτικό μας και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας, είτε να αναζητούμε απλές λύσεις που φοβούμε πως δεν υπάρχουν. Προσβλέπω λοιπόν στη συνεργασία μαζί σας για τις επικείμενες προτάσεις. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας. Ας συνεργαστούμε για να τα βγάλουμε πέρα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κύριος Μπάρτ Αντρες. Παρακαλώ. ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίτροποι, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα καταρχάς να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερως όλα αυτά τα σχόλια που κάνατε κατά τη διάρκεια της συζήτησης και κατανοώ και την απογοήτευση που εξέφρασαν ορισμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι σαφές ότι η διαχείριση της ροής των ετούντων άσυλο στην Ευρώπη αποτελεί μια δοκιμή αντοχής για όλους εμάς, για τις χώρες και για τη συνοχή εντός των ευρωπαϊκών κοινωνιών δεν έχει νόημα να χρησιμοποιήσουμε τη συζήτηση για το άσυλο προκειμένου να εξυπηρετήσει ο καθένας πολιτική σκοπιμότητα. Δεν έχουμε αυτό το περιθώριο, αυτή την πολυτέλεια. Οι απλουστευτικές λύσεις και το blame game, το να κατηγορεί ο ένας τον άλλον, ε, είναι κάτι το οποίο είναι κατώτερο των περιστάσεων. Πράγματι η αλληλεγγύη είναι το κλειδί. Συμφωνώ όμως με τους συναδέλφους που είπαν ότι καλά είναι τα λόγια, το θέμα είναι πώς θα μεταφραστούν στην πράξη. Η Προεδρία είναι εξαιρετικά ενεργή. Έχει αναλάβει δράση με τα κράτη-μέλη. Έχει μεταφράσει τα συμπεράσματα σε δράσεις. Υπάρχει έλεγχος των ε, ε, ε, υπάρχει παρακολούθηση των συνεωριακών ελέγχων. Επεξεργαζόμαστε ένα μοντέλο που θα τελειώσει τους διακινητές και το δικό τους επιχειρηματικό μοντέλο, γιατί αυτό πρέπει να σταματήσουμε. Είναι πιο περίπλακα τα πράγματα από ό,τι νομίζουμε και συμπάσχω κι εγώ, νιώθω κι εγώ απογοήτευση όπως και εσείς με, ε, λόγω όλων αυτών των ανθρώπων που βρίσκουν το θάνατο στις θάλασσες. Δεν υπάρχει ακόμα λευκός καπνός, αυτό είναι αλήθεια, αλλά από την άλλη δεν ε, υπάρχει κανένας λόγος να είμαστε απεσιόδοξοι. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τα hot spot, για τα ερωτήματα που τέθηκαν για το μέλλον της συνθήκης Σέγγεν, για την αρχή της μία επαναπροώθησης και για το θέμα της Τουρκίας. Καταρχάς, για τις αξίες μας. Πράγματι, αυτό το οποίο εξέφρασαν οι περισσότεροι είναι ότι εδώ δοκιμάζονται οι ευρωπαϊκές μας αρχές και αξίες. Αυτό είναι αληθές. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε ήσυχοι για το πώς θα αντιδράσουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες ε, από οποιοδήποτε μετερίζει και αν βρίσκονται. Ε, αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι το παν δυνατό για να βελτιώσουμε την κατάσταση με τους ε, μετανάστες που έρχονται ε, ε, στην Ευρώπη. Το είπε ο κύριος Πιτέλα, διακυβεύονται οι αξίες μας, αλλά δεν είναι εύκολο να εφαρμόσονται οι αξίες μας, γιατί από την άλλη υπάρχει ο φόβος και η αντιδράση στο φόβο των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Θα πρέπει να έχουμε διαφορετικές ταυτότητες στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, που να συνάδουν όμως οι διαφορετικές ταυτότητες με τις κοινέ δημοκρατικές ευρωπαϊκές αξίες. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό. Προσπαθούμε να χτίσουμε συνένεση. Άκουσα διάφορες ε, προτάσεις. Ε, είναι πρόβλημα όμως αυτό. Πρέπει να βρούμε λύσεις εντός της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Τώρα για την εξωτερική πολιτική και τις εξωτερικές αξίες μπορώ να αναφέρω κάποια μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, στήριξη από το ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και τις προϋπολογισμούς των κρατών μελών για να βοηθήσουμε την ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, για τους καταφλισμούς προσφυγών στο Ιράκ, στην Ιορδανία, στο Λίβανο και στην Τουρκία. Χθες ε, επέστρεψα από την Αντίσα Μπέμπα όπου συζήτησα το θέμα αυτό με την Ένωση Αφρικανικών Χωρών παρακολουθούμε στενά την εφαρμογή της συμφωνίας της Βαλέτα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει βοήθεια στους εταίρους μας στις χώρες διέλευσης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε ασφαλείς και δυνα... Ε, βιώσιμες δυνατότητες υποδοχής και κατάλληλες διαδικασίες για τους πρόσφυγες και τις οικογένειές τους μέχρι να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσής τους και θα εξετάσουμε μέτρα ε, βελτίωσης της κατάστασης. Πολλά μπορούν να υποθούν για όλο αυτό το θέμα, για την ε, αιτία αυτής της κρίσης θα είναι όμως αντικείμενο άλλες ε, συζήτησης, της συζήτησης για τη Συρία. Για τα hot spot. Πράγματι έχουν προχωρήσει τα πράγματα πολύ αργά. Έχουμε συμφωνήσει από αυτού. Ένα δίκτυο hotspot στην Ιταλία και στην Ελλάδα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για να μειωθεί η μεταναστευτική πίεση στην Ευρώπη. Και άλλωστε έτσι μπορούμε να ταυτοποιήσουμε ποιοι είναι οι επίκοοι τρίτων χωρών που χρειάζονται ε, ευρωπαϊκής προστασίας. Τα hotspot είναι απαραίτητα για να να καθυστερήσουν τις μεταναστευτικές ροές και να ε, ε, εγγυηθούν την ασφάλεια. Και στα hot spot ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα, θα εκδώσει έκθεση ε, ε, έχοντας ενημερώσει τις πληροφορίες και την αξιολόγηση που είχε από το φθινόπωρο του 2015. Θα έχουμε εκθέσεις προόδου κατά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου οι δηλώσεις να γίνουν πράξεις πρέπει κανείς να λειτουργήσει γρήγορα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούμε σε βάθος χρόνου, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα για την μακροχρόνια και μακροπρόθεσμη ε, συνεργασία. Εδώ πρέπει να δράσουμε βράχη πρόθεσμα. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε και είναι θεμητή η κριτική ότι τα πράγματα πηγαίνουν εξαιρετικά αργά. Από το Δεκέμβριο έχει σημειωθεί πρόοδος όμως και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Στην Ιταλία ε, έχουν γίνει λειτουργικές δύο νέες τοποθεσίες, το Πολτσάνο μεταξύ άλλων και η Ελλάδα δουλεύει έτσι ώστε στη Χίο και στη Λέρο να έχουμε δύο νέα hot spot απολύτως λειτουργικά σύντομα. Οι δυνατότητες στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί με τη στήριξη των κρατών μελών και με ε, τη βοήθεια των ειδικών υπηρεσιών του Οργανισμού των Ενωμένων Εθνών. Δεν έχουμε φτάσει στο τέλος του δρόμου, αλλά πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια με νέα δέσμευση και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα στείλει ένα ηχηρό μήνυμα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε να σημειώσουν ταχύτερη πρόοδο στην υποδοχή και καταγραφή των μεταναστών και προσφύγων. Η Ιταλία έχει ένα ποσοστό 100% δάκτυλοσκόπησης, λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων και καταγραφής ε, και όλη η αποβίβαση γίνεται στα hot spot και στην Ελλάδα επίσης από τα hot spot οι μετανάστες μπορούν να φύγουν με ferry boat μόνο εάν παρουσιάσουν αυτό το έγγραφο ταυτοποίησης και καταχώρησης, καταγραφής. Και η Ελλάδα πρέπει να λάβει ε, λογικά ε, μηχανήματα Eurodac ειδικά τις επόμενες ημέρες, περισσότερα τέτοιου είδους μηχανήματα. Πράγματι, ε, το Σέγγεν είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής συνεργασίας και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Όντως προσωρινά έχουν επιβάλει χώρες ε, την αναστολή ε, του Σέγγεν, ε, Σλοβακία, Σουηδία, Φιλανδία, Γερμανία, Αυστρία και ούτω καθεξής, Σουηδία. Μεταξύ άλλων, αυτή η προσωρινή εισαγωγή των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα συνάδει με τη συνθήκη Σέγγεν, προβλέπεται μέσα στη συνθήκη Σέγγεν. Βεβαίω είναι ζήτημα το ότι δεν έχει μειωθεί η μεταναστευτική πίεση και ο χρόνο τρέχει, ο χρόνο τελειώνει και το μέγιστο, η μέγιστη προθεσμία μπορεί να ανανεωθεί μόνο εάν ε, λειτουργήσουμε βάσει του άρθρου 26 της συνθήκης Σέγγεν Δηλαδή η Επιτροπή προτείνει ε, σύσταση που εγκρίνει το Συμβούλιο για την παράταση αυτού του προσωρινού καθεστώτος. Ε, αλλιως θα έχει λήξει η προθεσμία βάσει της οποίας ισχύει ο προσωρινός χαρακτήρας. Επομένως, οι Υπουργοί Εσωτερικών συζήτησαν το θέμα ατύπως στο Άμστερνταμ στις 25 και 26 Ιανουαρίου του 2016 και ευρεία στήριξη ήταν στην πρόταση να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μία πρόταση για συστάσεις βάσει του άρθρου 26 της Συνθήκης Σέγγεν η Προεδρία είναι δεσμευμένη να διατηρήσει το σύστημα Σέγγεν, να καταβάλει το ΠΑΝ, η Ολλανδική Προεδρία, ε, σε συνεργασία με την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και τα κρατη για να βρεθούν λύσεις στα κοινά μας προβλήματα. Τώρα, ως προς την αρχή της μη επαναπρόθεση, έχω κάποιε παρατηρήσει να κάνω για το ζήτημα αυτό. Είναι βασική αρχή, βεβαίω για να απαλύνουμε τις μεταναστευτικές πιέσεις στα κράτη-μέλη και για να γίνει η ταυτοποίηση των υπηκών τρίτων χωρών που χρειάζονται προστασία. Ως Συμβούλιο δουλεύουμε σκληρά έτσι ώστε το δίκτυο των hot spot να είναι λειτουργικό και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης έτσι όπως εγκρίθηκαν αυτές οι διαδικασίες το 2015. Σε αυτό το πλαίσιο προφανώς η αρχή της μη επαναπροώθησης παραμένει ε, πολύ σημαντική. Στην Τουρκία αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ε, ο καθορισμός του καταλόγου των χωρών ασφαλούς προέλευσης. Ε, είναι ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα, συζητείται στο Συμβούλιο αυτή τη στιγμή. Αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν αργότερα επί τη βάση της πολύ συγκεκριμένη αξιολόγησης που θα γίνει. Τώρα, ως προς το κοινό σχέδιο δράσης ΕΕ Τουρκίας, το Συμβούλιο το καλωσόρισε αυτό είναι μέλος μιας ευρύτερης ατζέντα, ενός ευρύτερου θεματολόγιου πολιτικής συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι στέλνονται χρήματα στα τουρκικά σύνορα, απαντώ στον κύριο Φερχόφστατ. Ε, θα συνεργαστούμε με την τουρκική κυβέρνηση έτσι ώστε να υπάρξουν εγγυήσεις και έτσι ώστε να μην είναι μια επιταγή εν λευκό προς τη χώρα αυτή. και θα πρέπει να ε, καταστεί καλύτερη κατάσταση των ε, προσφύγων στην Τουρκία. Στο πλαίσιο του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου είχαμε μια διάσκεψη στο Άμστερνταμ την περασμένη εβδομάδα όπου πολλοί ομιλητές είπαν ότι η κρίση μεταναστευτική και των προσφύγων ε, αποδεικνύει ότι χρειάζεται περισσότερη ευελιξία στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Πρέπει να έχουμε τους πόρους για να αντιμετωπίσουμε κρίσεις που δεν έχουν προβλεφθεί και θα κάνουμε προτάσεις κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία στον προπολογισμό μας. Κάτι το οποίο χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ. Εδώ πέρα ολοκληρώνατε.